Uh, Αγαπητοί φίλοι, παρακαλώ, καθίστε για να ξεκινήσουμε, για να ξεκινήσει αυτή η ακρόαση, για να γιορτάσουμε την Παγκόσμια Μέρα της Γυναίκας 2014 και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών, μια πρόκληση για όλους. Να σας ευχαριστήσω που είστε εδώ εκτιμούμε την αθρώα προσέλευση, γιατί το θέμα είναι σημαντικό. Προεδρεύω στην ε, Επιτροπή για τα Δικαιώματα των Γυναικών και την Ισότητα των Φύλων και για μας αυτό όντως αποτελεί ζήτημα προτεραιότητας τα τελευταία πέντε χρόνια τουλάχιστον και πραγματικά ανυπομονούμε να υπάρχουν θετικές δράσεις, ιδίως σε ό,τι αφορά και τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που περιμένουμε. Είναι λοιπόν σημαντικό το ότι βρισκόμαστε σήμερα εδώ. Πριν πω τίποτε άλλο, να καλωσορίσω τους συναδέλφους από τα Εθνικά Κοινοβούλια. Είναι χαρά μας που είστε εδώ τόσοι πολλοί. Και ένα θερμοκαλωσόρισμα και στους ευρωβουλευτές, αλλά και στους συμμετέχοντες στα διάφορα πάνελ, τους ομιλητές του πρώτου και δεύτερου πάνελ. και βεβαίως και όλους τους υπόλοιπους που παρίστανται. Υπόλοιπες και υπόλοιπους που παρίστανται. Απόψε. Ένας από τους κύριους λόγους για τους οποίους στεκόμαστε στο θέμα της βίας κατά των γυναικών ε, σε αυτήν τη συγκεκριμένη παγκόσμια μέρα για τις γυναίκες είναι ότι την περασμένη εβδομάδα εγκρίναμε μία έκθεση πρωτοβουλίας στην Ολομέλεια του Στρασβούργου όπου ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει μια συνολική στρατηγική, ένα νομοθέτημα σφαιρικό για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών. Το έχουμε ξαναπεί. Είχαμε ετοιμάσει μια έκθεση και πριν από τρία χρόνια που λέγαμε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Αγωνιστήκαμε για να καταλήξουμε στο αποτέλεσμα αυτό και στο παρελθόν, αλλά ως τώρα δεν έχουμε επιτύχει. Και όπως ίσως γνωρίζετε, αυτό το Ευρωκοινοβούλιο δεν μπορεί να υποβάλει νομοθετικές προτάσεις ή νομοσχέδια. Μόνο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να το κάνει αυτό. Γι' αυτό ζητήσαμε ένα σφαιρικό νομοθέτημα που να καλύπτει όλες τις εκφάνσεις της βίας κατά των γυναικών, όχι μόνο κάποιες πτυχές του φαινομένου. Το πρωί ακούστηκε μια μεταφορά ότι η βία κατά των γυναικών είναι σαν μπάζλ, ότι έχει διαφορετικά κομμάτια. Ένα είναι η σεξουαλική παρενόχληση, ένα άλλο είναι ο ακροτηριασμός των γυναικείων γεννητικών οργάνων και ούτω καθεξής. Δεν μπορεί κανείς να πιάσει ένα μόνο από τα κομμάτια και να μην δει την υπόλοιπη εικόνα. Πρέπει να ενώσει τα διάφορα κομμάτια και να δει όλες τις μορφές βίας από κοινού για να καταλάβει ποια είναι η συνολική εικόνα. Αυτή ήταν μια σύντομη εισαγωγή, δεν θέλω να μακρηγορήσω εγώ έχουμε και χρονικούς περιορισμούς. Να σας θυμίσω επίσης ότι υπάρχει διερμηνία σε όλες τις γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Απλώς βρείτε το σωστό κανάλι. Βλέπετε γύρω-γύρω στην αίθουσα τους αριθμούς και τις χώρες, τις γλώσσες των χωρών. Χρησιμοποιήστε λοιπόν και τα ακουστικά αν θέλετε. Επίση να πω ότι δυστυχώ ο πρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου δεν μπορούσε να είναι μαζί μα, ο κύριο Μάρτιν Σούλτ. Λυπάται θερμά γι' αυτό. Αλλά θα μας μιλήσει με ένα μήνυμα μέσω βίντεο και μετά από αυτό θα έχουμε και ένα σύντομο βίντεο για την εισαγωγή στο θέμα. Πρώτα απ' όλα όμως να έχουμε την ε, το μήνυμα του Μάρτιν Σούλτ προς εσάς με βίντεο. Παρακαλώ. Αγαπητοί συνάδελφοι των Εθνικών και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κυρίε και κύριοι, με μεγάλη χαρά σα καλωσορίζω στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη συνεδρίαση αυτή για την πρόληψη τη βία κατά των γυναικών. Όπω κάθε χρόνο, επ' ευκαιρία τη ε, Παγκόσμια ημέρα τη γυναίκα, είναι καλό να εντείνουμε τη συνεργασία μα. Λυπούμε ε, που πρέπει να πω ότι η βία κατά των γυναικών και η ενδοοικογενειακή βία ε, κυριαρχεί στον κόσμο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα. δεν γνωρίζει σύνορα γεωγραφικά, πολιτισμικά, κοινωνικά. Είναι απολύτως αφόρητο και απαράδεκτο και πρόκληση για την κοινωνία μας στο σύνολό της. Θα πρέπει να δούμε ποια είναι η εμπειρία στα κράτη-μέλη και ποιες είναι οι καλύτερες πρακτικές και για ποιο λόγο πιάνουν. Για να γίνουν καλές πολιτικές χρειάζονται και καλά στοιχεία συγκρίσιμα και στα 28 κράτη-μέλη, όπως αυτά που ε, σήμερα δημοσίευσε ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Ξέρετε ότι εμείς στην Ευρώπη έχουμε το νόμο για τα δικαιώματα των ε, θυμάτων και την Ευρωπαϊκή Εντολή Προστασίας. Είναι μενορόσημα, αλλά πρέπει να γίνουν πιο πολλά. Γι' αυτό χρησιμοποιούμε τώρα την νομοθετική ε, δυνατότητα που έχουμε για να ζητήσουμε περισσότερη στρατηγική δράση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ας ενώσουμε με τις δυνάμεις μας οι θεσμοί και η κοινωνία των πολιτών και διεθνώς για να είναι σε σεβαστά τα δικαιώματα όλων των γυναικών και η κεραιότητά τους. Ζητώ συγγνώμη κυρίες και κύριοι που δεν ε, μπορώ να παρευρίσκομαι ε, στην αίθουσα προσωπικά. Σας εύχομαι καλή επιτυχία στις εργασίες σας. Σας ευχαριστούμε. Γι' αυτό και τώρα το επόμενο σύντομο βίντεο, ένα κλιπάκι για την εισαγωγή στο θέμα. Ευχαριστούμε. Πρέπει λοιπόν να βρούμε τρόπους να καταπολεμήσουμε αυτό το πραγματικά έγκλημα. Παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Αυτό είναι. Πριν σας παρουσιάσω τους ομιλητές στο πρώτο πάνελ μας, να κάνω κάποιες παρατηρήσεις διαδικαστικές, ανιαρές ίσως, βαρετές, αλλά για να είμαστε σε μια θετική ατμόσφαιρα. Οι βουλευτές έχουν την ευκαιρία να καταγράψουν το χρόνο αγόρευσης τους στο έδρανο και θα διοργανώσουμε τη συζήτηση σε δύο τμήματα. Πρώτα απ' όλα θα επικεντρωθούμε στις εμπειρίες μας και την νομοθεσία σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο και στο δεύτερο τμήμα θα επικεντρωθούμε στις δυνατότητες στρατηγικής δράσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μπορείτε να επιλέξετε σε ποιο από τα δύο τμήματα της συζήτησης θέλετε να συμμετάσχετε, όμως πρέπει να συμπληρώσετε αυτό το έντυπο. Και την κάρτα για την αγόρευση. Βεβαίως, αν θέλετε, μπορείτε να πάρετε μέρος και στα δύο τμήματα της συζήτησης. Χρόνος αγόρευσης. Και εδώ θέλω να ακούσετε προσεκτικά. Όταν λέμε χρόνος αγόρευσης, εννοούμε ότι έχουμε περιορισμό τριών λεπτών. Όχι επειδή είμαι κακός, και δεν θέλω να διακόψω τον ρημό των ωραίων σκεψεών σας, αλλά έχουμε περιορισμό των πραγμάτων, διότι πρέπει όλοι και όλοι να έχουν την ευκαιρία να πάρουν το λόγο. Πέρυσι, που ήμουν μετριοπαθέστερος, πάλι είχαν όλοι αγόρευσης, αλλά είχα σκεφτεί, εντάξει, είμαι σκανδιναβός και είμαι πολύ αυστηρός με το χρόνο, ας κρατηθώ λιγάκι. Έδωσα σε πολλούς την ευκαιρία να μιλήσουν, πέντε ή έξι λεπτά, και το αποτέλεσμα ήταν ότι πολλοί τελικά δεν πήραν καθόλου το λόγο. Και εκείνοι είχαν θυμώσει μάλλον μαζί μου. Και είχαν και δίκιο. Το καταλαβαίνω. Οπότε θα είμαι πολύ αυστηρός αυτή τη φορά. Τρία λεπτά και το εννοώ για τον καθένα ή την καθεμία. Άλλοι τώρα που δεν είναι βουλευτές ή ευρωβουλευτές μπορούν να λάβουν το λόγο, αλλά μόνον εφόσον το επιτρέπει ο χρόνος μας. Αλλά τότε θα έχετε χρόνο μόνον ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Ελπίζω να καταλαβαίνετε αυτούς τους αυστηρούς, τους δυσάρεστους κανόνες, αλλά θέλω να λάβουν το λόγο στο δυνατόν περισσότεροι. Θα χτυπάω λοιπόν το μικρόφωνο όταν τελειώνει ο χρόνος αγόρευσης. Έχει Εντάξει, όχι με το μικρόφωνο. Ε, ελπίζω να αποδέχεστε το χρόνο των τριών λεπτών. Το ίδιο ισχύει και για τους συμμετέχοντες στα πάνελ. Και για σας ισχύει χρόνος αγόρευσης και περιορισμός. Σας παρακαλώ και εσείς να σεβαστείτε αυτό το όριο, ώστε να έχουν ε, την ευκαιρία οι συμμετέχοντες να θέσουν ερωτήματα μετά. Θα είμαι αυστηρός λοιπόν και με εσάς. Θα σας βάζω χαρτάκια μπροστά σας που θα λένε έχετε άλλα δύο λεπτά και ούτω καθεξής. Μπορεί να αισθάνεστε ότι δεν έχετε φτάσει προς το τέλος, αλλά θα πρέπει να βρείτε τρόπο να ολοκληρώσετε. Αυτό ήταν το βαρετό του κομμάτι. Αλλά πριν ξεκινήσουμε με το πρώτο πάνελ, να ευχαριστήσω τα Εθνικά Κοινοβούλια για τις γραπτές ενισφορές τους. Μας έχουν αποσταλεί μέσω της Επιτροπής των Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φίλων. Σας ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Και να ξεκινήσουμε τώρα με το πρώτο πάνελ, εμπειρίες και νομοθεσία σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Πρώτη μιλήτρια, κυρία Μπλάνκα Χερνάντες Ολιβέρ, υπεύθυνη από την Ισπανική κυβέρνηση για την ε, έμφυλη βία. Έχετε 10 λεπτά το μέγιστο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καλησπέρα σας. Αξιότιμοι εκπρόσωποι των αρχών, βουλευτές, ε, αξιότιμοι ε, εισηγητές, κυρίες και κύριοι, ιδιαίτερα προς την Ισπανική Αντιπροσωπεία. Σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε και την πρόσκληση να παρουσιάσω ε, στο ε, οίκο της Ευρωπαϊκής Δημοκρατίας ε, της θέσης της Ισπανικής Κυβέρνησης. Υιοθετούμε όλα τα θεμέλια των διεθνών οργανισμών για το θέμα αυτό. Η ανισότητα, οι διακρίσεις, η υποταγή της γυναίκας στον άντρα είναι θέματα γνωστά. Θα σας έλεγα πάρα πολύ σύντομα ότι η ισπανική εμπειρία μπορεί να βασιστεί σε μία λέξη που θέλω να σας διαβιβάσω. Οριμότητα. Τι σημαίνει αυτό. Στη χώρα μας αυτό είναι κάτι που δεν κυριαρχεί. Ε, αναγνωρίζουμε ότι έχουν ξεκινήσει πολιτικές πάρα πολύ σημαντικές και βιώσιμες που συνεχίζονται στο χρόνο και αποδίδουν καρπούς τώρα σιγά σιγά αλλά από την άλλη υπάρχει και αναγνώριση κάποιων στοιχείων ή κάποιων προκλήσεων που ακόμα δεν έχουμε καλύψει δεν έχουμε υλοποιήσει δεν έχουμε κατακτήσει, αν θέλετε. Οριμότητα λοιπόν σημαίνει αναγνώριση κάποιων πολιτικών που προχωρούν τώρα στο χρόνο ε, με επιτυχία και συνέχεια σε πολλές περιπτώσεις και αναγνώριση κάποιων τομέων που χρειάζεται ακόμα δουλειά. Καταρχάς θα ήθελα να σας διαβιβάσω ε, το εξής. Έχουμε Κάτι το ιστορικό που ξεκίνησε στη δεκαετία του 80 με την πρώτη μεταρρύθμιση ε, του ποινικού κώδικα. Έγινε κάτι ε, πάρα πολύ ε, σκληρό που συγκίνησε τον κόσμο. Πήγε μια γυναίκα σε ένα κανάλι τηλεοπτικό και κατήγγειλε τον άντρα της, τον σύζυγό της και μετά από λίγες μέρες τη σκότωσε μέσα στο δρόμο. Ε, από τότε υπάρχει ένα πριν και ένα μετά. Άρχισαν τα πρώτα σχέδια δράσης με έναν τρόπο που τώρα πλέον έχει μετατραπεί σε κάτι ε, που δεν μπορεί να γυρίσει πίσω ή να σταματήσει. Η χώρα μας λοιπόν έχει ποντάρει ε, σε αυτή την εξάλληψη της βίας κατά των γυναικών και των θυνών αυτών. Το είπαμε και σήμερα το πρωί στην Ισπανία όλο και περισσότερο η πολιτική εξάλληψη της βίας κατά των γυναικών βία που υφίστανται από το γεγονός και μόνο ότι είναι γυναίκες έχει ε, καταστεί εθνικό ζήτημα και ζήτημα του κράτους. Οι νόμοι γίνονται δεκτοί ε, ομόφωνα, τα ψηφίσματα στο Κοινοβούλιο επίσης. Το τελευταίο πρόγραμμα δράσης της κυβέρνησης ε, γνώρισε μεγάλη συνένεση στον κλάδο και οι γυναικείες οργανώσεις και σύλλογοι έχουν μία πάγια παρουσία, διότι οι γυναίκες ήταν αυτές που ξεκίνησαν όλη αυτή την προσπάθεια πριν από χρόνια δημόσια που τώρα υλοποιείται. Λοιπόν, η πρώτη επιτυχία πιστεύω της χώρας μας ήταν ότι ε, υπάρχει δημόσια δέσμευση και προσήλωση σε αυτό το θέμα που θεωρείται εθνική υπόθεση και ποντάρουμε σε αυτό. Ε, δεύτερον, θα ήθελα να σας δείξω μερικά από τα βιβλία και τις εκδόσεις που ε, έχουμε ε, κάθε μήνα ή κάθε χρόνο στην Ισπανία για την βία κατά των γυναικών. υφίσταται τη βία, επαναλαμβάνω, και μόνο επειδή είναι γυναίκες. Μιλήσαμε για τη σημασία των στοιχείων. Στην Ισπανία δεν αποσιωπώνται, ούτε αποκρύπτονται τα στοιχεία, όσο και αν καμιά φορά είναι αρνητικά. Και αυτά τα στοιχεία ε, τα χρησιμοποιούμε για τρεις σκοπούς. Πρώτον, για να γίνει γνωστό αυτό, κάνουμε μια ακτινογραφία του, προγράμματος, του προβλήματος. Το δεύτερον, το είπε και ο Πρόεδρος, για να προσανατολίσουμε τις πολιτικές μας, τις δημόσιες πολιτικές. Και το τρίτο, για μια εκστρατεία συνειδητοποίησης και ευαισθητοποίησης. Όποιος δεν θέλει, δεν μπορεί να πιστέψει ότι συμβαίνει κάτι τέτοιο, αρκεί να διαβάσει ε, τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τα Θεμέλια Δικαιώματα ή τις δικές μας στατιστικές δημοσίευσεις. Τρίτον, όπως σας είπα, η Ισπανία από τη δεκαετία του 80 έχει αρχίσει να δημιουργεί ένα πολύ μεγάλο και ε, στιβαρό κανονιστικό πλαίσιο. Ένα δημόσιο σύστημα προστασίας, ε, αρρωγής και πρόληψης. Κατά τη δεκαετία του 80 έχουμε τη μεταρρύθμιση του ποινικού κώδικα, στη συνέχεια το 2000 είχαμε δύο ε, θεμελιώδη ε, νομικά κείμενα το 2003 για την εντολή προστασίας, δηλαδή να μην φεύγει η γυναίκα από το σπίτι της, αλλά ε, να μπορεί ο δικαστής να αποφανθεί ότι δίνει 48 ώρες και ε, ε, μέσα σε 48 ώρες υπάρχουν ε, θέματα αστικά, ποινικά, κοινωνικά για την προστασία της γυναίκας και των παιδιών της. Επίσης ένας νόμος που είναι πρωτοπόρος είναι τα μέσα ε, ολοκληρωμένης προστασίας κατά της βίας με βάση το φύλλο. Υπάρχουν και ειδικά δικαστήρια πλέον και ειδική εισαγγελία για αυτά τα θέματα που ασχολείται με όλα τα θέματα που ε, μας απασχόλησαν το πρωί. Παιδεία, υγεία, ε, μέσα ε, μαζικής επικοινωνίας. Πρόσφατα, ε, το 2013, εγκρίθηκε και άλλος νόμος που αναγνωρίζει ε, την ε, δωρεάν νομική συνδρομή ανεξαρτήτως οικονομικών πόρων για οποιαδήποτε γυναίκα που καταγγέλει την κακοποίηση. Και τώρα επίσης έχουμε μεταρρύθμιση του, του ποινικού κώδικα για να συμπεριληφθούν όλα αυτά τα στοιχεία που αναφέραμε και το πρωί. Έχουμε νέο τύπο, νέες μορφές βίας κατά των γυναικών που χρησιμοποιούν και τις νέες τεχνολογίες. Τέταρτη επιτυχία που θα ήθελα να μου επιτρέψετε να σας αναφέρω για τη χώρα μου είναι ότι υπάρχει ε, πραγματικά ένα υπόδειγμα ε, ε, μέτρων. Το τηλέφωνο 016 πάνω από μία πενταετία, πάνω από 400.000 τηλεφωνήματα δωρεάν 24 ώρες το 24ωρο. Τα ηλεκτρονικά βραχιόλια για να ελέγχουμε ότι δεν πλησιάζει ο θήτης στο θύμα. Δικαιώματα ένταξη στην εργασία, σε ποσοστό στην κοινωνική ασφάλιση για να μπορούν αυτές οι γυναίκες που έπεσαν θύμα βίας με βάση το φύλλο να εντάσσονται. Έχουμε ξενώνες που ε, υποδέχονται τις γυναίκες και τα παιδιά τους ε, και επίσης ε, πολύ ευρεία χρηματοδότηση στο τελευταίο πρόγραμμα δάση κυβέρνηση, στην Εθνική Στρατηγική για την Καταπολέμηση και Εξάλληψη της Βίας κατά των Γυναικών, που σας έχουμε επίσης φέρει. Είναι 1,5 δισεκατομμύριο ε, τα κονδύλια, για την ακρίβεια 1,558. Είναι πολύ ενεχόμενοι ε, σε αυτή την υπόθεση. Γνωρίζετε ότι η χώρα μας είναι αποκεντρωμένη και οι περιφέρειες, οι αυτόνομες περιφέρειες έχουν αρμοδιότητες. Υπάρχει όμως και ειδικό οργανισμός που εκπροσωπώ εγώ ε, και είναι κυβερνητικός για την υπόθεση αυτή. Υπάρχουν επιτροπές κοινοβουλευτικές για την ισότητα, εθνικό παρατηρητήριο, όπου συμμετέχουν οι γυναικείες οργανώσεις ε, που έχουν περισσότερη σχέση με αυτό το θέμα και οι πιο σημαντικές. Καθώς επίσης και η τοπική αυτοδιοίκηση συμμετέχει ακόμα και η δικαιοσύνη μέσω ειδικού παρατηρητηρίου που έχουν ε, στο δικαστικό σώμα. Επόμενο θέμα, κάτι που θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικό εμείς στην Ισπανία. Όλο και περισσότερο ο κόσμος συνειδητοποιεί ότι δεν είναι θέμα γυναικών αυτό. Δεν είναι κάτι που απασχολεί μόνο τις γυναίκες ή αφορά μόνο τις γυναίκες που κατέχουν δημόσια αξιώματα. Δεν μπορούν από μόνες τους να τερματίσουν τη βία κατά των γυναικών που επαναλαμβάνω την υφίστανται απλώς και μόνο επειδή είναι γυναίκες. Και η Ισπανία τι θέλει, όλο και περισσότερο να ενέχεται και η υπόλοιπη κοινωνία. Όπως σας είπα, μέσω εταιριών, φαρμακείων, υγεία, ε, σχολεία, συνδικάτα, όλοι. Για ένα τελευταίο που θα ήθελα να σας ε, πω και να σας διαβιβάσω. Έχουμε εδώ ορισμένε εικόνε από τι δράσει μα στον αθλητισμό, στον πολιτισμό. Το τελευταίο που θα ήθελα να σα πω και σημαντικό είναι η πιο πρόσφατη εκστρατεία που άρχισε από την Ισπανία. Ε, εκστρατεία που λέγεται Υπάρχει έξοδο το ζήτησαν οι ίδιες οι γυναίκες που έπεσαν θύματα αυτής της βίας για να καταλάβουμε ότι μετά την βία υπάρχει ελπίδα για διαφορετική ζωή γιατί στην Ισπανία λέγουν τα στοιχεία ότι το 70% των γυναικών που έχουν υποστεί αυτή τη βία έχουν βγει από τη βία αυτή και αυτό ισχύει και για τις ίδιες και για την κοινωνία γενικώ για τη χώρα μου ολόκληρη και ελπίζω, θέλω να ελπίζω και για την Ευρώπη και για τον κόσμο υπάρχει δυνατότητα ε, να δημιουργήσουμε μια κοινωνία χωρίς χωρίς βία κατά των γυναικών. Έχουμε προκλήσεις ακόμα, ε, πιο ευάλωτες ομάδες, συντονισμός, αναγνώριση διαφόρων μορφών βίας κατά των γυναικών και κυρίως να συνεχίσουμε να ενημερώνουμε και να καταρτίζουμε τους επαγγελματίες για να ε, προλαμβάνουν, να μπορούν να προβλέπουν μέσα από ε, τα γυαλιά εντός αγωγικών που θα έχουν αναπτύξει και το ένστικτο αυτό τα σημεία. Θα ήθελα να τελειώσω με αυτό, Πρόεδρε, ότι υπάρχει έξοδος, υπάρχει διέξοδος και ε, θέλουμε να οικοδομήσουμε μια κοινωνία χωρίς βία κατά των γυναικών. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ, που ήρθατε και που μας παρουσιάσατε την πολύτιμη εμπειρία σας στην Ισπανία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τώρα, περνάω στην επόμενη ομιλήτρια ε, την κυρία Μαρία Ινές Γκόμες Ροντρίγκες Φοντίνια, κοινωνιολόγο και διευθύντρια της μη κυβερνητικής οργανωσής Ουνίνιο το παιδί από την Πορτογαλία. Και πάλι 10 λεπτά. E Γεια σας, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που έχω εδώ δίπλα μου την Ισπανίδα φίλη που ανέφερε πολύ σωστά πως ε, πρέπει να οικοδομήσουμε μια κοινωνία χωρίς βία κατά των γυναικών. Πολύ σωστά. Και εγώ ακριβώς ε, γι' αυτό θα ήθελα να μιλήσω για την οικοδόμηση μιας ε, κοινωνίας χωρίς βία κατά, κατά των γυναικών. Θα σας μιλήσω λοιπόν για την δική μου εργασιακή εμπειρία τα τελευταία 40 χρόνια δίπλα σε νέες ε, ιερόδουλες από τις οποίες και από τους οποίους νέους έμαθα πολλά πράγματα γιατί με εμπιστεύθηκαν και μου ε, διηγήθηκαν την πορεία τους, τα αισθήματά τους, τα όνειρά τους με μια λέξη τη ζωή τους. Ξεκίνησα να εργάζομαι στην οργάνωση Ουνίνιου όταν ήμουν 30 χρονών, το 75. Ε, τότε είχαμε την επανάσταση των ε, γαριφάλων και την μεταπολίτευση στην Πορτογαλία. Ήταν, ε, ήταν μια μεταβατική περίοδος για μας. Ε, επικράτησε μια εφορία απελευθέρωσης και σε αυτήν ακριβώς την περίοδο ήρθαν αντιμέτωποι με μια πραγματικότητα που αγνοούσα. Είναι, ήταν η πραγματικότητα κάποιων κοριτσιών που ε, ζούσαν σε ένα ε, καταφύγιο προσπαθώντας να βγουν από τον κόσμο της πορνείας. Άκουσα ε, ιστορίες πρωτοφανείς απρόσμενες ε, για κοπέλες που έτυχαν εκμετάλλευση από την ίδια τους την οικογένεια για παιδιά που εξαναγκάστηκαν να εργαστούν για μια φτώχεια που ε, χαρακτήριζε την παιδική τους ηλικία ξώματα τα οποία είχαν χάσει την αξία τους από τη βία που είχαν δεχτεί διαπίστωσα την ε, ε, απόσταση που είχε δημιουργηθεί ανάμεσα στο σώμα και στο πνεύμα ή την ψυχή τους. Ε, πολλές ε, γυναίκες, αναζη, πολλά κορίτσια αναζητούσαν τους πελάτες σε, σε μπάρι, στους δρόμους ε, και προσπαθούσαν να βρουν μια διέξοδο εκεί, αλλά τελικά δεν έβρισκαν. Προσπάθησα να τη βρουν στο καταφύγιο στο οποίο τις γνώρισα. Ε, πολλές άλλες όμως ε, παραμένουν ε, στο δρόμο με τα όνειρά τους. Ε, είδα την απογοήτευση και την απόγνωση. Μου λέγαν δεν ζω, επιζώ. Είναι μια συνεχής βία η ζωή μου. Ένιωσα την, ε, τις τύψεις τους. Παρ' όλα αυτά οι περισσότερες έλεγαν «Ε, δεν το αξίζω αυτό. Είδα γυναίκες να πεθαίνουν, είδα τα μπαρ πολυτελείας ή τα μπουρδέλα, είδα τα διαμερίσματα στα οποία συναντούσαν τους πελάτες τους, είδα τα παιδιά τους, είδα κορίτσια να ανεβαίνουν με τους πελάτες τους σκάλες για να συναντηθούν μαζί τους στα διαμερίσματα πολυκατοικιών. Είδα πλούσιους να αγοράζουν κορίτσια με πολυτελή αυτοκίνητα. Είδα γυναίκες να αγοράζουν τρυφερότητα από άντρες. Κατάλαβα ότι η πορνεία λειτουργεί ως αγορά με προσφορά και ζήτηση. Προσφορά από τις γυναίκες, ζήτηση από τους άντρες που αγοράζουν. Κατάλαβα ότι στις περισσότερες περιπτώσεις παρεμβαίνει και ο μαστροπός, ένας, μια, ένα τρίτο άτομο. Ε, ο ιδιοκτήτης ενδεχομένως ενός ξενοδοχείου ή του πορνίου ε, κλπ. κλπ. Το γεγονός ότι ο πελάτης πληρώνει ε, τον απενοχοποιεί ε, του δημιουργεί μια απόσταση από το αντικείμενο που είναι η γυναίκα. Έμαθα επίσης ότι η γυναίκα αισθάνεται αντικείμενο, εργαλείο για αυτόν τον άντρα, για να ικανοποιήσει τις φαντασιώσεις του. Ε, μου λέγανε, ε, είμαι ανακυκλώσιμη. Οι πελάτες έρχονται από όλες τις κοινωνικές τάξεις. Αυτό που αλλάζει είναι το που αναζητεί τις γυναίκες. Μπορεί να είναι ένα μπαρ πολυτελείας για τους πιο πλούσιους, όπου και αναζητούνται γυναίκες με ένα συγκεκριμένο κοινωνικό στάτους, αλλά μπορεί να είναι και άλλα σημεία, άλλα μέρη. Γι' αυτό το λόγο, όταν μπήκα μια φορά σε ένα μπαρ πολυτελείας, είδα γυναίκες που έμοιαζαν να, να ανήκουν σε ανώτερες κοινωνικές τάξεις με οικονομική άνεση και ευμάρεια. Όμως στην πραγματικότητα δεν διέφεραν πολλοί από άλλες γυναίκες οι οποίες εκπορνεύονταν σε μέρη πολύ πιο φτωχά. Είδα λοιπόν ότι η προσφορά προσαρμοζόταν στη ζήτηση. Έμαθα ότι η πορνεία ε, πλήττει την σεξουαλικότητα είδα ότι η, η κοινωνία έχει χρησιμοποιήσει την πορνεία ως ένα εμπόρευμα. Και θα έπρεπε να βρούμε έναν τρόπο να περάσουμε από το χρήμα που χρησιμεύει για τα πάντα στο χρήμα που ε, προωθεί αξίες. Ε, η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας ε, θεωρεί ότι η πορνεία αρνείται την σεξουαλικότητα του ανθρώπου. Αρνείται την ανάγκη του για τρυφερότητα, για να δεχτεί ένα χάδι, ένα άγγιγμα. Και ταυτόχρονα απειλεί την σεξουαλική και την σωματική υγεία γενικότερα. Πρέπει η σεξουαλικότητα να μοιράζεται και να τη ζούμε με οριμότητα και ισότητα. Στην πορνεία η πράξη ε, ταπεινώνεται και γίνεται εμπορικό αντικείμενο. Η σεξουαλικότητα γίνεται και πάλι, χρησιμοποιείται με τρόπο βίαιο. Πολλές από τις κοπέλες μου λέγαν το σώμα μου βρίσκεται στο δωμάτιο, αλλά η ψυχή μου αλλού. Πολλές από αυτές έκαναν εμετόπανο στους πελάτες τους. Πολλές δεν αναγνώριζαν τον ίδιο τον εαυτό τους. Άρα για άλλαξε κάτι τα τελευταία χρόνια με ρωτούν πολλοί. Και τους απαντώ ναι, άλλαξαν πράγματα. Ε, έχουμε τώρα πια οργανώσεις, επαγγελματικές ε, οργανώσεις που ζητούν την ομοποίηση της πορνείας ή των δικτύων ε, ε, εκμετάλλευσης. Έχουμε ολόκληρες οικογένειες οι οποίες βρίσκονται μέσα στην απόλυτη φτώχεια. Είδα την Τρόικα να ε, συνομωτεί με, τις, ε, με την κυβέρνηση να αφαιρέσουν ακόμα και την ελάχιστη ελπίδα που υπάρχει. Βλέπω πια μια Ευρώπη όπου δεσπόζουν τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα και μεγάλη μεγάλοι οικονομικοί όμιλοι. Βλέπω ευάλωτες κοπέλες να στρατολογούνται στην πορνεία. Και τελειώνω λέγοντάς σας ότι μια ομάδα γυναικών που βρίσκεται σε μεταβατική φάση μου ζήτησε να σας πω το εξής. Μου ζήτησε να σας πω το εξής. Το σώμα μας δεν μας ανήκει. Ε, ανήκει στον μαστροπό από τον οποίο αγοράζουμε τρυφερότητα και την επιθυμία των πελατών. Ευχαριστώ. Thank you so much. Ευχαριστούμε πολύ. Ήταν πολύ συναισθηματική η ομιλία σας. Μιλήσατε κυρίω για την πορνεία και κάποια στιγμή να διαβάζατε την, τον λόγο σας. ήταν λίγο σαν να ακούγεται ποιήση εδώ. Σας ευχαριστούμε πολύ λοιπόν. Να πάμε στην τελευταία συμμετέχουσα στο πάνελ, την κυρία Ντόρι Λομόρο, μέλος της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων της Ιταλικής Γερουσίας. Έχετε το λόγο. 10 λεπτά. Θέλω κατά πρώτον να ευχαριστήσω τον πρόεδρο της Επιτροπής για τα Δικαιώματα της Γυναίκας και την Ισότητα των Φίλων του Ευρωκοινοβουλίου και τους συναδέλφους βουλευτές που αφιέρωσαν αυτήν την κοινοβουλευτική συνάντηση στο θέμα της πρόληψης και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών. Επίσης που έδωσαν στην Ιταλική Βουλή τη δυνατότητα να παρουσιάσει σύντομα την εθνική μας νομοθεσία για αυτό το τόσο σημαντικό θέμα. Χαιρετίζω λοιπόν όλους τους συναδέλφους των Εθνικών Κοινοβουλίων με τους οποίους περάσαμε μαζί και το πρωί εδώ στις Βρυξέλλες στην ενδιαφέρουσα συζήτηση που είχαμε στις 25 Νοεμβρίου ε, του 2013 γιορτάσαμε τη διεθνή ημέρα για την καταπολέμηση της βίας, ε, της, κατά της έμφυλης βίας. Σε αυτή την περίοδο στην Ιταλία τα μέσα μαζικής ενημέρωση αφιέρωσαν πολύ χρόνο σε αυτό το τεράστιο φαινόμενο που έχει πάρει ανησυχητικέ διαστάσει στη χώρα μας ε, και ήδη από το παρελθόν. Μιλώ για τις γυναικοκτονίες κατά κύριο λόγο. Το 2012 έχασαν τη ζωή του στην Ιταλία 124 γυναίκες ενώ 130 το 2013. Παρόλο που η χώρα μας δεν διαθέτει ακόμη νόμους ε, υποχρεωτικής συλλογής δεδομένων για το φαινόμενο αυτό, τα αριθμητικά στοιχεία που έδωσα είναι από μη κυβερνητικέ οργανώσεις ε, συλλεγόμενα συνήθως. Πάντως η βαθιά οικονομική κρίση που γνωρίζει η Ιταλία, ε, όπως και η υπόλοιπη Ευρώπη, έχει πραγματικά πλήξει τον κοινωνικό ιστό και έχει θέσει εν κινδύνο την ακαιρεότητα της γυναίκας στο πλαίσιο της οικογένειας και της κοινωνίας. Από μία έρευνα που διεξήγαγε το Ιταλικό Ίδρυμα Στατιστικής το 2007 προκύπτει ότι 6.743.000 γυναίκες από τα 16 έως τα 70 έτη έχουν γνωρίσει κακοποίηση ή σωματική βία, ψυχολογική ή σεξουαλική επίσης βία. Ε, για τις γυναίκες ε, για μια γυναίκα στις 3 μεταξύ 16 και 70 ετών. Ένα εκατομμύριο γυναικών έχουν πέσει θέματα βιασμού ή απόπειρα βιασμού. Το 14,3% των γυναικών επίσης ε, έχουν γνωρίσει σωματική ή σεξουαλική βία από τον ίδιο του τον σύντροφο. Το 24,7% των γυναικών ε, δει συμπεριφορά από άλλον άντρα εκτός από τον σύντροφο και 2.077.000 γυναίκες έχουν πέσει θύματα Τη επίμονη παρακολούθηση, όπως λέγεται, του stalking από τον σύντροφό του στη στιγμή του χωρισμού. Ε, τα αριθμητικά αυτά στοιχεία δεν δίνουν ένα την πραγματική εικόνα τη κατάστασης διότι τα περισσότερα από αυτά τα επεισόδια βίας δεν καταγγέλλονται. Μόνο τα τελευταία 20 χρόνια λοιπόν ο εθνικό νομοθέτη. ναι, <clears throat> μόνο τα τελευταία 20 χρόνια ο εθνικός νομοθέτης ε, επιχείρησε τα πρώτα σταθερά βήματα για να καταπολεμήσει το φαινόμενο της βίας κατά των γυναικών. Με μια πολιτιστική επανάσταση, επανάσταση στην νοοτροπία. Κάτι που αφορά ολόκληρη την Ιταλική κοινωνία. Θυμίζω ότι το ελαφρυντικό του εγκλήματος τιμής που προβλεπόταν στον ποινικό μας κώδικα από την περίοδο του φασισμού καταργήθηκε μόλις το 1981. Έτσι λοιπόν προέκυψαν μια σειρά από νόμους, μεταξύ των οποίων ο νόμος 66 του 1996, ε, ρυθμίσεις κατά της σεξουαλικής βίας, που ορίζει την βία κατά των γυναικών ως αδίκημα έγκλημα κατά της προσωπικής ελευθερίας και ο νόμος 154 του 2001 που έχει τον τίτλο «Μέτρα κατά της βίας στις οικογενειακές σχέσεις». Το 2009 με και είναι μια πολύ σημαντική ημερομηνία αυτή και για την Ιταλία με τον νόμο υπαριθμών 38 ο οποίος σχεδόν ομόφωνα ψηφίστηκε από την Ιταλική Βουλή, ε, ε, προβλέφθηκε στην Εθνική Νομοθεσία το ε, έγκλημα της επίμονης παρακολούθησης ως έγκλημα κατά της ηθικής ελευθερίας. Επίσης, αυτό θεωρείται ένα σοβαρό στοιχείο που επιβαρύνει τις δολοφονίες εφόσον έχει προηγηθεί αυτή η επίμονη παρακολούθηση από, την, από τον, έχει προηγηθεί του φόνου. Αυτό λοιπόν είναι κάτι που ε, Επιτέλους έφερε την, Ιταλία την Ιταλία στην ε, διεθνή ε, πορεία που είχαν ακολουθήσει και άλλες χώρες. Η Επιτροπή CDAW και η έκθεση για την Ιταλία της 25ης Ιουνίου 2012 που ε, υπεγράφει από την ειδική συγγήτρια των Ηνωμένων Εθνών για τη Βία κατά των Γυναικών, της αίτια και τις επιπτώσεις του Τρία Μπαντζού, έδειξε ότι τα στοιχεία για την Ιταλία είναι ανισχυτικά. Το ίδιο επιβεβαίωσε και το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για την Ισότητα των φίλων σχετικά με την Ιταλία και επίσης και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου ε, της 6 Δεκεμβρίου 2012. Έτσι, η έκθεση αυτή εντοπίζει πως η οικογενειακή βία ε, αφορά όλες τις γυναίκες σε όλη μας τη χώρα χωρίς διάκριση εδαφική, περιφερειακή ή κοινωνική και πρέπει να γίνουν στην Ιταλία όλες οι σχετικές προσπάθειες με ειδικά νομοθετικά εργαλεία ή με την ίδρυση κυβερνητικών φορέων που να ασχοληθούν με την προώθηση και την προστασία των δικαιωμάτων των γυναικών αλλά παρά το γεγονό αυτό και όλε τι προσπάθειε που έγιναν, δεν υπήρξε πραγματική μείωση των γυναικοκτονιών ή βελτίωση των συνθηκών ζωή των γυναικών ή των κοριτσιών, των νεαρών γυναικών. Το 2013 ο Ιταλό νομοθέτη, μετά από αποτρόπαια ε, περιστατικά της δολοφονίας γυναικών από τους πρώην συντρόφους τους, γυναικών ενήλικων ή εφήβων, ε, έλαβε ακόμα πιο δραστικά μέτρα για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών. Η δολοφονία μιας 15χρονης από τον πρώην φίλο της οδήγησε την Ιταλία τον Ιούνιο του 2013 να κυρώσει την σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και την ενδοοικογενειακή βία η οποία είχε συνταχθεί στην ε, Κωνσταντινούπολη στις 11 Μαΐου 2011 και στην οποία ε, προσπέγραψε η Ιταλία ε, την 27 Σεπτεμβρίου του 2012. Ε, ο νόμος κύρωσης εγκρίθηκε ομόφωνα και από τα δύο σκέλη του Κοινοβουλίου. Αυτή η κύρωση που έχει προφανώς συμβολική αξία ε, είναι για τη χώρα μας ένα σημαντικό βήμα και μια επιπλέον δέσμευση για την εισαγωγή ε, ειδικών μέτρων που πρέπει να προλάβουν και να τιμωρούν ένα φαινόμενο το οποίο έχει λάβει πραγματικά ανησυχητικέ διαστάσει. Το 2013 επίση στην Ιταλία είχαμε τον νόμο 119, ο οποίο προβλέπει και κατεπίγουσε διατάξει σε περίπτωση που απειλείται η ασφάλεια και επίση προβλέπει ειδικέ διατάξει για την καταπολέμηση τη έμφυλη βία. Πρόκειται για ένα λεπτομερέστατο νομοθέτημα το οποίο την ε, αντιμετώπιση της βίας ε, κατά των γυναικών τη θέτει στο κέντρο του ενδιαφέροντός του και το ίδιο ε, απασχόλησε ε, την εισηγήτρια των συνταγματικών υποθέσεων της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων της Γερουσίας. Ο νόμος αυτός έχει σκοπό να δώσει συγκεκριμένα εργαλεία για να προβλεφθεί και να αντιμετωπιστεί ποινικό η περίπτωση κακοποίησης ε, στην οικογένεια, η σεξουαλική βία, η επίμονη παρακολούθηση και μέτρα πρόληψης και προστασίας των θυμάτων. Πολλές από τις διατάξεις προβλέπουν την προσαρμογή της Ιταλικής νομοθεσίας στα πλαίσια της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης. Το 2012 λοιπόν 12 είχαμε τα πρώτα στάδια και τα 2013 την υλοποίηση. Ένα ολόκληρο τμήμα του νόμου αφορά την πρόληψη και την καταπολέμηση της έμφυλης βίας, ιδιαίτερος προβλέπεται η ανάκληση της άδεια παραμονής για ανθρωπιστικούς ή μάλλον η έκδοση άδεια παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους για αλλοδαπές που είναι θύματα κακοποίησης στη χώρα μας. Το ίδιο και η ενίσχυση του δικτύου των εδαφικών υπηρεσιών και των ε, κέντρων για την προσφορά βοήθειας ή των κέντρων υποδοχής σε όλη τη χώρα. Το άρθρο 46, σύμφωνα και με την σύμβαση της Κωνσταντινούπολη, προβλέπει επιβαρυντικά ε, στοιχεία κατά των ε, αυτουργών και των ενόχων. Ιδίως για όλα τα αδικήματα που αφορούν τη ζωή, την σωματική ακαιρεότητα, την προσωπική ελευθερία, την κακοποίηση ε, στην οικογένεια, την ενδοοικογενειακή κακοποίηση, καθώς και μια σειρά από ποινικέ δράσεις, τις οποίες θα παραλείψω τώρα για να προσπαθήσω να ολοκληρώσω και να περάσω στα συμπεράσματά μου. Να πω λοιπόν ότι η Ιταλική Γερουσία χαιρετίζει εκθέσεις του Ευρωκοινοβουλίου για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών Τελευταίο βήμα ήταν ε, η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για, την, ε, για το θέμα αυτό και θέλω εδώ να ευχαριστήσω και την εισηγήτρια που είναι παρούσα. Η διαρκή συμμετοχή της Ιταλικής Βουλής στις πρωτοβουλίες για κοινοβουλευτική συνεργασία ε, Γερουσίας και Επιτροπής θα, του Ευρωκοινοβουλίου δείχνει την πίστη μα στη συνεργασία μεταξύ κοινοβουλίων που δίνει πολλέ νέε δυνατότητε. Εκφράζω λοιπόν την ευχή τα Εθνικά Κοινοβούλια και το Ευρωκοινοβούλιο να μπορέσουν σταδιακά να, να δημιουργήσουν ένα δημοκρατι... μια δημοκρατική ομάδα για να εξετάσουν προβληματισμού που έχουν να κάνουν με την ισότητα των φύλων και κυρίω την βία κατά των γυναικών. Αυτέ τι ημέρε και με αυτά τα λόγια θα κλείσω, διότι είναι πολύ συγκεκριμένη η συνεισφορά μου και αφορά τα βιώματά μου αυτή τη στιγμή δικάζεται ένας α, ανήλικος αυτούργος τη στιγμή που έγιναν ε, τα περιστατικά που εξετάζονται και πατέρας της μικρής και εδώ υπάρχει ειδική ρύθμιση στην Ιταλική νομοθεσία που ε, δίνει ειδική, ειδικές ε, δυνατότητες στον κατηγορούμενο με μια ποινή που τη στιγμή που εκδικάστηκε η υπόθεση δεν ήταν η κατάλληλη. Θα πρέπει λοιπόν εδώ να τελειώσω με αυτή τη σκέψη και με αφορμή αυτό το περιστατικό ότι πρέπει να δρούμε προληπτικά για να αντιμετωπίσουμε και να αναχαιτήσουμε την βία κατά των γυναικών στην ε, κοινωνία. Έχουν γίνει επιτέλου κάποια θετικά βήματα σε νομοθετικό επίπεδο προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά μένουν ακόμη πολλά να κάνουν, ιδίω στο κοινωνικό πλαίσιο που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή και βεβαίω πρέπει να ευαισθητοποιήσουμε γι' αυτό και όλου του πολίτε. Ευχαριστώ. Thank Σας ευχαριστώ πολύ ε, για την προθυμία σας να έρθετε στην ακρόασή μας και να μας δώσετε μια εικόνα της συζήτησης που γίνεται στην Ιταλία και χαίρομαι πάρα πολύ που η Ιταλία ήταν από τις πρώτες χώρες που κύρωσαν ε, την ε, σύμβαση της Κωνσταντινούπολης. Είναι πάρα πολύ καλή και θα παρακαλούσα και θα επιθυμούσα όλες οι χώρες να την κυρώσουν. Λοιπόν, τώρα ακολουθεί συζήτηση, ερωτήσεις αν έχετε, σχόλια. Θα ήθελα μόνο να πω το εξής. Τρία λεπτά έχετε, όπως είπαμε, αλλά ε, μην προσπαθήσετε να τα πείτε όλα σε τρία λεπτά και να μιλάτε πάρα πολύ γρήγορα, γιατί δεν θα σας προλαβαίνουν οι διερμηνείς σε αυτή την περίπτωση. Σας παρακαλώ λοιπόν, προσπαθήστε να μιλήσετε τρία λεπτά με κανονική ομιλία και να μην προσπαθήσετε να χωρέσετε ό,τι έχετε να πείτε μέσα σε τρία λεπτά. Αλλιώς είναι δύσκολο να σας καταλάβουμε γιατί δεν προλαβαίνουν οι διερμηνεί να σα μεταφράσουν. Ωραία. Λοιπόν, τρία ονόματα για να ετοιμάζεστε. Η Λέιλα Χερσικόβατ. από τη Σλοβενία. Στη συνέχεια ο κύριος Λέριντα, πρόεδρος της Επιτροπής ε, της Αρμόδιας της Γερμανικής Βουλής και μετά από την ε, Ευρωβουλή η κυρία Γκουρμάη. Αυτή είναι οι τρεις πρώτοι. Παρακαλώ. Η κυρία Λέιλα Χερσκόβατς. Έχετε το λόγο. Τρία λεπτά παρακαλώ. Κυρίες και κύριοι, Είναι πολύ καλό που είμαστε συγκεντρωμένοι σήμερα εδώ και ελπίζω αυτό να γίνει και στο μέλλον. Πάντως πρέπει να πω ότι η βία κατά των γυναικών δεν είναι ένα απλό φαινόμενο. Έχει προεκτάσει σε όλη την κοινωνία και εδώ θα πρέπει να επικεντρωθούμε στην πρόληψη αυτού του φαινομένου. Έχουμε μια καλή νομοθετική βάση όπως την πρόληψη της αντικογενειακής βίας ή τα εθνικά προγράμματα για την ε, πρόληψη της αντικογενειακής βίας 2009-2014 και συγκεκριμένα προγράμματα με ειδικότερου στόχου και πιο συγκεκριμένα μέτρα. Οι κανόνες συνεργασίας μεταξύ αστυνομίας και άλλων κυβερνητικών ε, φορέων είναι σημαντική βοήθεια. Το ίδιο και το σύνολο κανόνων για την πρόληψη της ενδοκογενειακής βίας με την εργασία ομάδων από πολλές διαφορετικές ε, επιστήμες και κλάδους, αλλά και την δημιουργία κέντρων ε, βοήθειας εφόσον χρειάζεται στήριξη το θύμα. Στο πρόγραμμα δράση 2009-2014 έχουμε ορίσει μια συγκεκριμένη στρατηγική για να επιτύχουμε στο δυνατόν περισσότερου στόχου, να μην καταπολεμήσουμε την ενδοοικογενειακή βία και να ευαισθητοποιήσουμε τον, το κοινό για το πόσο απαράδεκτη είναι οποιαδήποτε μορφή βία και στην οικογένεια και στην κοινωνία γενικότερα. Η Ειδική Επιτροπή τη ε, Βουλή μα για την Ισότητα των Γυναικών για την ζωή των φίλων και τα δικαιώματα των γυναικών, ενημερώνεται συστηματικά για την, ε, τα στάδια υλοποίηση του προγράμματο αυτού για την πρόληψη της ενδοικογενειακή βίας και υπάρχει και διπηρεσιακή ομάδα εργασία για την καταπολέμηση της εμπορία ανθρώπων. Πέρσι η Σλοβενία συμμετείχε σε πολλές συζητήσεις και διαλόγους για την εξάλληψη της βίας κατά των γυναικών και η περσινή έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την κατάσταση σε σχέση με τα δικαιώματα των γυναικών όπου γίνεται λόγος για την πρόληψη και την καταπολέμηση ή την εξάλληψη τίποτα μορφής βίας κατά των γυναικών ε, είναι κάτι το οποίο μας απασχόλησε και εμάς και βεβαίω συμμετείχαμε σε όλα τα στάδια προετοιμασία τη έκθεση αυτή. Παρά τα πολυάριθμα μέτρα που υιοθετήθηκαν σε διεθνέ επίπεδο, δεν υπάρχει κανένα συγκεκριμένο κείμενο για την εξάλληψη τη βία κατά των γυναικών που να είναι δεσμευτικό για όλε τι χώρε του κόσμου. Δεσμευτι... Νομικώ δεσμευτικά επίπεδα υπάρχουν μόνο σε συγκεκριμένα κράτη όπως η Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της Ινδοοικογενειακής βίας, όπου δεν ε, υπάρχει ακόμη κύρωση από την πλευρά της Σλοβενίας. Σίγουρα τα πράγματα θα μπορούσαν να είναι καλύτερα. Χρειάζεται συνεργασία περισσότερων ε, φορέων, ώστε να είναι αποτελεσματικότερη η προσπάθεια καταπολέμησής μας και θα πρέπει να εντείνουμε τις προσπάθειες υλοποίησης των διαφορών νομοθετικών εργαλείων που έχουμε στα χέρια μας, όπως και να κυρώσουμε σύντομα την σύμβαση. Γι' αυτό λοιπόν αναλαμβάνω προσωπικά δέσμευση και υπόσχομαι ως εθνική βουλευτής ότι θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ για να κυρωθεί σύμβαση και από τη Σλοβενία στο δυνατόν συντομότερα. Μπορείτε να ολοκληρώσετε. Ναι θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε και σε αυτό το τομέα. So much for Σας ευχαριστούμε γι' αυτό. Και τώρα ο κύριος Ρέβιερ. Τρία λεπτά. Ευχαριστώ πολύ, Είμαι κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα Δικαιώματα των Γυναικών. Είμαι ομόλογό σας και εγώ από τη Γερμανική Βουλή, στην Αρμόδια Επιτροπή Γυναικών και ε, Νεολαίας και Οικογένειας. Ε, Σα ευχαριστώ πάρα πολύ για τη διοργάνωση αυτής της ακρόασης και ε, είναι και πάρα πολύ επίκαιρη αυτή η υπόθεση Είμαστε στις 5 Μαρτίου, στις 6 Μαρτίου 2013, πριν από ένα χρόνο, δημιουργήσαμε μια τηλεφωνική γραμμή παροχής βοηθείας, όπως είπε και η Ισπανίδα συνάδελφος, που απορρέει από αντίστοιχο νόμο που περάσαμε και υπάρχει η δυνατότητα κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, να μπορούν οι γυναίκες που έχουν πέσει θύμα βίας δωρεάν να τηλεφωνούν σε αυτόν τον αριθμό και να έχουν την ευκαιρία ε, παροχής βοήθειας υπάρχει ανάγκη γιατί στη Γερμανία 40% περίπου και 35% ε, λέει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός ε, είναι οι γυναίκες που ζουν τη βία ιδιαίτερα μέσα στην οικογένεια. Τουλάχιστον μια φορά στη ζωή τους έχουν υποστεί σωματική ή σεξουαλική βία και μάλιστα 58% ε, έχουν υποστεί σεξουαλική παρενόχληση. Στις γυναίκες με αναπηρίες ή προβλήματα διπλασιάζεται σχεδόν το ποσοστό. Μόλις 20% μόνο των γυναικών που έχουν υποστεί χρησιμοποιούν τις ε, υπηρεσίες παροχής συμβουλών. 37% ε, το δεν το γνωρίζουν στη Γερμανία ότι υπάρχει αυτό ή το γνωρίζουν ανελιπώς. Συγγνώμη, Ε, Γι' αυτό δημιουργήσαμε αυτή τη τηλεφωνική γραμμή για να μπορούν οι γυναίκες που δεν το γνωρίζουν ε, να φτάνουν στη βοήθεια, ακριβώς στην αρχή μιας βίαιης σχέσης, να μπορούν χωρίς δυσκολία να επευθύνονται σε κάποιον. Βλέπετε εδώ ε, μία φύσα, είναι μια γυναίκα που έχει πάει στη γυναικολόγο ε, Προηγουμένω τι έχει κάνει όμω πριν φτάσει στη γυναικολόγο. Έχει σηκώσει το τηλέφωνο, έχει τηλεφωνήσει σε κάποιον όταν την κακοποιεί ε, κάποιο στο σπίτι, ο σύζυγο ή κάποιο άλλο πρόσωπο. Γι' αυτό έχουμε δημιουργήσει αυτή τη δυνατότητα με το δωρεάν τηλεφωνικό αριθμό. Καθένας, η κάθε γυναίκα ανώνυμα, ε, δεν χρειάζεται να δώσει το όνομά τη, να μιλάει με αρμοδίου, καλά καταρτισμένου, σε 15 γλώσσε Υπάρχει αυτή η δυνατότητα και επίσης Ε, μπορούν να απευθύνονται και μέλη της οικογένειας, γείτονες, φίλοι, το συγγενικό ή το ευρύτερο περιβάλλον, ε, επαγγελματίες, 70 ε, είναι οι αρμόδιες που εργάζονται εκεί και με βάρδιες είναι 24 ώρες, το 24 ώρο των γυναικών που έχουν υποστεί συζυγική βία, σεξουαλική βία, βιασμό, ε, καταναγκαστικούς γάμους, στόκινγκ, ε, ε, πορνεία, το είπε η συνάδελφος από την Πορτογαλία ή ακόμα και ακροτηριασμό των γενετικών οργάνων, κάτι που έχει να κάνει ιδιαίτερα με γυναίκες μετανάστριες και ε, όποιος ε, ε, θέλει βοήθεια, όποια γυναίκα μπορεί να δεχτεί τη βοήθεια κοντά στο σπίτι της και πάντα διαφημίζεται αυτό το νούμερο με φυλάδια σε εφημερίδες κτλ. Ελπίζω ότι είμαστε σε σωστό δρόμο να βοηθούμε όσο μπορούμε περισσότερες γυναίκες. Ευχαριστώ για την υπομονή σας. Ευχαριστώ πολύ για τη συνεισφορά σας και τώρα θα ακούσουμε δύο ευρωβουλευτές. Πρώτα την κυρία ε, γκουρμάι, θα έχουν την ευκαιρία να μιλήσουν οι προβουλευτές. Οι ίδιοι κανόνες ισχύουν, τρία λεπτά αυστηρά και θα είμαι εξίσου αμήλικτος. Μπορείτε να βλέπετε πόσο χρόνο καταναλώσετε. Υπάρχει ένα ρολόι επάνω στην οθόνη σας. Παρακαλώ κοιτάτε το. Η κυρία Γκουρμάη, έχετε το λόγο για τρία λεπτά. Καταρχήν θα ήθελα να σας ε, να συγχαρώ την Ιταλία για την ισότιμη εκπροσώπηση ανδρών και γυναικών στην καινούργια κυβέρνηση. Ε, καλωσορίζω αυτή το, το αυτή σημερινή εκδήλωση είναι μια από τις πιο σημαντικές παραβίες ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρόλε τις προσπάθειες και τις εκστρατείες τα νούμερα ακόμα είναι πολύ ψηλά. Και τα στοιχεία τα οποία δημοσιεύθηκαν, ε, σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά, μία, μία στις τρεις ε, γυναίκες στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει υποστεί βία, σωματική ή σεξουαλική βία. Ε, δεν θα αναφέρω πολλά άλλα νούμερα, μόνο ένα. Κάθε μέρα στην Ευρώπη 7 γυναίκες χάνουν τη ζωή τους εξαιτίας της ενδοοικογενειακής βίας. Γι' αυτό το λόγο είναι σημαντικό να εστιάσουμε σε αυτό το θέμα. Μία βδομάδα μετά την υιοθέτηση της έκθεσης Παρβάνοβα. Υποστηρίζω τις προτάσεις της κυρίας Παρβάνοβα. Είναι αιτήματά μας εδώ και χρόνια. Εδώ και χρόνια υπενθυμίζουμε ότι χρειάζεται μια σφαιρική προσέγγιση για να αντιμετωπίσουμε το φαινόμενο. Δεν, δεν μπορούμε απλώς να ε, τιμωρούμε ε, τους δράστες. Πρέπει να, ε, φέρουμε, να στήσουμε εκστρατείες ευαισθητοποίησης, ενημέρωσης, κατάρτισης κλπ. Χρειαζόμαστε μια ε, συνολική στρατηγική σε ευρωπαϊκό επίπεδο και κοινοτική νομοθεσία. Ένα κείμενο ευρωπαϊκό, νομοθεσία ευρωπαϊκή, την οποία έχει ζητήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επανειλημμένο στο παρελθόν. Χρειαζόμαστε ένα αρμονισμένο ορισμό για την βία κατά των γυναικών στα κράτη-μέλη. Επίσης, κοινέ προδιαγραφές για την αστυνομική συνεργασία διασυνοριακά, που είναι πολύ σημαντικό για την προστασία των θυμάτων. Για να είμαστε αποτελεσματικοί χρειαζόμαστε επίσης ασφαλή στατιστικά στοιχεία. Γι' αυτό το λόγο και η, έκθεση της, ε, του Οργανισμού Θεμελιών Δικαιωμάτων, της Υπηρεσίας Θεμελιών Δικαιωμάτων είναι πολύ σημαντική. Τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν πλέον από τους πολιτικούς αλλά και από τους νομικούς. Το άλλο σημείο που συνδέεται με την εκπαίδευση και την ευαισθητοποίηση είναι ότι η βία αυτή είναι ριζωμένη όσο οποιαδήποτε άλλη. Γι' αυτό το λόγο χρειαζόμαστε ε, να καταπολεμήσουμε το πρόβλημα στα θεμέλια του, στη ρίζα του, με, με εκπαίδευση. Πρέπει το θέμα να επιστρέψει στην ευρωπαϊκή πολιτική ατζέντα και να μην το συζητούμε μόνο τις μέρες που είναι πριν ή λίγο μετά την Διεθνή ημέρα της ε, γυναίκας. Είναι ένα σοβαρό θέμα το οποίο δεν μπορούμε να ανεχθούμε πλέον. Αυτό θα πρέπει να γίνει σαφές. Τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα πρέπει να πάρουν, ε, να αναλάβουν δράση. Χρειαζόμαστε εκστρατείε όπως αυτές στο παρελθόν, στην οποία έχω συμμετάσχει, στην οποία συμμετείχα και έδειξε ότι μπορεί να αποδώσει καρπούς. Ευχαριστώ. Ο λόγος στην κυρία Κλάς τώρα, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ για το θέμα. Και θα ήθελα να πω επίσης ότι οι αριθμοί και τα παραδείγματα που ακούστηκαν είναι κυριολεκτικά τρομακτικά. Πονάει η καρδιά μας και η ψυχή μας. Και ε, το είδαμε αυτό και από την ταινία προηγουμένως. Όλοι είπαν τι έχει γίνει μέχρι τώρα. Περνούν νόμοι, συμβάσεις, μέτρα καταπολέμηση της βίας, ναι σε όλα αυτά. Αλλά ε, διερωτώ αρχίζουμε αρκετά νωρίς και εγκαίρως, γιατί αρχίζουμε εμείς κατόπιν εορτής, όταν έχει συντελεστεί η βία και την έχουμε εντοπίσει. Πώς ορίζεται όμως η βία, είμαστε σε θέση ε, εγκαίρως και νωρίς να αναγνωρίζουμε φαινόμενα βίας κατά των γυναικών, πριν φτάσει πραγματικά στη χειροδικία. Ε, γυναίκες με μελανιές, με πληγές, ορατές, σωματικές, αυτές είναι οι γυναίκες που είναι θύματα βίας. Έτσι ορίζεται η βία. Εμένα δεν μου αρκεί αυτό αγαπητοί συνάδελφοι. Νομίζω θα πρέπει πολύ νωρίτερα να ρίξουμε το βλέμμα μας και να, την προσοχή μας να στρέψουμε. Υπάρχει και η ψυχική βία και θα πρέπει να συμπεριληφθεί. Η βία κατά των γυναικών είναι και ψυχική. Είναι και οι γυναίκες που δεν έχουν αυτοπεποίθηση. Ε, και γυναίκες και τα κορίτσια αλλά και οι άνδρες και τα γόρια. Εκεί θα πρέπει να δράσουμε στην παιδεία, στην εκπαίδευση υποχρεωτικά σε όλα τα σχολεία. Όπως εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, ζητάμε συχνά ε, σεξουαλική διαπαιδαγώγηση. Δεν μιλώ γι' αυτό. μιλάω για τις αξίες της ανθρώπινης επαφής και επικοινωνίας να μαθαίνουμε στο σχολείο. Ότι θα πρέπει να σεβόμαστε άνδρες και γυναίκες ε, να υπάρχει πολύ μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση, ε, όχι με την έννοια της διαπαιδαγώγησης. Δυστυχώς στην οικογένεια αυτό δεν γίνεται. Σήμερα έχει αλλάξει η ζωή στην οικογένεια. Γι' αυτό θα πρέπει περισσότερο το κράτος και το σχολείο να ασχοληθεί με αυτό. Και θα ήθελα να παρακαλέσω και τους συναδέλφους από τα Εθνικά Κοινοβούλια και να ρωτήσω αν το έχουμε σκεφτεί αυτό και σε ποιο βαθμό το υλοποιούμε. Δηλαδή, πολύ νωρί προληπτικά, να λέμε και στα παιδιά μας ποια είναι η κοινωνία και πώς θα πρέπει να φερόμαστε ο ένας τον άλλον. Γιατί πιστεύω ότι ένας άνδρας που ε, έχει αυτοσεβασμό και αυτοπεποίθηση δεν είναι βίαιος και δεν θα είναι βίαιος ποτέ κατά των γυναικών. Και αυτό θα πρέπει να κληθούμε όλοι και να ενθαρρυνθούμε να εφαρμόσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και τώρα τρεις ομιλητές ακόμα για να ετοιμάζονται. Η κυρία Κτένα από την Τουρκία, η κυρία Έλσα Παΐς από την Πορτογαλία και στη συνέχεια η Σάννα Φιροπόβιτς από το Μαυροβούνιο. Από την Τουρκία παρακαλώ, η πρώτη κυρία. Τρία λεπτά. Hello. Γεια σας. Προέρχομαι από την Τουρκία. Είμαστε υποψήφια χώρα και ε, είμαι μέλος του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης ο στόχος είναι τεράστιος να προλάβουμε την βία κατά των γυναικών. Γι' αυτό το λόγο η κυβέρνησή μας υπέγραψε την σύμβαση της Κωνσταντινούπολης ε, το Μάιο του 2011. Έχει υπογραφεί από 27 χώρες και μάλιστα αυτό έγινε το Φεβρουάριο του 2013 αυτή η σύμβαση. Όμως δυστυχώς μέχρι σήμερα μόνο τρεις χώρες την ε, έχουν επικυρώσει την σύμβαση της Κωνσταντινούπολης. Τουλάχιστον αυτό ίσχυε μέχρι το Φεβρουάριο του 2013. Ε, ε, ε, σήμερα έμαθα ότι και η Μάλτα θα επικυρώσει αυτή τη σύμβαση ως τέταρτη χώρα. Ως πρώτη χώρα που επικυρώσαμε τη σύμβαση της Κωνσταντινούπολης είμαστε περήφανοι αλλά ταυτόχρονα έχουμε και μια μεγάλη ευθύνη διότι πριν από τη σύμβαση της Κωνσταντινούπολης η Τουρκία είχε πορεύσει τη ΣΥΝΤΑΦ η οποία ε, έγινε με σημαντικό κομμάτι του δικαίου μας. Από το 1998 διαθέτουμε τον νόμο περί προστασίας οικογένειας και το 2004 ξεκινήσαμε την ε, εκστρατεία stop στην βία εναντίον των γυναικών. 435 εκπαιδευτικά προγράμματα για αυτό το θέμα ξεκίνησαν και ε, ε, μεταξύ των 2009 και 2010. Στο τέλος του 2010 τα εκπαιδευτικά προγράμματα ε, είχαν αγγίξει 60.000 άτομα. Σύμφωνα με την σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, κάναμε σημαντικές μεταρρυθμίσεις στην ομοθεσία μας. Υπ' αυτή την έννοια προετοιμάσαμε και προσαρμόσαμε το νόμο περί προστασίας οικογένειας και της περιπρόληψης των γυναικών, ε, της βίας εναντίον των γυναικών σε συνεργασία με την αντιπολίτευση. Ο νόμος έχει, είχε ως στόχο να προστατευτούν οι γυναίκες και γενικότερα ο πληθυσμός εναντίον της βίας. Ε, δεν φιδόμεθα προσπαθειών προκειμένου να α, αποφύγουμε το φαινόμενο. Ε, όταν ε, ε, οι γυναίκες δεν έχουν κοινωνική ασφάλιση, τα αντίστοιχα, οι αντίστοιχες δαπάνες καλύπτονται από το κράτος. Ε, προβλέπουν, προβλέπει ο νόμος ε, εντολές απομάκρυνσης ή αποφυγής. Επίσης, άτομα τα οποία έχουν υποστεί βία ή κινδυνεύουν, προστατεύονται και με άλλους τρόπους. Καταφύγια, μετακίνησή τους σε άλλη διεύθυνση μέτρα προσωρινής προστασίας ε, για τα θύματα, ε, κοινωνική και ψυχολογική στήριξη και άλλες κοινωνικές υπηρεσίες. Φτάσατε στα τρία λεπτά. Αλλαγή ταυτότητας και άλλων ε, εγγράφων κλπ. Κάποιος για, τα, για τους θύτες, για τους υποψήφιους θύτες επίσης υπάρχουν μέτρα για παράδειγμα απομάκρυνσή τους από την οικογένεια και άλλες. Ευχαριστώ πολύ που μας προσκαλέσατε. Ευχαριστούμε πολύ. Επόμενη ομιλήτρια, κυρία Έλσα Παΐς από την Πορτογαλία. Τρία λεπτά. Κυρίε και κύριοι, κύριε Πρόεδρε, εξ ονόματο τη Πορτογαλική Βουλή, θέλω να συγχαρώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την πρωτοβουλία τη, καθώ και το Ίδρυμα για τα Θεμελιώδη Δικαιώματα, που μα παρουσίασε σήμερα στοιχεία στην ε, διάσκεψη αυτή. Η βία κατά των γυναικών είναι μια σοβαρή παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ήταν μια από τις πρώτες πολιτικές προτεραιότητες της Πορτογαλίας. Από το 1999 έχουμε στρατηγικό σχέδιο για την καταπολέμηση και της ενδοικογενειακής βίας και ε, προγράμματα για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων ή τον ακροτηριασμό των γυναικείων γενετικών οργάνων σε συνεργασία με μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Από το 2002 η ενδογενειακή η ενδοοικογενειακή βία είναι ένα κοινό ε, αδίκημα, ένα αναγνωρισμένο αδίκημα και έγκλημα στην ε, Πορτογαλία. Το 2009 έχουμε ένα νέο πλαίσιο που προσπαθεί να συντονίσει την πρόληψη, την προστασία των θυμάτων και την τιμωρία των ε, δραστών με ηλεκτρονικά μέσα προκειμένου να μπορούν να υποβάλουν τις μαρτυρίες τους τα θύματα και να εντοπιστούν οι διώκτες, οι δράστες. Είναι ένα αναγνωρισμένο λοιπόν έγκλημα ε, η βία ε, στην Πορτογαλία. Η Πορτογαλία ήταν ένα από τα πρώτα κράτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση που αναγνώρισε και κύρωσε την ε, σύμβαση της Κωνσταντινούπολης επίσης. Τώρα, οι προκλήσεις για το μέλλον είναι πολλά θα πρέπει να μας αποσχολήσουν. Έχουμε κάνει πολλά ήδη για, τον, για την πρόληψη, την καταπολέμηση, την προστασία των γυναικών, αλλά πρέπει να προβλέψουμε ως προτεραιότητα στην ημερήσια διαταξή μας και την ενίσχυση της ε, ιδιότητας ε, των πολιτικών δικαιωμάτων και δεν ξέρουμε εάν μπορούμε να κερδίσουμε άλλους αγώνες, εάν δεν γίνει μια πραγματική προσπάθεια για την ευαισθητοποίηση στα θέματα των δικαιωμάτων των πολιτών, της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης και αν αυτό δεν τεθεί στο κέντρο της παιδείας, της εκπαίδευσης και της προσπάθειας ευαισθητοποίησης. Χρειάζεται μια συνολική ενημερωτική εκστρατεία σε ευρωπαϊκό επίπεδο, που να ενισχύει και τις δικές μας εθνικές στρατηγικές ε, κατ' επέκταση. Το θέμα αυτό πρέπει να γίνει ένα θέμα προτεραιότητας σε αυτούς τους καιρούς της διότι η καταπολέμηση της ενδοκενειακής βίας είναι ένας τρόπος ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας, ε, κύριε Πρόεδρε. Οι γυναίκες ε, με τις θέσεις απασχόλησης και με την ε, ενασχόληση με τα παιδιά τους ουσιαστικά προσφέρουν ανταγωνιστικότητα στην οικονομία των ευρωπαϊκών χωρών, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με τη σωστή συμμετοχή τους λοιπόν γίνονται ανταγωνιστικότερες οι οικονομίες μας. Και αυτό το μήνυμα θέλω να περάσει στο Ευρωκοινοβούλιο. Να ενδυναμωθεί μια σφαιρική, συνολική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών. Ευχαριστούμε. Επόμενη μιλήτρια, κυρία Σάντρα Φιλιππόβιτς από το Μαυροβούνιο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι. Είναι για μένα ιδιαίτερη τιμή ευκαιρία που έχω να σας μιλήσω και να σας απευθύνω το λόγο και να σας χαιρετήσω από την Αρμόδια Επιτροπή του Κοινοβουλίου του Μαυροβουνίου. Είναι κοινωνικό πρόβλημα όλων των χωρών μας η ενδοοικογενειακή βία και η γενικότερη βία κατά των γυναικών. Η δική μου χώρα έχει ε, εγκρίνει πρόσφατα σχετική νομοθεσία το 2010 τον Αύγουστο για την προστασία των γυναικών από την οικογενειακή βία που είναι ο πρώτος εξειδικευμένος νόμος που τιμωρεί σε εθνικό επίπεδο ε, αυτά τα φαινόμενα. Αντίστοιχα η στρατηγική ακολούθησε το 2011 για την περίοδο 2011-2015. Στις 25 Νοεμβρίου του 2011 υπογράψαμε ένα πρωτόκολλο για τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να δρουν οι θεσμοί της χώρας σχετικά με την ενδοοικογενειακή βία και αντίστοιχες ε, ε, συμβάσεις και του Συμβουλίου της Ευρώπης. Την 1η Μαρτίου του 2013 εγκρίθηκαν από τη Βουλή του Μαυροβουνίου. Και έτσι ήμασταν από τις πρώτες χώρες που κυρώσαμε αυτή τη ε, σημαντική διεθνή σύμβαση. Οι γυναίκες δίνουν ένα πολιτικό αγώνα από το Δεκέμβριο 2012 και μάλιστα γυναίκες πολιτικοί ε, πρωτοστατούν σε αυτή την προσπάθεια για να καταπολεμηθεί όσο γίνεται περισσότερο η βία κατά των γυναικών και η βία στο σπίτι και στο ε, χώρο εργασίας. Συμμετέχουν βουλευτές, ε, άνδρες και γυναίκες και μέλη όλων των πολιτικών κομμάτων. Έχουμε επίσης νόμο για την προστασία από την βία που βασίζεται στο φύλλο, προστασία των ε, θυμάτων ε, και επίσης κυρώσεις προβλέπονται και επίγοντα μέτρα για να προστατεύονται οι γυναίκες, δικαίωμα σε νομική και ψυχολογική ε, αρρωγή, καθώς επίσης και ιατρική περίθαλψη. Επίσης, ε, οι αρχές και η εισαγγελία, η κοινωνική λειτουργή, ιδρύματα υγείας θα πρέπει να συνεργάζονται και συντονισμένα να προστατεύουν πλήρως τα θύματα ε, της ε, βίας κατά των γυναικών. Έχουμε και καταφύγια και ξενώνες για τις γυναίκες και τα παιδιά τους που είναι στα χέρια και κρατικών θεσμών και ΜΚΟ και δίνουν πραγματικά βοήθεια και καταφύγιο σε αυτές τις γυναίκες. Και τήρησα και το χρόνο μου και σας ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία που μου δώσατε να σας μιλήσω. Ευχαριστώ πολύ. Τι έκπληξη ήταν αυτή. Τελειώσατε νωρίτερα. Πριν εξαντληθεί το τρίλεπτο. Μπράβο σας. Λοιπόν, τώρα έχουμε άλλους δύο μιλητές για αυτό το θέμα. Όσοι έχετε εγγραφεί στον κατάλογο θα μπορέσετε να μιλήσετε και στο επόμενο πάνελ. Θα είστε οι πρώτοι που θα μιλήσετε στο επόμενο πάνελ. Γιατί θα πρέπει να έχουν την ευκαιρία να απαντήσουν και οι κυρίες. Άλλοι δύο και μετά οι υπόλοιποι που δεν έχετε πάρει το λόγο τώρα θα μιλήσετε στη συνέχεια και μάλιστα πρώτοι από το επόμενο πάνελ. Μην ανησυχείτε, δεν σας έχουμε ξεχάσει. Λοιπόν, πρώτος κάποιος από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Μπαλντακίνο και μετά η κυρία Κιουτσούκ από την ε, Τουρκία. Παρακαλώ. Thank you, Mr. President, ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να σας ευχαριστήσω που μου δίνετε το λόγο. Είναι ένα πολύ σημαντικό, ε, μια πολύ σημαντική εκδήλωση αυτή. Κυρίως γιατί περιμένουμε και την Παγκόσμια Μέρα των Γυναικών και οι γυναίκες αυτόν τον καιρό ούτως ή άλλως αντιμετωπίζουν και βία και φαινόμενα προς ενεργεία, περικοπές των μισθών και ούτω καθεξής. Στην Ολομέλεια την περασμένη εβδομάδα εγκρίναμε την έκθεση για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών. Ε, τι έχουμε στα χέρια μας, πέρα από τις ασυντήσεις με τα εθνικά κοινοβούλια και μια συνάδελφο από την Βουλή της Μάλτας, με την οποία μιλήσαμε πριν ξεκινήσουμε επιβεβαιώθηκε, αλλά το είπε και το πανέλ, ότι θα κυρώσει και η Μάλτα την σύμβαση της Κωνσταντινούπολης. Ένα βήμα στη σωστή κατεύθυνση. Πιστεύω πάντως ότι εμείς ως Ευρωκοινοβούλιο πρέπει να έχουμε και να, ε, να, καταρτήσουμε περισσότερες στρατηγικές ε, πλατφόρμες για την καταπολέμηση της βίας πώς με την σύνταξη εκθέσεων, με άλλα μέτρα, όμως πρέπει η φωνή μας να ακουστεί ακόμη πιο δυνατά. Ε, πρέπει να ακουστεί η φωνή των Ευρωβουλευτών του Κοινοβουλίου. Διότι αν δεν ακουστούν αυτά, δεν προβληθούν, δεν προωθηθούν όσα έχουν γίνει στο Ευρωκοινοβούλιο, δεν θα τα ξέρει ε, ο κόσμος, οι πολίτες. Και πρέπει να φτάσουμε στα αυτιά των πολιτών. Πρέπει να αξιοποιήσουμε ακόμη περισσότερο τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Βρισκόμαστε στη γενιά του Facebook. Νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε ώστε το μήνυμα να περάσει τα σύνορα και των 27, των 28 συγγνώμη, κρατών μέλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Και τώρα τελευταία παρεμβαίνουσα η κυρία Κιουτσίκ από την Τουρκία. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχήν να σας πω ποια είμαι. Ονομάζομαι Σεντεφ Κιουτσούκ. Είμαι βουλευτής από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολιτευσής, το Λαϊκό Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Για μας τις ε, γυναίκες βουλευτές του, της Τουρκικής Βουλής, ανεξαρτήτως από που προερχόμαστε, από δεξιά, από τη δεξιά όπως εδώ η συναλφός μου ή από την αριστερά όπως εγώ, θεωρούμε ότι τα θέματα τα σχετικά με τις γυναίκες έχουν προτεραιότητα. Ασφαλώς μπορεί να τα κοιτάμε με διαφορετικό τρόπο και να έχουμε διαφορετικές ιδέες για το πώς θα τα λύσουμε. Όμως οι διακρίσεις εναντίον των γυναικών έχουν, είναι τόσο πολύ ριζωμένες στην κοινωνία μας που οι διαφορές μας δεν έχουν σημασία. Σε όλα τα μέρη του κόσμου, σε όλα τα καθεστώτα και σε όλες τις κοινωνίες ε, υφίσταται ανισότητα μεταξύ των φύλων και η δική μας κοινωνία δεν αποτελεί εξαίρεση. Μάλιστα η Τουρκία έχει και κακό παρελθόν σε ό,τι αφορά τη βία εναντίον των γυναικών. Στην Τουρκία σχεδόν το 50% των γυναικών υφίστανται σεξουαλική, φυσική ή σωματική βία στη ζωή τους. Μόνο πέρσι 228 γυναίκες έχασαν την ε, ζωή τους από τους συντρόφους τους, αδελφούς τους, πατεράδες τους ή συζύγους τους ή ακόμα και από ξένους. 10.000 γυναίκες εκτέθηκαν σε βία. Η βία εναντίον των γυναικών δεν είναι ανεκτή ε, για κανένα πολιτικό ή θρησκευτικό λόγο. Οι γυναίκες μας δεν μπορεί να είναι θύματα της αντίληψης ότι άντρες και γυναίκες δεν μπορεί να είναι ίσοι ή της αντίληψης ότι οι γυναίκες πρέπει να περιορίζονται στο ρόλο της καλής συζύγου, καλής νοικοκυράς και καλής μητέρας. Δεν έχουμε το δικαίωμα ούτε να συγκαλύψουμε, ούτε να, να αναβάλουμε, ούτε ε, να αγνοήσουμε την πραγματικότητα. Πριν από δύο χρόνια, σε συνεργασία μεταξύ της ε, συμπολίτευσης και της αντιπολίτευσης, εγκρίναμε ομόφωνα την σύμβαση της Κωνσταντινούπολης και τον νόμο για την προστασία των γυναικών και της οικογένειας από τη βία θα πρέπει να παραδεχτούμε ότι αυτά είναι σημαντική πρόοδος. Όμως ε, τα ψηφίσματα δεν αρκούν για να λυθούν τα προβλήματα. Ε, υπάρχουν σημαντικές δυσκολίες στην εφαρμογή τους, στην εφαρμογή του νόμου. Ε, κατά την άποψή μου, η όλοι οι κρατικοί αξιωματούχοι, αστυνομικοί, δικαστές, τοπική αυτοδιοίκηση και κυρίως οι πολιτικοί ηγέτες θα πρέπει να αλλάξουν την, τον τρόπο με τον οποίο βλέπουν τα πράγματα. Διότι το, όλο αυτό το θέμα έχει σχέση και με τη δημοκρατία και με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ε, θα πρέπει επίση οι γυναίκε να συμμετάσχουν περισσότερο στην οικονομική ζωή. Είμαι πεπισμένη ότι οι γυναίκε στην Τουρκία και στον υπόλοιπο κόσμο θα μπορούν να ζήσουν πιο ήσυχα και με μεγαλύτερη ασφάλεια την επόμενη φορά που θα συναντηθούμε. Ευχαριστώ. Uh, ευχαριστώ πολύ. Πριν δώσω το λόγο ε, στα μέλη του πάνελ μας για να πατήσουν σύντομα. Ευχαριστώ όλους σας για το σεβασμό του χρόνου. Μπράβο, πολύ ωραία τα πήγατε και συνεχίστε στον καλό δρόμο. Λοιπόν, μπορούν να απαντήσουν οι κυρίες ε, δύο λεπτά Κάστη, Θέλετε να αρχίσετε σας παρακαλώ, κυρία Ερνάντης Ολιβέ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Σημειώνουμε όλες τις τοποθετήσεις και δείχνουν όλες μεγάλη προσήλωση. Από πλευράς της Ισπανίας ένα καταλεκτικό σχόλιο θα έλεγα ότι οι δύο μεγάλοι κίνδυνοι που νομίζω ότι υπάρχουν ε, στη βία κατά των γυναικών στις διάφορες εκφάσεις είναι πρώτον το γεγονός ότι είναι αόρατη, το συζητήσαμε αυτό, ότι είναι αόρατη η βία και σιωπηρή. Η σιωπή των γυναικών είναι πραγματικά ε, πολύ γνωστή. Όλα τα στοιχεία που έχουμε και από τη δική μου χώρα δείχνουν ότι το θέμα αυτό για να αντιμετωπιστεί θα πρέπει να είναι δημόσιο. Κάθε μήνα τα στοιχεία διατίθενται στο κοινό για να γνωρίζει ο κόσμος και κάθε φορά που έχουμε ένα θύμα, μια γυναίκα που χάνει τη ζωή της, αυτό καταγράφεται και καταγγέλλεται. Αυτή η σιωπή είναι ακόμα χειρότερη όταν οι γυναίκες που ε, την αντιμετωπίζουν είναι οι πιο ευάλωτες, ηλικιωμένε, αγρότησες, ε, γυναίκες με αναπηρία, οι κοπέλες οι έφηβες που ακούστηκε το θέμα τους εδώ θα πρέπει να ασχοληθούν μαζί τους. Αυτός είναι ο πρώτος κίνδυνος, ότι αυτή η βία είναι αόρατη. Ο δεύτερος κίνδυνος, πολύ σημαντικός, είναι ότι πιστεύουμε ότι αυτό δεν μπορεί να αλλάξει. Αυτό είναι κίνδυνος, να πιστεύει κάποιο ότι είναι νομοτέλεια, ότι έτσι και αλλιώ πάντα θα υπάρχει αυτό. Και αυτή η αντίληψη είναι η ε, νίκη και ο θρίαβος όλων εκείνων και μιλώ σε αρσενικό γένος, αν και μπορεί και οι γυναίκες να το πιστεύουν, ότι η γυναίκα πρέπει να είναι υποταγμένη στον άνδρα και έτσι να κάνουμε έτσι είναι η ζωή και η νομοτέλεια. Στη χώρα μου αντίθετα πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε ότι μπορεί να αντιστραφεί αυτό, όπως σας είπα να οικοδομήσουμε μια ε, κοινωνία χωρίς βία κατά των γυναικών και με ισότητα. Στην Ισπανία τώρα ολοκληρώνουμε την κύρωση της σύμβασης της Κωνσταντινούπολης. Με μεγάλη χαρά μοιράστηκα το πάνελ αυτό μαζί σας. Ευχαριστώ πολύ πολύ. Yes, please, go ahead. Παρακαλώ. Ευχαριστώ που μου ξαναδίνετε το λόγο. Ήθελα μόνο να εκφράσω κάποιες σκέψεις. Μετά από όσα άκουσα, μου φαίνεται ότι εδώ όσοι έχουμε συγκεντρωθεί συμφωνούμε ότι η βία κατά των γυναικών είναι κυρίως η ενδοοικογενειακή βία. Έτσι μου φάνηκε. Όλοι εδώ γύρω από όλες οι παρεμβαίνουσες είπαν ότι η βία κατά των γυναικών σχεδόν ταυτίζεται με την ενδοοικογενειακή βία. Το βρίσκω παράξενο που κανείς ούτε στην Πορτογαλία δεν κάνει λόγο για την βία των γυναικών που ε, εκπορνεύονται ή των γυναικών που είναι ε, θύματα των δικτύων εμπορίας ανθρώπων. Κυρίες και κύριοι, μιλάμε για την βία κατά των γυναικών και την ισότητα των φίλων Η πορνεία δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται με αδιαφορία. είναι ένα θέμα στα οποία ε, υπάρχουν ε, σοβαροί διαχωρισμοί μεταξύ των πολιτικών κομμάτων. Κάποιοι τα βλέπουν από μία σκοπιά, κάποιοι όλοι. Το λέω για να προκαλέσω και τη σκέψη μας, διότι εργάζομαι στον τομέα αυτό εδώ και 30 χρόνια. 30-40 χρόνια. Γνωρίζω πάρα πολύ καλά το πρόβλημα αυτό. Βλέπω μπροστά μου ε, πρόσωπα κορίτσια που πραγματικά ε, μπορεί να έχουν ε, προβλήματα σοβαρά. Το ε, φαινόμενο αυτό επίσης οδηγεί σε απώλειες ζώων. Οι γυναίκες αυτές που μπορεί να υπονεύονται, οι γυναίκες αυτές που είναι θύματα εμπορίας, πρέπει να μας κάνουν να σκεφτούμε το εξής. Μία γυναίκα στην Ινδία μπορεί να χρειαστεί να πουλήσει το σώμα της για να ε, θρέψει τα παιδιά της. Αλλά δεν είναι αυτή η αρχική, ο αρχικός σκοπός. Ε, μάλλον η γυναίκα μπορεί να χρησιμοποιήσει το σώμα της όπως επιθυμεί. Γι' αυτό δεν φαίνεται να αντιλαμβανόμαστε τη σοβαρότητα του ζητήματος. Επίσης συμφωνούμε ότι ο ακροτηριασμός είναι συνέπεια μιας νόσου, μιας ασθένειας. Ο καθένας μπορεί να χρησιμοποιεί όμως το σώμα του όπως θέλει. Η ενδοκογενειακή βία και το είδαμε εδώ με τις ανησυχίες που εκφράστηκαν και είναι θεμητές οι ανησυχίες αυτές, συμφωνώ απολύτως, η ενδοκογενειακή βία ε, γίνεται αντιληπτή ως βία κατά των γυναικών. Και συμφωνούμε με αυτό. Αλλά τι γίνεται με τη γυναίκα που ε, μπορεί να είναι θύμα ξυλοδαρμού από έρωτα, από τον φίλο της, Αυτά πρέπει να απασχολήσουν τη σημερινή ομάδα που έχει συγκεντρωθεί εδώ. Μιλάμε για ισότητα των φύλων και διάκριτα των γυναικών. Μιλάμε για έναν τρόπο ε, της ε, ποδηγέτησης των γυναικών από τους άντρες. Μιλάμε για την πορνεία που σημαίνει ότι οι γυναίκες γίνονται αντικείμενο εκμετάλλευσης από τους άντρες. Δηλαδή εκπληρώνουν τις ε, σεξουαλικές τους φαντασιώσεις. Και με συγχωρείτε, αλλά ήθελα να πω σε αυτή την ομάδα προσκεκλημένων. Βρισκόμαστε σε ένα θεσμικό όργανο που ε, θα μπορούσε να ασχοληθεί και με το θέμα αυτό και επειδή εργάζομαι σε ένα φορέα με κοινωνικές ανησυχίες στη χώρα μου θα πρέπει να διερωτηθούμε τι γίνεται και με αυτό δεν μπορούμε να το παραβλέπουμε. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε επίπεδο ευρωβουλευτών, μας απασχολεί η έμφυλη βία. Εάν αποσκιοπούμε αυτό το είναι έκφανση της βίας, αυτό το θεσμικό όργανο, δεν θα προχωρήσουμε. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα συμφωνήσω με την ε, παρέμβαση της Πορτογαλίδας, κοινωνικής λειτουργού που προηγήθηκε. Και υπάρχει και μια διάσταση που δεν μπορούμε να παραβλέψουμε στο φαινόμενο που σήμερα συζητούμε. Και Ακριβώς επειδή η οικογένεια ήταν πάντα η αιστεία χώρος που μπορούσε κανείς να είναι ήρεμος και οι συναισθηματικές σχέσεις ήταν ένα καταφύγιο από όσα συμβαίνουν εκτός, Γι' αυτό μας απασχολούν τόσο πολύ αυτές οι εκφάνσεις, τα, οι πτυχές της ενδοκογενειακής βίας. Οι γυναίκες δεν μπορούν ούτε στο σπίτι τους πια να είναι ήσυχες και ήρεμες. Και να εκφράσω και την εξή σκέψη έχοντας ακούσει όσα υπόθηκαν. Φαίνεται ότι υπάρχει γενική συμφωνία ως προς την ανάγκη να υπάρξει κάποια παρέμβαση, να υπάρξει δράση. Αυτό που επιδιώκουμε να κάνουμε στα διάφορα εθνικά κοινοβούλια είναι να δώσουμε σάρκα και οστά στις, ε, προθέσεις, τις νομοθετικές προθέσεις που μπορεί να έχουμε στη δράση που έχουμε σχεδιάσει. Δεν υπάρχουν όμως επίστηκα στατιστικά δεδομένα. Αυτό σημαίνει ότι Κάτι τέτοιο θα πρέπει να προβλεφθεί ως υποχρέωση των κατομελών. Το είπε και η Ισπανίδα ε, συμμετέχουσα που μίλησε προηγουμένω. Δεν υπάρχουν στατιστικά στοιχεία. Μας διαφεύγουν πολλά αριθμητικά στοιχεία. Οι γυναίκε δεν τολμούν να καταγγείλουν ε, τα φαινόμενα αυτά. Μέσω των ε, ε, διαφόρων μηχανισμών που προβλέπονται. Μπορεί να υπάρχουν δικαστικοί μηχανισμοί όπως της αναγκαστικής απομάκρυνσης της προσφοράς ε, καταφυγίου, της ε, αναγκαστικής απομάκρυνσης ενός βίαιου ε, συντρόφου ή συζύγου. Εδώ λοιπόν να πω ότι πραγματικά εμένα με εξέπληξε και ήθελα να το πω αυτό, εξεπλάγει, δεν θυμάμαι το επιθετό σας, με την Ευρωβουλευτή που φάνηκε επιφυλακτική για το κατά πόσον έχουμε αρκετούς, ε, αρκετή νομοθεσία για τα θέματα αυτό. Μα κοιτάξτε, τα κοινοβούλια αυτό κάνουν ακριβώς και σίγουρα η νομοθεσία επηρεάζει και τα ήθη και τα έθιμα. Αυτή είναι η δουλειά της. Και να πω ότι εδώ υπάρχει ένα μήνυμα που είναι δύσκολο να περάσει. Ένα μήνυμα που πολλές φορές το λέμε δειλά. Δηλαδή η κοινωνική και οικονομική ανάκαμψη που τόσο χρειάζονται στην Ευρώπη και την Ιταλία καθώς και η κρίση που γνωρίζουμε σήμερα κάνει τους ανθρώπους πιο επιθετικούς και αυτό έχει επιπτώσεις και στη ζωή των γυναικών και ως προς την πρόνοια επειδή λέμε ότι ε, υπάρχουν ε, γενικά φαινόμενα που επηρεάζουν ε, την συμπεριφορά των ανθρώπων λόγω της κρίσης. Αυτοκτονίες επιχειρηματιών που έχουν καταστραφεί οικονομικά. Γυναίκες που τις εγκαταλείπουν οι σύζυγοί τους. Βλέπουμε ότι και τα ακραία οικονομικά φαινόμενα μπορεί να έχουν αντίκτυπο στην επέκταση των φαινομένων βίας η βία κυρίως όμως κατευθύνεται κατά των παιδιών και των γυναικών. Να μην το ξεχνάμε αυτό. Δουλειά λοιπόν ενός κοινοβουλίου, μιας κυβέρνησης αλλά και της Ευρώπης εφόσον ασχολείται με τα θεμελιώδη δικαιώματα είναι ακριβώς εκεί να παρέμβει. Στο επίπεδο της πρόνοιας, της κοινωνικής πολιτικής χρειάζονται κάποιες δράσεις, κάποιες ενέργειες κοινωνικής πολιτικής που έχουν να κάνουν και με τον πολιτισμό ενός κράτους τον ίδιο. Και είναι πραγματικά εκπληκτικό που κάποια κράτη δεν έχουν καταφέρει να, να κυρώσουν την ε, σύμβαση της ε, Κωνσταντινούπολης. Πολλά τα καταλαβαίνω. Αυτό γιατί, γιατί να μην έχουμε φτάσει στον ελάχιστο ε, αριθμό που χρειάζεται από την άποψη των κυρώσεων για να μπορέσει να λειτουργήσει επιτέλους η σύμβαση αυτή γι' αυτό είμαι αρκετά υπερήφανη. Η Ιταλική Βουλή δεν ήταν και επίκαιρη ακριβώ, αλλά τουλάχιστον δεν καθυστερήσε πάρα πολύ. Ε, στην Ιταλία συνήθω αυτό συμβαίνει. Όταν ερχόμαστε ε, αντιμέτωποι με ένα πρόβλημα, τότε ε, αναγκαζόμαστε να αναλάβουμε τις ευθύνες μας. Αλλά είναι δύσκολο να ε, φέρει κανείς τους βουλευτές σε αυτή την ε, φάση ακριβώς του να, δουν, να έρθουν αντιμέτωποι με ένα πρόβλημα και να μην μπορούν πλέον να υποχωρήσουν. Έτσι λοιπόν ως γυναίκες της Ευρώπης πρέπει να κάνουμε όλη τη δράση που χρειάζεται ώστε τα εθνικά κοινοβούλια να οδηγηθούν να δράσουν πρέπει και στο εσωτερικό του κάθε κοινοβουλίου να ασχοληθούμε με τον προγραμματισμό και την κατεύθυνση όλων των εργασιών προς αυτή την πορεία. Σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα μια ακόμα φορά να ευχαριστήσω τους ομιλητές που συνεισέφεραν στη συζήτηση. Θα κάνουμε αλλαγή φρουράς εδώ. Θα, θα έρθει η κυρία κουδάκι ε, εδώ και εσείς θα εγκαταλείψετε. Okay, dear colleagues, we will now... Λοιπόν, να συνεχίσουμε. Παρακαλώ, καθίστε. Μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου πάνελ θα γίνει μια εισαγωγή εκ μέρους της, ε, του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης πολύ καλό σημάδι που θέλετε να μιλήσετε. Δυστυχώς δεν έχουμε διάλειμμα καφέ, οπότε αρχίζετε να μιλάτε μεταξύ σας. Κι εγώ αν ήμουν από εκείνη τη μεριά το ίδιο θα έκανα. Αλλά πρέπει να συνεχίσουμε. Την περασμένη εβδομάδα εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθετήσαμε ένα νομοθετικό ψήφισμα και σήμερα, κατά σύμπτωση, ο Οργανισμός Θεμελιώδη και Μάλιστα Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, υπέβαλε μια έκθεση ε, που έγινε πάνω σε 42.000 ε, γυναίκες για την έμφυλη βία. Είναι κάτι πρωτοφανές, είναι κάτι καινούριο. Αυτά τα στοιχεία μόλις έχουν βγει από το φούρνο, ζεστά-ζεστά και φρέσκα. Θα δώσω το λόγο στην κυρία Τζοάννα Γκούντι, επικεφαλής του Τμήματος Ελευθεριών και Δικαιοσύνης στον Οργανισμό Θεμελιών Δικαιωμάτων. Σας δίνω 10 λεπτά. Ευχαριστώ. Οι επίσημες στατιστικές για αυτά τα θέματα ε, λείπουν. Γι' αυτό το λόγο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μας ζήτησε και το Συμβούλιο ε, το επιβεβαίωσε να υποβάλουμε μια μελέτη να προετοιμάσουμε μια μελέτη. Και αυτό έγινε πριν από μερικά χρόνια. Τώρα έχουμε τα αποτέλεσματα αυτής της μελέτης. Είναι πανευρωπαϊκή μελέτη για την εμφυλιβία. Με δύο λόγια ε, ήταν ε, ένα τυχαίο δείγμα γυναικών 18-74 ε, ετών σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήρθαμε σε επαφή με μία μόνο γυναίκα σε κάθε νοικοκυριό, τυχαία. Όλες οι συνεντεύξεις έγιναν ζωντανά στο σπίτι τους. Μερικές φορές οι συνεντεύξεις διήρκεσαν μέχρι και δύο ώρες. Χρησιμοποίησαμε... Ε, προσωπικό, γυναίκες, ε, έμπειρες που έπαιρναν τις συνεντεύξεις και χρειαστήκαμε δύο χρόνια ε, να, μελετήσουμε, να κάνουμε την έρευνα και να μελετήσουμε τα αποτελέσματα. Καλύψαμε και τις 28 χώρες και τα 28 κράτη-μέλη. Κάναμε 1.500 συνεντεύξεις ανά κράτος μέλος και συνολικά πήραμε 42.000 συνεντεύξεις από γυναίκες. Τι, ζητήσαμε; τι ρωτήσαμε ρωτήσαμε για τις καθημερινές τους εμπειρίες σε ό,τι αφορά βία, βία περιστατικά. Σωματική και σεξουαλική βία από συντρόφους ή όχι, ψυχολογική βία, επίμονη παρακολούθηση, ε, παρενόχληση, ε, παρενόχληση στον κυβερνοχώρο. Τους ρωτήσαμε τι έγινε για σας, τι, τι σας συνέβη πριν κλείσει τα 15 χρόνια από ενήλικους, ε, τις ρωτήσαμε αν γνωρίζουν τον νόμο και τα δικαιώματά τους και, τους, ε, και τις ρωτήσαμε τις εμπειρίες τους ε, μετά τα 15 και τους τελευταίους 12 μήνες ιδιαίτερα. Τα αποτελέσματα. Ε, μία στις τρεις γυναίκες κατά μέσο όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν θύμα ψυχο, σωματικής ή σεξουαλικής βίας από τα 15 τους και μετά. Το 8% των γυναικών τους τελευταίους 12 μήνες. 22% των γυναικών έχουν δεχτεί, ε, ήταν θύματα βίας από το σύντροφό τους. 11% των γυναικών έχουν γίνει θύματα κάποιου τύπου σεξουαλικής βίας. 5% από τις 42.000 γυναίκες δήλωσαν ότι έχουν βιαστεί. Μία στις δύο γυναίκες είπε ότι έχει δεχτεί σεξουαλική ε, ε, κακοποίηση και μία στις πέντε τους τελευταίους 12 μήνες. Τι τις ρωτήσαμε. Τις ρωτήσαμε ε, του κάνω μια σειρά ε, ερωτήσεων για συγκεκριμένα περιστατικά βίας. Αν του, τις ε, έχουν σπρώξει, αν τι έχουν χαστουκίσει, αν τους έχουν πετάξει ένα σκληρό αντικείμενο, αν τι έχουν τραβήξει από τα μαλλιά, αν τους, έχουν χτυπήσει με τη γροθιά, αν έχουν γροθοκοπηθεί δηλαδή, αν τις έχουν κάψει, αν έχουν προσπαθήσει να τις πνίξουν, να τις κόψουν κλπ. Ακόμα και αν βγάλουμε την πρώτη κατηγορία τους προξήματος που είναι ίσως χαμηλό κατόφλι βίας, μία στις τέσσερις γυναίκες, 25% των γυναικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση λένε ότι έχουν, ήταν θύματα τουλάχιστον μία από αυτές τις υπόλοιπε πράξεις. Σεξουαλική βία από σύντροφο ή μη σύντροφο από την ηλικία των 15 ετών και μετά. Και πάλι ρωτήσαμε 42.000 γυναίκες. Ε, εξαναγκαστήκατε σε σεξουαλική πράξη από κάποιον που σας ε, συγκρατούσε με τη βία. Ε, ε, σας αναγκαστήκατε να λάβετε μέρος σε σεξουαλική δραστηριότητα χωρί, χωρίς να το θέλετε επειδή δεν μπορούσατε να ανοιχτείτε κλπ. 9 εκατομμύρια γυναίκες στο σύνολο στο σύνολό τους ε, σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, αντιστοιχούν στις ε, θετικές απαντήσεις του βιασμού. Ο μέσος όρος είναι περίπου 11% σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τουλάχιστον μία πράξη σεξουαλικής βίας. Τώρα, κατευθύνονται οι γυναίκες, πού καταφεύγουν οι γυναίκες σε τέτοιες περιπτώσεις σεξουαλικής βίας. Ε, ρωτήσαμε με ποιον έρχεστε σε επαφή σε περιπτώσεις σεξουαλικής βίας από ε, το σύντροφό σας. Σε μεγάλη πλειοψηφία στις υπηρεσίες υγείας. Νοσοκομεία ή άλλες υπηρεσίες υγείας. Εκεί πηγαίνουν καταρχήν. Πολύ λιγότερες στην αστυνομία. Ε, ακόμα λιγότερες σε καταφύγια ε, για γυναίκες ή για ε, κοινωνικές υπηρεσίες ε, προστασίας που είναι πολύ λίγες ενδεχομένως στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα πιο σημαντικά περιστατικά όμως τα αναφέρουν στους γιατρούς, στα κέντρα υγείας, γιατί αυτά είναι και τα πιο κοντινά τους. Τις ρωτήσαμε για την επίμονη παρακολούθηση, το stalking. Ε, όταν ε, ένα συγκεκριμένο άτομο επιμένει να σε παρακολουθεί ή να σε απειλεί. Παραδείγματα ε, επίμονης παρακολούθησης που δώσαμε ήταν κάποιος να σε περιμένει έξω από το σπίτι σου, έξω από τη δουλειά σου χωρίς συγκεκριμένο σοβαρό λόγο, να σε παρακολουθεί συνεχώς, να, κάνει, να σου κάνει τηλεφωνήματα χωρίς να μιλάει κλπ. Το αποτέλεσμα 18% των γυναικών έχουν υποστεί επίμονη παρακολούθηση μετά την ηλικία των 15, 5% των γυναικών τους τελευταίους 12 μήνες. Ορισμένες γυναίκες ε, τυχάνουν παρακολούθηση παρακολούθησης ε, για πάνω από δύο χρόνια, μία στις πέντε συγκεκριμένα και το 23% των θυμάτων άλλαξαν το, τη διεύθυνση email τους ή το τηλέφωνο, αριθμό του τηλεφώνου τους σε, πιο σοβαρές περιπτώσεις. Πρέπει να δούμε λοιπόν και άλλες περιπτώσεις βίας κατά, στον, κατά των γυναικών. Ε, σεξουαλική ε, παρενόχληση ε, Έχουμε αυτό μπορεί να κυμαίνεται από μια, ε, ένα απλό άγγιγμα ανεπιθύμητο όμως μέχρι ε, σεξουαλικά σχόλια, προσβλητικά σχόλια ή λήψη SMS ε, ε, που είναι και αυτά προσβλητικά και, δεν είναι, και είναι επίσης ανεπιθύμητα, με σεξουαλικά υπονοούμενα κλπ. Έχουμε στοιχεία για κάθε μία από αυτές τις κατηγορίες, έτσι. το ε, πάνω, από το 50% των γυναικών έχουν ε, υποστεί ε, τέτοιου είδους βία. Μία στις ε, πέντε τους τελευταίους 12 μήνες πριν την ε, ε συνέντευξη. 32% των θυμάτων αναφέρουν ότι ο θήτης ήταν το αφεντικό, ένας συνάδελφος ή ένας πελάτης. 75% των γυναικών σε θέσεις, υψηλές θέσεις ε, αναφέρει ότι ε, έχει ε, υποστεί αυτή την πράξη. 20% των νέων γυναικών, 18 με 29 ετών, έχουν υποστεί αυτή την πράξη μέσω του ίντερνετ. Μέσω δηλαδή SMS κλπ. Κατόπιν, βία κατά τη διάρκεια της παιδικής ηλικίας τι μας είπαν οι γυναίκες για την σεξουαλική κακοποίηση που έχουν δεχτεί ως παιδιά. Γιατί δεν ρωτήσαμε τις ε, γυναίκες μόνο για το τι του συνέβη μετά τα 15, αλλά και τι του συνέβη πριν τα 15 από ενήλικες. Ε, μας λένε ότι όταν ήταν παιδιά, ένας ε, ενήλικος τους εξέθεσε τα γεννητικά του όργανα 8%, τους ανάγκασε να ε, ποζάρουν γυμνές μπροστά σε φωτογραφική μηχανή 1%, τους άνοιξε τα γεννητικά όργανα στο στήθος 5%, ε, τους εξανάγκασαν να αγγίξουν, τις εξανάγκασαν να αγγίξουν γεννητικά όργανα άλλου 1% κλπ ή τις ανάγκασαν σε ερωτική πράξη. 1% συγκεκριμένα είπε ότι εξαναγκάστηκε σεξουαλική πράξη ως παιδί. 12% του συνόλου ε, ήταν θύμα μιας τουλάχιστον από αυτές τις ε, πράξεις. Και το 90% των θητών ήταν άντρες. Τι μπορεί να γίνει. Πρόληψη. Ε, απαντήσεις σε ό,τι αφορά την πρόληψη, αλλά σε διάφορα επίπεδα. Ε, πολιτική εκπαίδευση, διάφοροι καινούργιοι τρόποι μέσω του ίντερνετ κλπ. Ε, γιατί όταν μιλάμε για πρόληψη πρέπει να κάνουμε ένα βήμα πίσω και να δούμε πώς μπορούμε να αποφύγουμε εξ αρχής τη βία. Γιατί τώρα έχουμε μια ε, πολύ σαφή εικόνα της ε, κατάστασης στην Ευρώπη και δεν είναι καθόλου καλή. Ε, τα στοιχεία μας είναι διαθέσιμα ε, μέσω του ιστοτόπου μας και μπορείτε να τα συμβουλευτείτε. Ευχαριστώ. That Ακριβώς 10 λεπτά. Διάνα. Ε, δηλαδή με ακρίβεια δευτερολέπτου. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε και μας ενημερώσατε. Και όταν σας άκουσα ίδιος σήμερα το πρωί, σκέφτηκα αμέσω ότι είναι πάρα πολύ πολύτιμη αυτή η πληροφόρηση για μας, ιδιαίτερα στη χάραξη πολιτικής. Γιατί Περιμέναμε πάρα πολύ τα στοιχεία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν θέλει να πετύχει κάτι, αν θες να αλλάξει κάτι, θα πρέπει να γνωρίζει πώ έχει πρώτα απ' όλα η κατάσταση. Και τα στατιστικά στοιχεία είναι πάρα πολύ σημαντικά ω φωτογράφηση, να ξέρουμε πώ έχει η πραγματικότητα, μία αποτύπωση για να δει από εκεί και πέρα τι πρέπει να κάνει και ποια είναι τα καλύτερα εργαλεία για να το αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα. Νομίζω λοιπόν ότι θα είναι τεράστια η χρησιμότητα για πολλούς και για εμάς τους πολιτικούς και για την κοινωνία των πολιτών των στοιχείων αυτών. Σας ευχαριστώ πολύ. Και περνάμε στο επόμενο πάνελ. Θα το, έχουμε την ευκαιρία να ανταλλάξουμε απόψη για τις διάφορες ε, δυνατότητες δράσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, πάντα στην καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών. Όπω είπα προηγουμένω, την περασμένη εβδομάδα με μεγάλη πλειοψηφία ενέκρινε μια έκθεση πρωτοβουλία στο Κοινοβούλιο νομοθετικού περιεχομένου της κυρίας Παρβάνοβα ήταν η έκθεση για συγκεκριμένες προτάσεις νομοθετικής φύσεως σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Έχουμε τρει κυρίες και πάλι στο πάνελ. Θα ακούσουμε πρώτα την κυρία Ντανιέλα Μπανκέ που είναι ε, η ε, Διευθύντρια ε, Ισότητα στη Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ που με προσκαλέσατε σήμερα σε αυτή την ε, διακυβνοβουλευτική συνεδρίαση και τη συζήτηση για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών. Ευχαριστώ που προβλέψατε αυτή την εκδήλωση, τη δυνατότητα να συναντηθούμε και να συζητήσουμε αυτό το τόσο σοβαρό ζήτημα. Κυρίες και κύριοι, καθημερινά γυναίκες και κορίτσια είναι θύματα εξευτελισμού, εκφοβισμού, επιθέσεων, ακροτηριασμού των γενετικών τους οργάνων, ξυλοδαρμών ή φόνου, επειδή είναι γυναίκες ή απλά νεαρά κορίτσια. Συμβαίνει παντού αυτό, ε, σε κάθε χώρα εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η μελέτη που δημοσιεύτηκε σήμερα από τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων μας λέει ότι μία στις τρεις γυναίκες στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πέσει θύμα κάποιας μορφής σεξουαλικής ή σωματικής βίας από την ηλικία των 15 ετών. Η μελέτη επίσης δείχνει το θέμα της έλλειψης στοιχείων, διότι μόνο ένα στα τρία θύματα της έμφυλης Βία το καταγγέλει. Το πιο και αναφέρουν, αναφέρουν μόνο τα σοβαρότατα περιστατικά, ε, τα πιο πρόσφατα και σοβαρά περιστατικά στην αστυνομία της άλλες ε, δυνάμεις καταστολής. Άρα αυτό δείχνει ότι έχουμε περιορισμένη γνώση του συνόλου του φαινομένου. Επίσης η μελέτη ρίχνει φως στις διαφορές μεταξύ κρατών μελών σε ό,τι αφορά τις εμπειρίες ε, της βίας, την απόκριση της πολιτική, εκπόνησης πολιτικής και το πώς αντιδρούν οι υπεύθυνοι φορείς. Αλλά και ως προς τις νέες μορφές βίας, τις οποίες να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή στο μέλλον, όπως τη βία στον κυβερνοχώρο ή τις μορφές βίας με νέα τεχνολογικά μέσα. Η βία κατά των γυναικών οπωσδήποτε παραμένει ένα από τα πλέον διαδεδομένα φαινόμενα παραβίασης των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Είναι αποτέλεσμα ιστορικών α, ε, ε, άνησης κατανομής ε, της εξουσίας μεταξύ ανδρών και γυναικών. Η ιδέα των γυναικών οδηγεί στην διόνυση της ανισότητας των φύλων, επηρεάζει την κοινωνία στο σύνολό της και έχει πολύ μακροχρόνιες συνέπειες σε ό,τι αφορά την απασχόληση των γυναικών, την οικονομική τους κατάσταση και την κατάσταση της υγείας τους και όχι μόνον. Σε ό,τι αφορά λοιπόν την βία κατά των γυναικών, πολλές φορές διαπράτεται από κάποιο γνωστό σύντροφο, μέλος της οικογένειας ή και οι γυναίκες που έχουν ε, γνωρίσει τη βία πολλές φορές έχουν συναισθηματική εξάρτηση από τον ε, επιτιθέμενο ή πολλές φορές έχουν οικονομική εξάρτηση από αυτόν. Σε πολλές περιπτώσεις το θύμα πέφτει επανειλημμένος θύμα της βίας με συγκεκριμένους κύκλους που γνωρίζουν μια περίοδο ηρεμίας ή την επιστροφή του επιτιθέμενου. Πολλές φορές ε, βρίσκεται σε σύγχυση το θύμα γνωρίζοντας ε, ένα συνδυασμό αγάπης, ενοχής, ε, θλίψης και πολλές φορές είναι ένα κοινωνικό στίγμα η βία, ε, γιατί υπάρχει και η περίπτωση να γίνει γνωστό ε, το θέμα αυτό ή πολλές φορές θεωρείται κάτι το τετριμένο, το καθημερινό, ε, επειδή το γνωρίζει σε συστηματική βάση. Πολλές φορές το θύμα αποσιωπά τη βία και δύσκολα ζητά βοήθεια από τις αρχές της αρμόδιες υπηρεσίας. Οι καταγεγραμμένες υποθέσεις είναι μόνο ένα μικρό ποσοστό του συνόλου του φαινομένου. Κυρίες και κύριοι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι κάνει για να αντιμετωπίσει τη βία κατά των γυναικών. Κατά πρώτον, να θυμίσω ότι η βία είναι μία από τις πέντε προτεραιότητες στην πολιτική για την ισότητα των φύλων όπως έχουν οριστεί στη στρατηγική μας για την ισότητα των φύλων που καλύπτει τα έτη 2010 2015. Η βία λοιπόν κατά των γυναικών έχει μια προεξάρχουσα θέση μεταξύ των προτεραιοτήτων των πολιτικών μας. Σε ό,τι αφορά τα εργαλεία μας, να τονίσω ότι στις ιδρυτικές συνθήκες δεν υπάρχει συγκεκριμένη νομική βάση για να καταπολεμήσουμε την βία κατά των γυναικών. Η κατεξοχήν λοιπόν ευθύνη είναι ευθύνη των κρατών μελών. Η ευθύνη για την πρόληψη, την τιμωρία των εγκληματικών ενεργειών, την προστασία και τη στήριξη των θυμάτων της βίας. Πέραν όμως αυτού, να τονίσω και το εξής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει πραγματικά ασχοληθεί εντατικά με την ε, αξιοποίηση των αρμοδιότητων σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να στηρίξει τα κρατημέλη στην πρόληψη και την καταπολέμηση όλων των μορφών της βίας κατά των γυναικών. Δική μας φιλοδοξία είναι να διασφαλίσουμε ότι όλες μας οι δράσεις συμπληρώνουν τις εθνικές και να μπορέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να υποφεληθεί από την προστιθέμενη αξία που παράγεται. Ένα σημαντικό βήμα σε αυτή την κατεύθυνση είναι να βελτιώσουμε τη γνώση του συνόλου του φαινομένου της βίας Γι' αυτό η μελέτη που ετοίμασε το Ίδρυμα για τα Θεμελιώδη Δικαιώματα είναι για μας πολύ σημαντική. Συνεργάζεται με όλους τους ε, αρμόδιους φορείς, τη Eurostat, το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για την Ισότητα των Φύλων στο Βίλνιους, τον Οργανισμό για τα Θεμελιώδη Δικαιώματα, όπως είπα, για να έχουμε όλο και περισσότερες πληροφορίες για το φαινόμενο της βίας. Μόνο με περισσότερες πληροφορίες και δεδομένα μπορούμε να εκπονήσουμε τις κατάλληλες πολιτικές και να καταγράψουμε το τι πρόοδος επιτελείται. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επίσης ε, αντιμετωπίζει την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών από τη σκοπιά της καταπολέμησης της ανισότητας των φύλων και της διακριτικής μεταχείρισης στα πλαίσια των ευρωπαϊκών πολιτικών γενικότερα. Τα θύματα της βίας πρέπει να ε, προστατεύονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πρέπει να υπάρχουν νόμοι για την δίωξη των ε, δραστών και την προστασία των θυμάτων. Έχουμε εγκρίνει ένα συνολικό νομικό πλαίσιο για πολιτικά και ποινικά ζητήματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το πλαίσιο αυτό συμπεριλαμβάνει οδηγία για την εμπορία ανθρώπων, που πολύ συχνά είναι γυναίκες, μια οδηγία κατά της σεξουαλικής ε, παρενόχλησης, εκμετάλλευσης και χρήσης των ε, παιδιών και την παιδική πορνογραφία, το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψη για ποινικά ζητήματα με κανονισμό που ισχύει σε περιπτώσει δικαιωμάτων των πολιτών και εξίσου σημαντικό, πιο πρόσφατο, η οδηγία για τα δικαιώματα των θυμάτων εγκληματικών ενεργειών Τονίζεται εκεί η ανάγκη για την παροχή προστασίας σε θύματα έμφυλης βίας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτή τη στιγμή συνδράμει τα κρατημέλη στην υλοποίηση της, ε, του νομικού αυτοπλαισίου σε εθνικό επίπεδο και ε, καταμετρούμε την πραγματική μεταφορά του. Η Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης που αναφέρθηκε ήδη σήμερα για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και την ενδοοικογενειακή βία. Είναι ένα άλλο σημαντικό νομοθέτημα το οποίο θα επιτρέψει να έχουμε περισσότερη πρόοδο στον τομέα που μας αφορά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκμεταλλεύεται κάθε δυνατή ευκαιρία για να απευθύνει εκκλήσει στα κράτη-μέλη, ώστε το καθένα ξεχωριστά να κυρώσουν αυτή τη σύμβαση. Παρακαλώ, ενθαρρύνετε τα εθνικά σα κοινοβούλια, τι κυβερνήσει σα, να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα ώστε να κυρωθεί επιτέλου αυτή η σύμβαση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι αποφασισμένη να αξιοποιήσει πλήρω τα ε, το πρόγραμμα για τα νέα δικαιώματα, την ηθαγένεια και την ε, ιδιότητα των πολιτών ώστε να διοργανώσει ε, ενημερωτικές εκστρατείες, συστηματική ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και να παράσχει χρηματοδότηση σε κυβερνήσεις με κυβερνητικές οργανώσεις και δίκτυα που ασχολούνται με την πρόληψη και την εξάλληψη κάθε μορφής βίας. Τέλος, θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας στην πρόσφατη ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που εγκρίθηκε προσφάτως για την εξάλληψη του φαινομένου του ακριτοριασμού των γυναικείων γενετικών οργάνων. Το ε, φαινόμενο αυτό είναι ένα φαινόμενο κατάφορης παραβίασης των δικαιωμάτων των γυναικών και παιδικής ε, κακοποίησης. Ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης έχουν προβλέψει εξωτερικά και εσωτερικά μέτρα ώστε να έχουμε μια καλύτερη κατανόηση του φαινομένου αυτού, να υπάρξει πρόληψη του φαινομένου με τη συνεργασία των κοινοτήτων των θυμάτων και να παράσχουμε και προστασία στα θύματα με την πολυτομεακή συνεργασία με την πραγματική δίωξη του φαινομένου αυτού της κλειτοροδεκτομής στα κράτη-μέλη και με την παροχή στήριξης στα θύματα αλλά και την προληπτική δράση στα, στις περιοχές του κόσμου το φαινόμενο αυτό απαντάται ακόμη με τις ακόλουθες δράσεις που έχει προβλέψει. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύεται να ε, καταμετρά και να σημειώνει την πρόοδο που έχει επιτελεστεί σε διάφορες δράσεις όπως τις έχουμε ορίσει στην ανακοινωσή μας επισίως. Ολοκληρώνοντας, να πω ξανά ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι αποφασισμένη να συνεχίσει να στηρίζει τα κράτη-μέλη στην προσπάθεια εξάλληψης οποιασδήποτε μορφής βίας κατά των γυναικών. Θέλουμε να έχουμε στοχευμένες και συνεπείς πρωτοβουλίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θέλουμε να αξιοποιήσουμε πλήρως τι αρμοδιότητε της Ευρωπαϊκής Ένωση σε αυτόν τον τομέα. Πιστεύουμε ότι τόσο η δράση όσο και η συνεργασία σε όλου του τομεί είναι καθοριστική σημασία. Να συνεχίσουμε λοιπόν να συνεργαζόμαστε στενά για να εξαλείψουμε τελείω την μορφή της έμφυλης, τη κάθε μορφή έμφυλη βίας στην Ευρώπη. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σα. Σα ευχαριστώ πολύ, Ντανιέλα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι παρευρίσκεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και απευθύνεται σε εμά και επίσης ομιλεί για τις απόψεις και τις πράξεις της. Ε, ε, χαίρομαι πάρα πολύ που ε, βρήκε το χρόνο και ήρθε να μας μιλήσει να μας εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και τώρα θα περάσουμε στην επόμενη ομιλήτρια που είναι η κυρία Σίλβια Γουόλμπι, καθηγητής κοινωνιολογίας στην έδρα της UNESCO για ε, έρευνα φύλου στο Πανεπιστήμιο Λάνκαστερ του Ηνωμένου Βασιλείου. Έχετε το λόγο παρακαλώ για ένα δεκάλεπτο. Σας ευχαριστώ πολύ. Σήμερα θα σας μιλήσω για τρεις εργασίες που κάναμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση. πρώτο το κόστος της βίας κατά των γυναικών. Δεύτερον, τις ε, νομικές πρόπτικες. Υπάρχουν πολλές ε, πρόπτικες βέβαια. Και το τρίτο έχει να κάνει με μια επισκόπηση για την πολιτική αυτή παγκοσμίω. Λοιπόν, θα εξετάσω πέντε διαφορετικούς τρόπους αντίληψης και σκέψης για στρατηγική δράση για να τερματιστεί η βία κατά των γυναικών. Θα αρχίσω από τα νομικά ζητήματα και θα συνεχίσω με τα οικονομικά που είναι η πιο παραδοσιακή αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ασχοληθώ λίγο ε, με την ισορροπία των φύλων σε θέση λήψη αποφάσεων, την έρευνα και τη στρατηγική, ε, στρατηγικό σχεδιασμό. Πρώτον, το νομικά λοιπόν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει μία σειρά οδηγιών τα τελευταία χρόνια που έχουν να κάνουν με τη βία κατά των γυναικών. Έντολες προστασίας, τράφικινγκ, σεξουαλική κακοποίηση παιδιών, δικαιώματα θυμάτων αλλά και τα θέματα της παρενόχλησης που είναι παλαιότερα ε, αλλά και που συνιστούν κατά κάποιο τρόπο και αυτά βία κατά των γυναικών. Πώς θα προχωρήσουμε. Δύο είναι οι στρατηγικές εναλλακτικές λύσεις και τις βλέπουμε μπροστά μας. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέλει το άρθρο 2.25, θέλει μεγάλη δράση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να γίνει η μεγάλη αρχή, να αρχίσουμε και πάλι ε, να σκεφτόμαστε ε, μια δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ευρεία. Η άλλη προσέγγιση είναι η βαθμία και σταδιακή, βήμα-βήμα, ε, με οδηγία μετά την οδηγία για να δημιουργηθεί μια ισχυρή βάση και βαρύ και να φτάσουμε στον ίδιο στόχο. Είναι κάπως διαφορετικές οι στρατηγικές και τις βλέπετε να κάθονται μπροστά σας ε, των διαθεσμικών οργάνων. Εάν μου επιτρέψετε τώρα να πάω στα επόμενα μικρά βήματα, θα μπορούσαμε να πούμε για παράδειγμα ότι ε, στη συνθήκη της Λισαβόνας και τη συνθήκη της λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχουν τα άρθρα 82 και 83 και μπορείτε να δείτε αρμοδιότητες για θέματα ποινικού δικαίου. Ποια είναι η πρόθεση εδώ, να υπάρχει ένας κοινός χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, έτσι ώστε να υπάρχει και αμοιβαία αναγνώριση ε, των δικαστικών αποφάσεων. Και για να το καταφέρει κανείς αυτό χρειάζεται ελάχιστες προδιαγραφές και κοινά πρότυπα για ε, να ξέρουμε ότι πάνω κάτω ε, μιλάμε για το ίδιο πράγμα και έχουμε τα ίδια πρότυπα. Λοιπόν, για να δούμε και μερικά άλλα στοιχεία σχετικά. Και να μην ξεχνάμε και τον νόμο περί των διακρίσεων. Το δίκαιο αυτό έχει αναπτυχθεί πολύ ε, ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπό όρους ε, ίσης αμοιβή για ίδια εργασία. Θα μπορούσε ένα είδος βίας που ονομάζεται παρενόχληση να ενταχθεί εδώ και η σεξουαλική και η παρενόχληση λόγω του φίλου. Η βία κατά των γυναικών που βασίζεται στο φύλλο είναι ένα υποσύνολο της σεξουαλικής παρενόχλησης και θα μπορούσε να γίνει αντιληπτή με τον ίδιο τρόπο αλλά είναι μάλλον μια μικρή εμ, πτυχή παρά μεγάλη. Ποια είναι οι περιορισμοί εδώ, όπως γνωρίζετε. Ποια είναι τα όρια του επίπεδου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στα κράτη-μέλη δεν υπάρχουν όρια σε εθνικό επίπεδο για την νομοθεσία, αλλά σε ευρωπαϊκό είναι συγκεκριμένα τα πράγματα που μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι θα μπορούσατε να κάνετε, ας πούμε, στη σταδιακή προσέγγιση. Να δούμε το βιασμό. Όταν ένας βιαστής φεύγει από μια χώρα, ε, ε, ε, μάλλον ο φερόμενος για να είμαστε σωστοί, που έχει κατηγορηθεί για βιασμό, φεύγει από μια χώρα και πάει σε μια άλλη χώρα. Μπορεί κανείς να θεωρήσει ότι θα ισχύσουν οι ίδιοι στην άλλη χώρα. Πρόσφατα είχαμε πολύ μεγάλη αντιπαράθεση γι' αυτό για περιπτώσεις που χρειάστηκαν μήνες να λυθούν. Δεν θα ήταν καλύτερο να έχουμε ισότητα έτσι, δικαστική με αμοιβαία αναγνώριση των δικαστικών αποφάσεων, ας πούμε στο θέμα της ε, υπόθεσης του βιασμού. Έτσι από μικρά βήματα να μην υπάρχει ε, εξαίρεση, να υπάρχει ένα ελάχιστο όριο. Υπάρχει ας πούμε χώρος ε, για να έχουμε μια οδηγία για το βιασμό όπως ε, είναι εντολή προστασίας και η προστασία των θυμάτων από τράφικινγκ. Ε, το αντίστοιχο θα μπορούσε να γίνει για την ενδοοικογενειακή επίθεση. Κάθε χώρα έχει νόμους σχετικά. Δηλαδή είναι ποινικά κολάσιμο να βιοπραγείς εις βάρος κάποιου. Ε, ορισμένες χώρες δέχονται εξαίρεση εντός του γάμου. Για ποιο λόγο. Κανείς δεν θεωρεί ότι χρειάζεται κάτι τέτοιο. Θα πρέπει να υπέλθει δικαστική επίσης ε, σαφήνεια και να λέει η ε, οδηγία ότι δεν εννοείται βιοπραγία εντός γάμου ή εντός οικογενείας. Αυτά είναι λοιπόν παραδείγματα για να δείξουμε πώς μπορεί να συνεχιστεί αυτή η σταδιακή υιοθέτηση ε, οδηγιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ε, στη συνέχεια με δέσμες να ε, έχουμε τη σωστή εφαρμογή παντού. Θα ήθελα και πάλι να πω ότι η βία που έχει βάσει το φύλλο συνδέεται πάρα πολύ στενά με την παρενόχληση για λόγους φύλου που υπάρχει ε, η διαναγνωρισμένη ε, αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ας πούμε στο εργατικό δίκαιο ή ε, στην πώληση και διανομή αγαθών και υπηρεσιών. Θα μπορούσαμε να το επεκτείνουμε λίγο παραπάνω, ίσως βάσει του άρθρου 19. Αυτή είναι η σταδιακή προσέγγιση. Αυτό που θέλει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με το ψήφισμα είναι να ορίσουμε έναν τομέα. Η έμφυλη βία είναι ένα πεδίο που θα πρέπει να νομοθετήσουμε και να έχουμε οδηγία πάνω σε αυτό. Αυτό είναι ένα βήμα ίσως ριζοσπαστικό που θέλει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αλλά είναι η άλλη προσέγγιση. Έρχομαι τώρα στην οικονομία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε μακρά αρμοδιότητα για την οικονομία και παραδοσιακά ήταν το θέμα της ίσης αμοιβή για ίδια εργασία. Και εκεί βασίστηκε η ισότητα του φύλου για να προχωρήσει αυτή η υπόθεση. Η βία κατά των γυναικών είναι ένα μειονέκτημα για την οικονομία, βλάπτει την οικονομία, βλάπτει την δυνατότητα εργασίας των γυναικών. Άρα είναι και οικονομικό ζήτημα και μπορούμε να το κάνουμε ευρωπαϊκή αρμοδιότητα στα πλαίσια της οικονομίας. Να δούμε ας πούμε τι γίνεται με τους ανθρωπίνους πόρους στην οικονομία και πώς αυτοί βλάπτονται. Το άρθρο 153, επανένταξη στην αγορά εργασίας. Εντάξει, ιστορικά αυτό είναι για τον άνθρακα και το χάλιβα, Αλλά το θέμα είναι πώς μπορούν οι γυναίκες να ενταχθούν. Τι γίνεται με τα ευρωπαϊκά διορθωτικά ταμεία. Υποτίθεται ότι και αυτά έχουν να κάνουν με οικονομική διάσταση. Δεν θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν. Όπως έχει γίνει στην Ελλάδα, ας πούμε, για να συμμετέχουν περισσότερο γυναίκες στην οικονομία. Ε, μήπως μπορούμε να ανατρέξουμε ακριβώς στα κονδύλια αυτά και ευρύτερα και αποτελεσματικότερα να τα χρησιμοποιήσουμε. Οι μεγάλες ευρωπαϊκές οικονομικές κατευθυντήριες γραμμές δεν θα μπορούσαν να αναγνωρίσουν ότι η βία κατά των γυναικών ε, συνιστά ζημία κατά της ευρωπαϊκής ε, οικονομίας. Μπορούμε να το προεκτείνουμε και να το προβάλλουμε και με βάση τη Βρετανική εμπειρία. 228 δισεκατομμύρια ευρώ ε, υπολογίζεται αυτή η ζημία ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ορίστε, η οικονομία είναι ένας κατεξοχήν κλάδος που έχει αρμοδιότητα η Ευρωπαϊκή Ένωση και θα μπορούσε κανείς με τρόπο καινοτόμο να συμπελάβει και αυτά τα στοιχεία του φύλου. Έρχομαι τώρα στην έρευνα. Πολλοί λέγουν ότι θα χρειαζόμαστε περισσότερη έρευνα. Να την έχουμε, ωραία. Τι γίνεται με τον ορίζοντα του 2020. Υπάρχει εκεί πουθενά το φύλλο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να το εντοπίσει κανείς στο μεγάλο ερευνητικό πρόγραμμα. Ίσως την επόμενη φορά να βάλουν περισσότερο gender mainstreaming, δηλαδή περισσότερα θέματα φύλου και της βίας κατά των γυναικών στα ερευνητικά προγράμματα. Δηλαδή λίγο παραπάνω για την αρμοδιότητα η ισορροπία του φίλου στη διαδικασία ε, λήψης των αποφάσεων. Ο ΙΕ το έχει ζητήσει αυτό στι ένοπλες σειράξει. Ξέρουμε ότι είναι σημαντικό να συμμετέχουν οι γυναίκες στην επίλυση διαφορών και ε, ιδιαίτερα ε, μειώνοντας έτσι και τη βία κατά των γυναικών. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να προχωρήσουμε, η μεγάλη η ριζοσπαστική, η μικρή, τα σταδιακά βήματα, αλλά δεν είναι μόνο θέμα νόμου, είναι και οικονομίας και ισορροπίας ε, φύλου στη λήψη των αποφάσεων, στρατηγικό σχεδιασμός και περαιτέρω έρευνα χρειάζεται. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank you very much. Σας ευχαριστώ πολύ. Ήταν πάρα πολύ συγκεκριμένες, εξαιρετικά συγκεκριμένες οι προτάσεις σας. Μετά από αυτό δεν μπορεί κανείς να έρθει να ρωτήσει και τι να κάνουμε. Πολύ εκτιμώ τα όσα μας είπατε και θα σας δώσουμε και ε, ένα παράδειγμα. Είπατε τι κάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τι ζητάει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πραγματικά σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και τώρα ερχόμαστε στην τελευταία ομιλήτρια από το πάνελ. Θα είστε η φωνή της κοινωνίας των πολιτών. Χαίρομαι πάρα πολύ ε, που έχω την ευκαιρία να δώσω το λόγο στην κυρία Βιβιάν Τάιτελμπαουμ, πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Λόμπι Γυναικών. Έχετε κι εσείς ένα δεκάλεπτο, παρακαλώ. And, uh, Ευχαριστώ πολύ. Θα ξεκινήσω και εγώ ευχαριστώντας σας, ε, Πρόεδρε Μίκαελ, για αυτή την πρόσκληση είναι χαρά και τιμή για μένα που βρίσκομαι εδώ σήμερα για να γιορτάσουμε κατά κάποιο τρόπο την Διεθνή ημέρα της γυναίκας με την Επιτροπή των Δικαιωμάτων των Γυναικών και της Ισότητας των Φίλων που πρέπει να πούμε παίζει ένα κρίσιμο σημαντικό ρόλο προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι τα δικαιώματα των γυναικών και η ισότητα μεταξύ των γυναικών και των ανδρών θα παραμείνουν στην πολιτική ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε όλες τις πολιτικές της. Όπως πολλοί από σας γνωρίζουν, το Ευρωπαϊκό Λόμπι Γυναικών είναι η μεγαλύτερη συμμαχία μη κυβερνητικών οργανώσεων ε, δικαιωμάτων των γυναικών στην Ευρώπη, με μέλη σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς επίσης τη Σερβία, την Μακεδονία, Λεωμίλητρια και την Τουρκία. Είναι πολύ επίκαιρο και σημαντικό που βρίσκομαι εδώ σήμερα και μιλώ εκ μέρους όλων των γυναικών που αντιπροσωπεύουμε, προκειμένου να μοιραστώ μαζί σας ε, τις ανησυχίες ε, και τις προκλήσεις ε, που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες σε όλη την Ευρώπη σε ό,τι αφορά την ε, βία κατά των γυναικών. Σήμερα ακούσαμε πως η βία κατά των γυναικών εξακολουθεί να είναι ένα ε, φαινόμενο που υπάρχει σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα αποτελέσματα, τα αριθμητικά στοιχεία που μας έδωσε η Υπηρεσία Θεμελιών και ε, μας εκπλήσουν. Ε, δε, μάλλον δεν μας εκπλήσουν παρόλο που είναι πολύ εντυπωσιακά. Εμείς εδώ και χρόνια ε, έχουμε προειδοποιήσει για το εύρος του φαινομένου, την επιμονή του και τις ε, συνέπειες του. Η βία κατά των γυναικών είναι εμπόδιο στην ισότητα των δύο φύλων. Τα στοιχεία και τα γεγονότα που υπέβαλε ο Οργανισμός Θεμελιών Δικαιωμάτων αποδεικνύουν το πόσο σημαντικό είναι να δράσουμε γρήγορα. Ήδη από το 1999 το Ευρωπαϊκό Λόμπι Γυναικών είχε ε, ανακαλύψει ότι μία στις πέντε ε, γυναίκες ε, ήταν θύμα ενδοκινιακής βίας στην Ευρώπη. Βλέπουμε ότι σήμερα το, νούμερο αυτό δεν έχει αλλάξει. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη πράξει αρκετά προκειμένου να αντιμετωπίσει αυτό, το, αυτή τη σημαντική παραβίαση των ε, ανθρωπίνων δικαιωμάτων των γυναικών και ευχαριστούμε πολύ την κυρία Επίτροπο, την κυρία Ρέντινγκ για τα εργαλεία που ανέτσι την νομοθεσία προκειμένου ε, να προβλάβουμε την βία των γυναικών όπως για παράδειγμα την Ευρωπαϊκή Εντολή Προστασίας και την Οδηγία των Δικαιωμάτων των Θυμάτων. Η συμπερίληψη των, του, των δικαιωμάτων γυναικών σε αυτή την οπτική, ε, σε αυτά τα όργανα, σε αυτά τα εργαλεία ήταν σημαντικό ε, κλειδί για να εγγυηθούμε την προστασία και την βοήθεια των γυναικών που είναι θύματα. Το πρόγραμμα Δάφνη είναι επίσης πολύ σημαντικό προκειμένου να μελετήσουμε και να προλάβουμε την ε, βία των γυναικών και προκειμένου να θέσουμε σε εφαρμογή σχέδια και προγράμματα για να κάνουν πραγματική αλλαγή στη ζωή των γυναικών. Μαζί με τα μέλη μας συνεχίζουμε να εργαζόμαστε στην βελτίωση της συνειδητοποίησης σε ό,τι αφορά την βία των γυναικών. Πέρσι δημοσιεύσαμε το δεύτερο βαρόμετρο του παρατηρητήριου μας. Αυτή τη φορά αφορούσε τους βιασμούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο βιασμός ε, είναι ε, η μορφή της σεξουαλικής βίας που περισσότερο πιο οριζόντια τιμωρείται ε, και έχει κωδικοποιηθεί σε όλες τις εθνικές νομοθεσίες. Εξακολουθεί να είναι η μορφή της βίας που είναι πιο πολλά καλά κρυμμένη. Ε, αντιπροσωπεύει πράξεις που χρησιμοποιούν οι άντρες ε, ομαδικά και ατομικά για να εξασφαλίσουν ε, την, την ισχύ τους, να διατηρήσουν τον έλεγχο, που ασκούν ε, επί των γυναικών. Από, τις, από 32 χώρες με τις οποίες ήρθαμε σε επαφή, μόνο 5 έχουν ε, ε, προσαρμόσει την ομοθεσία τους στη, στους ορισμούς της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης. τα, στοιχεία που έχουμε είναι πολύ φτωχά, με ελάχιστες εξαιρέσεις, σχεδόν δεν έχουμε καθόλου στοιχεία για, τα θύματα, για, γυ, για γυναίκες θύματα. Εκτιμάται γενικά ότι το 90% των βιασμών δεν καταγγέλλονται και οι υπηρεσίες, ε, ε, οι κοινωνικές υπηρεσίες ε, λείπουν ή είναι τελείως ανύπαρκτες. Τα στοιχεία αυτά υποστηρίζουν την άποψη ότι η Ευρώπη μπορεί να κάνει κάτι παραπάνω. Την περασμένη εβδομάδα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέτησε δύο σημαντικέ εκθέσει για τη βία κατά των γυναικών. Μία για την βία κατά των γυναικών και μία για την πορνεία και την σεξουαλική εκμετάλλευση. Και οι δύο εκθέσει ζητούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση περισσότερη δράση. Ε, οι ευρωβουλευτές ε, έκαναν την ίδια αξιολόγηση της κατάστασης. Οι γυναίκες ε, προστατεύονται με τρόπο άνισο στην Ευρωπαϊκή Ένωση ακόμα. Εξαρτάται το που μένουν, που διαβιούν δηλαδή το, η, η πρόσβαση για παράδειγμα στην δικαιοσύνη και το αν θα τις ακούσει κάποιος εξαρτάται που ζουν. Ε, επίσης τα στερεότυπα έχουν παίζουν σημαντικό ρόλο και εμποδίζουν την αλλαγή της νοοτροπίας. Από τη μια μεριά η, ε, μέσα στο πλαίσιο της λιτότητας οι γυναίκες ε, επιστρέφουν στον παραδοσιακό τους ρόλο ως δεύτερο άτομο που κερδίζει χρήματα στο σπίτι. Κάτι που διονύζει τα στερεότυπα για τους ρόλους και τις ευθύνες του καθενός στην οικογένεια. Αυτό έχει συνέπεια στις επιλογές που κάνουν τα κορίτσια σε ό,τι αφορά την εκπαίδευσή τους και την καριέρα τους, καθώς επίσης έχει επίπτωση και στην οικονομική ανεξαρτησία των γυναικών. Από την άλλη πλευρά, το φαινόμενο της υπερβολικής σεξουαλικής δραστηριότητας αυξάνεται στην Ευρώπη, ε, οι σεξιστικές διαφημίσεις γίνονται καθημερινότητα ε, ενώ η δημόσια σφαίρα πορνοποιείται. Βλέπουμε όλο και περισσότερες εικόνες που δίνουν, στέλνουν το μήνυμα ότι το σώμα των γυναικών και η σεξουαλικότητά τους ε, είναι διαθέσιμα για τις φαντασιώσεις των ανδρών ε, και προωθείται περισσότερο η εμφάνιση και λιγότερο η αυτοπεποίθηση. Αυτό έχει άμεση επίπτωση στη σχέση μεταξύ ανδρών και γυναικών και ε, σε ό,τι αφορά την, ε, το ευάλωτο των γυναικών και των κοριτσιών ε, στην αντρική βία. Τα δύο ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καταγράφουν αυτή την κατάσταση και τη διαφορά των νομοθεσιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Την, του χρόνου η Ευρωπαϊκή Ένωση μαζί με όλες τις χώρες του πλανήτη θα γιορτάσουν 20 χρόνια από την πλατφόρμα του, δράσης του Πεκίνου ένα εργαλείο του, ένα, ένα έγγραφο του ΟΗΕ κλειδί για την πρόθεση των δικαιωμάτων των γυναικών και την υλοποίηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών. Η βία εναντίον των γυναικών είναι ε, μία από τις 12 περιοχές οι οποίες, τις οποίες προσδιορίζει η πλατφόρμα 20 χρόνια μετά την υιοθέτησή της. Πώς είναι δυνατόν να είναι τόσο επίκαιρη αυτή η πλατφόρμα δράσης του Πεκίνου οι παγκόσμιες, ε, ε, εμφανίζονται παγκόσμιες μετακινήσεις, ε, ζητούν τέλος τη βία εναντίον των γυναικών και ζητούν από αυτούς που να να δράσουν. Την περασμένη εβδομάδα πήραμε μέρος στην δεύτερη ε, στη δεύτερη εκστρατεία ε, συλλογής ενός δισεκατομμυρίου, μια παγκόσμια δράση για την βία κατά των γυναικών. Πολλοί ευρωβουλευτές μάλιστα συμμετείχαν και ε, μας βοήθησαν να ζητήσουμε το 2016 να είναι έτος Ευρωπαϊκής Ένωσης για το τέλος της βίας κατά των γυναικών. Πρέπει να προλάβουμε τη βία. Αυτό είναι ε, ευθύνη όλων των πολιτών. Όμως δεν μπορούμε να πετύχουμε σε αυτό αν οι κυβερνητικοί φορείς δεν δράσουν και ε, δεν σε δεν σταθούν στο ύψος των περιστάσεων σε ό,τι αφορά την υποχρέωσή τους ε, να νομοθετήσουν, ε, να εξασφαλίσουν πρόσβαση στη δικαιοσύνη για όλες τις γυναίκες, συμπεριλαμβανομένων των γυναικών με ιδιαίτερες ανάγκες όπως οι μετανάστριες, ε, τις ε, λεσβίες, ε, τις διασεξουαλικές, τις νέες, τις πιο ηλικιωμένε κλπ. Χρειαζόμαστε μέτρα και υπηρεσίες για να στηρίξουμε τις γυναίκες, να τις βοηθήσουμε να επιβιώσουν τις βίες και να φτιάξουν μια καινούρια ζωή. Και χρειαζόμαστε μια αλλαγή νοοτροπίας. Το Ευρωπαϊκό Λόμπι Γυναικών πιστεύει ότι οι δράσεις πρόληψης, ε, είτε είναι εκστρατείες ε, συνειδητοποίησης, ευαισθητοποίησης, ε, κατάρτισης προσωπικού, ενίσχυσης της δράσης των ίδιων των νέων γυναικών, δουλειά με τα παιδιά και με άντρες, δραστηριότητες στο σχολείο, συμπερίληψη των γυναικών, των γυναικών στην, στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα κλπ. μπορεί να είναι αποτελεσματικά μόνο αν ε, ενταχθούν σε ένα συνολικότερο πλαίσιο ε, κατά πολέμηση της βίας κατά των γυναικών. Η νομοθεσία δίνει ένα μήνυμα στην κοινωνία. Άντρε και γυναίκε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να περιμένει άλλα 20 χρόνια. Καλούμε τα κράτη-μέλη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εργαστούν μαζί με το νέο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να δώσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση μια ε, προοδευτική μεταρρυθμιστική στρατηγική για να δώσουμε τέλο σε όλε τι πράξει βία κατά των γυναικών. Αυτό είναι το μα ενώπιον των ευρωεκλογών. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, Βιβιάν. Νομίζω μπορούμε να πούμε ότι ο νόμος δεν αλλάζει τα πάντα, αλλά είναι ένα πολύ ισχυρό εργαλείο, ένα πολύ ισχυρό μήνυμα προς την κοινωνία, εάν θέλει κανείς να προκαλέσει αλλαγές. Αλλά πρέπει να γίνουν κάποια βασικά βήματα πριν μπορέσει να εγκριθεί κάποιος νόμος. Είναι πολύ σημαντικό για πολλούς από τους συναδέλφους στην Επιτροπή μας το Ευρωπαϊκό Λόμπι Γυναικών και πραγματικά εκτιμάμε ιδιαίτερα τη δουλειά σας και το έργο σας γενικότερα. Ευχαριστώ πολύ λοιπόν για όσα κάνετε. Τώρα να ξεκινήσουμε την συζήτηση. Να ακούσουμε πρώτα βουλευτές και ευρωβουλευτές. Σχόλια και παρατηρήσεις με τον κανόνα που αφαιρμόσαμε και πριν. Τρία λεπτά Εάν κάποιος ξεπεράσει το όρο, θα τον διακόψουμε. Πρώτη, πρώτες ομιλήτριες, η κυρία Ρεπούση από την Ελλάδα, η κυρία Καζάκα από την Λετωνία και μετά ο κύριος Φωκλής Φίτης από την Κύπρο. Η κυρία Ρεπούση από την Ελλάδα πρώτα. Έχετε το λόγο για τρία λεπτά. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω καταρχήν να εκφράσω τη χαρά μου που βρίσκομαι ανάμεσά σας και επίσης την αίσθησή μου ότι καμιά φορά η ελληλεγγύη ανάμεσα στις γυναίκες υπερβαίνει τα εθνικά σύνορα. Αισθάνομαι σήμερα πολύ πιο αλληλέγγυα μαζί σας από ότι ε, ίσως με το Εθνικό μου Κοινοβούλιο που κυριαρχείται όπως και άλλα εθνικά κοινοβούλια από άντρες. Η έρευνα του ΦΡΑ ήταν πάρα πολύ σημαντική. Ο πρώτος λόγος κατά τη γνώμη μου είναι ότι έδειξε με αριθμούς, κατέστησε ορατή τη βία κατά των γυναικών. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι κανείς δεν δικαιούται σήμερα να κάνει ότι δεν γνωρίζει το πόσο εκτεταμένη είναι η βία και το πόσο αφορά όλες τις χώρες. Κατέριψε επίσης κάποια στερεότυφα αναφορικά με τη βία κατά των γυναικών, για παράδειγμα το στερεότυπο του βορρά με τον νότο. Άρα πιστεύω ότι η δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων αυτών θα είναι πάρα πολύ σημαντική για να αναλάβει και η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης τις ευθύνες τους απέναντι σε αυτό το φαινόμενο. Δεν είναι δυνατόν να οδεύουμε στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και οι Ευρωπαίοι πολίτες γυναίκες να εξακολουθούν να είναι θύματα εκτεταμένης βίας, φυσικής, σεξουαλικής και ψυχολογικής στον ιδιωτικό και στο δημόσιο χώρο. Τι κάνουμε λοιπόν. Νομοθετικές ρυθμίσεις, οπωσδήποτε, οι νομοθετικές ρυθμίσεις είναι πάρα πολύ σημαντικές για να αντιμετωπίσουμε το φαινόμενο. Να επικυρώσουμε ε, τη σύμβαση της Ισταμπούλ, να θωρακίσουμε τον νομικό μας πολιτισμό, αλλά κατά την άποψή μου χωρίς συνολική αντιμετώπιση του φαινομένου δεν μπορούμε να το μειώσουμε, δεν μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Μην ξεχνάμε ότι η βία συνιστά την ακραία μορφή των σχέσεων κυριαρχίας ανάμεσα στα δύο φύλλα, των σχέσεων εκμετάλλευσης, θα έλεγα, ανάμεσα στα δύο φύλλα. Αυτή είναι η δομή της βίας κατά των γυναικών και αν δεν αντιμετωπίσουμε συνολικά τη δομή φοβάμαι ότι οι γυναίκες θα εξακολουθήσουμε να είμαστε θύματα της βίας. Στην Ελλάδα, για παράδειγμα, για να φέρω μερικά παραδείγματα, ψηφίσαμε το 2006 ένα πάρα πολύ σημαντικό νόμο γιατί αναγνώριζε το βιασμό ε, σε ενδοοικογενειακό πλαίσιο. Αυτό υπήρξε πολύ σημαντικό αλλά πολύ λίγες γυναίκες κατήγγυλαν το φαινόμενο και πολύ λιγότερες έφτασαν στα δικαστήρια γι' αυτό. Ε, θα βλέπω ότι ο χρόνος μου ε, έχει τελειώσει και δεν θέλω να πάρω περισσότερο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Thank you Σας ευχαριστώ πολύ. Ναι, βλέπετε το χρόνο, θέλετε να παρακολουθείτε το χρόνο. Σας παρακαλώ, λάβετε το υπόψη. Και τώρα το λόγο έχει η κυρία Κασάκα από τη Λετωνία. Παρακαλώ. Για τρία λεπτά κι εσείς. Ευχαριστώ. ημέρα σε όλους σας. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που μας προσκαλέσατε στη διάσκεψη αυτή και να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη διοργάνωση και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις προτάσεις της η βία κατά των γυναικών, η καταπολέμηση της βίας, της ενδοοικογενειακής, ε, των διακρίσεων, η προώθηση της ισότητας, όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά θέματα. Ε, και η ενδοοικογενειακή βία δεν αφορά μόνο τις γυναίκες αλλά και τα παιδιά. Ε, πραγματικά είναι πολύ χρήσιμα. Σας ευχαριστώ και για τη μελέτη του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων Δυστυχώς η Λετωνία είναι μία από τις χώρες που έχει ε, τα, ε, περισσότερα, ή από τα περισσότερα κρούσματα βίας κατά των γυναικών. Τα ποσοστά είναι της τάξης του 30 με 39%. Γι' αυτό θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους σας ε, και τις ΜΚΟ και τα Εθνικά Κοινοβούλια που συμμετείχαν σε αυτή την προσπάθεια για να εγκριθούν οι νόμοι κατά της ενδοοικογενειακής βίας. Τέλος, Βρισκόμαστε ε, πλέον σε μια φάση όπου ε, δεν θα πρέπει να απομονώνεται το θύμα σε περίπτωση ε, βίας, αλλά ο δράστης, ο θήτης, για να σπάει αυτός ο φαύλος κύκλος. Δυστυχώς οι στατιστικές στην περίπτωσή μας δεν ομιλούν υπέρ μας. Και βλέπουμε ότι η Λετωνία είναι μάλιστα και από τις χώρες δωρήτριες εντό εισαγωγικών χώρες προέλευσης του τράφικινγκ και είναι θύματα οι γυναίκες αυτές οι λετονές ε, είναι πολύ ψηλότερα τα ποσοστά από ορισμένες άλλες χώρες θα θέλαμε λοιπόν να βεβαιωθούμε ότι τα ε, σεξουαλικά και αναπαραγωγικά δικαιώματα των γυναικών γίνονται σεβαστά και στις επόμενες ευρωεκλογές αυτό το θέμα θα μας απασχολήσει και πάλι θα ήθελα να σας αναφέρω τα βήματα που θα πρέπει να κάνουμε για να μειωθεί η βία κατά των γυναικών. Πρώτα απ' όλα πιστεύω ότι θα πρέπει να ασχολούνται με την πολιτική περισσότερες γυναίκες για να επηρεάζουν τη λήψη των αποφάσεων σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και βεβαίως ευρωπαϊκό επίπεδο για να έχουμε ισότητα φίλων, εκρίζωση της φτώχειας και της βίας στη συνέχεια. Διότι όπως βλέπουμε και από τη μελέτη ε, σε χώρες που υπάρχει μεγάλη φτώχεια. Οι στατιστικές της βίας κατά των γυναικών δείχνουν ότι είναι υψηλότερη η βία αυτή και θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ε, τις απαραίτητες υπηρεσίες υποδοχής των γυναικών για να μπορούν να ξαναμπαίνουν στην αγορά εργασίας και να γίνονται πιο ανεξάρτητες και οικονομικά. Μια άλλη ε, πρόταση για εκείνους που παίρνουν τις αποφάσεις και τους πολιτικούς είναι η συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και τώρα το λόγο έχει ο κύριος Σοφοκλής Φίτης, παρακαλώ, από την Κύπρο. Ε, κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι, το θέμα που πραγματεύεται η σημερινή συνάντηση είναι δυστυχώς πάντα επίκαιρο, αφού ταλανίζει τις κοινωνίες μας διαχρονικά. Η έμφυλη βία εμποδίζει τις γυναίκες να συμμετέχουν ισότιμα στην κοινωνία και να απολαμβάνουν πλήρως τα ανθρώπινα τους δικαιώματα. Το Συμβούλιο της Ευρώπης έχει εκπονήσει έρευνα για το οικονομικό αντίκτυπο της βίας κατά των γυναικών και των εμποδίων που παρεμβάλλονται στην ενεργό συμμετοχή τους στην κοινωνία. Την έχουμε αναλύσει σήμερα. Σύμφωνα με τους σχετικούς υπολογισμούς, το, κόστο, το κόστος αυτό στην Ευρωπαϊκή Ένωση ανέρχεται στα 16 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Θα ήθελα να σας ενημερώσω για την πρόοδο που επιτελείται στον τομέα της πρόληψης της βίας κατά των γυναικών στη χώρα μου. Η Κυπριακή κυβέρνηση, παρά την οικονομική κρίση, έχει θέσει ψηλά στις προτεραιότητες της και έχει εκφράσει δημόσια την πολιτική της βούληση και δέσμευση για την περαιτέρω καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών. Καθώς η Κύπρος βρίσκεται σε πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής η κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε εμπεριστατωμένη μελέτη κατάθρων εξέτασης των υποχρεώσεων που προκύπτουν από τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης και κοστολόγηση αυτών των υποχρεώσεων. Στο μεταξύ όμως, το αρμόδιο Υπουργείο υλοποιεί ήδη μέτρα και πολιτικές που εμπίπτουν στο πεδίο δράσης του με σκοπό την εναρμόνιση της Κυπριακής Δημοκρατίας με τις πρόνοιες της Σύμβασης. Σε συνεργασία με την νομική υπηρεσία, Προωθεί επίσης την ψήφιση σειράς νομοθετικών μέτρων που περιλαμβάνονται στη Σύμβαση για ποινικοποίηση όλων των μορφών βίας κατά των γυναικών και αύξηση των προβλεπόμενων ποινών. Επίσης προετοιμάζεται η τροποποίηση του ποινικού κώδικα ώστε να επεκταθεί η δικαιοδοσία των Κυπριακών δικαστηρίων για εκδίκαση των αδικημάτων βίας Αυτά προβλέπονται επίσης στη Σύμβαση και ασφαλώς αν διαπράχθησαν έναντι οποιοδήποτε προσώπου με συνήθη διαμονή στην Κυπριακή Δημοκρατία. Και αυτό ανεξάρτητα από το αν διαπράχθηκαν εκτός της Κυπριακής Δημοκρατίας και αν αποτελούν αδίκημα στη χώρα που διαπράχθησε. Παράλληλα, προωθείται αναβάθμιση του ρόλου της αστυνομίας ώστε να καταστεί αποτελεσματικότερη στην πρόληψη και στην άμεση ανταπόκρισή της σε περιστατικά βίας. Ενώ μέσω του Εθνικού Μηχανισμού για τα Δικαιώματα της Γυναίκας ενισχύονται οργανώσεις και φορείς στην υλοποίηση προγραμμάτων και εκστρατιών ευαισθητοποίησης του κοινού και ενθάρρυνσης των θυμάτων να προσφεύγουν στις αρμόδιες υπηρεσίες για βοήθεια καθώς και στη δικαιοσύνη. Thank you σας ευχαριστώ πολύ. Επόμενοι τρεις ομιλητές τώρα. Η κυρία Κουλιάνο από την Ιταλία, η κυρία Ρώσα Μαρτίνες από την Ισπανία και η κυρία Έλσα Παΐς από την Πορτογαλία. Η κυρία Κούλιανο. Thank Ευχαριστώ. Θα προσθέσω και εγώ τις δικές μου ευχαριστίες σε αυτές των συναδέλφων προς το Ευρωκοινοβούλιο, το Συμβούλιο της Ευρώπης και όλες τους οργανισμούς που διοργάνωσαν αυτή την εκδήλωση προκειμένου να μελετήσουμε και να συζητήσουμε το φαινόμενο αυτό. Τους ευχαριστώ για την ποιότητα των δεδομένων που μας παρουσίασαν που είναι μια απαραίτητη βάση για οποιοδήποτε είδους έργο σε εθνικό ή ευρωπαϊκό επίπεδο. και προσωπικές είναι αυτές ευχαριστίες, αλλά και εξ ονόματος της Ιταλικής Βουλής και του Προέδρου της Ιταλικής Βουλής, της κυρίας Μπολτίνη, που είναι πραγματικά γνωστή για την πείρα της στον χώρο της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Έχει διδραματίσει ένα σημαντικότατο ρόλο σε όλη τη βουλευτική θητεία για τα θέματα που τόνισε και η συνάδελφος γερουσιαστής, η κυρία Ντορίζ Λομόρο η κύρωση της σύμβασης της ε, Κωνσταντινούπολης και οι κανόνες για την καταπολέμηση και την πρόληψη της κακοποίησης και της βίας είναι σοβαρά γεγονότα. Από την πολιτιστική σκοπιά της αλλαγής της νοοτροπίας και δεδομένης της Ιταλικής πραγματικότητας είναι σημαντικό ότι προβλέφθηκε ως αδίκημα πλέον, ως εγματική ενέργεια η η βία. Επιτέλους έχει πάρει και κοινωνικές διαστάσεις η βία κατά των γυναικών, η οποία είναι μια, δεν είναι νόσος, είναι μια μάστιγα που επιτείνει τις κοινωνικές διαφορές. Για όσους πήραν το λόγο να πω ότι εφόσον σχεδιάζουμε ευρωπαϊκή δράση δεν θα πρέπει να επικεντρωθούμε στο να συντονίσουμε απλώς τα διάφορα το παδράσεις, αλλά να παρέμβουμε κυρίως ε, στο επίπεδο της εκπαιδείας, της στήριξης και της πρόληψης. Πρέπει να υπάρχει ένα ενιαίο πλαίσιο σε ό,τι αφορά τις εθνικές πολιτικές αλλά και τις ευρωπαϊκές. Διότι κατά την άποψη μου η συστηματική προσέγγιση είναι το πλέον σημαντικό ζήτημα, διότι πολλές φορές οι αποκρίσεις μας είναι μια αντίδραση στα όσα συμβαίνουν και αυτό δεν αρκεί. Και μια τελευταία παρατήρηση, η βία και η κακοποίηση δεν είναι ένα θέμα μόνο δικαιωμάτων, είναι πολύ βαθύτερο όπως σωστά μας ε, δείχνουν ε, τα δεδομένα που ακούσαμε από το πρωί η αξιοπρέπεια, ο σεβασμός που πρέπει να διέπουν τις σχέσεις, τις διαπροσωπικές, δεν είναι θέμα μόνο πολιτιστικό ή νοοτροπίας ή νομοθεσίας. Είναι κυρίως θέμα νοοτροπίας. Εάν δεν δράσουμε διατομεακά, όπως πολλές συνάδελφοι τόνισαν, δεν θα έχουμε αποτελέσματα, γιατί χρειάζεται κοινή δράση. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ και η κυρία Ρος Μαρτίνος, τώρα από την Ισπανία. Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πολύ για τη διοργάνωση αυτής ε, της ημερίδας. Είναι πάρα πολύ σημαντική σε ένα τόσο σημαντικό θέμα όπως είναι η βία κατά των γυναικών. Αυτή είναι η πιο ομή έκφαση και έκφραση των ανισοτήτων. Χρόνο με το χρόνο ε, πέφτουν θύματα υπερβολικά πολλές γυναίκες, απλούστατα για το λόγο ότι είναι γυναίκες και μόνο. Αλλά όχι μόνο γυναίκες και τα παιδιά τους, ε, ανήλικα παιδιά, αγόρια και κορίτσια. Η κρίση όλους μας πλήττει, αλλά εκείνοι που είναι πιο ευάλωτοι πλήττονται περισσότερο ακόμα οι γυναίκες που βρίσκονται σε κατάσταση τέτοια κακοποίησης πιο δύσκολα ε, φεύγουν από ε, αυτή την κλιμάκωση. Ε, χρειάζονται μια ελάχιστη βοήθεια και μια εξασφάλιση ότι θα ξαναβρούν τη ζωή τους και η κρίση δεν είναι ένα τείχος ανυπέρβλητο. Εκεί θα πρέπει να βρεθούν οι κυβερνήσεις αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση πολύ περισσότερο από ποτέ και σήμερα που γνωρίζουμε και τα στοιχεία από τη μελέτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι πάρα πολύ σημαντικό να εργαστούμε σε εκστρατείες πρόσληψης, ενημέρωσης και ουσιαστικής προστασίας αλλά και συνειδητοποίησης, προστασίας και των θυμάτων και των παιδιών τους για να μην κλαίμε κάθε χρόνο θύματα από αυτές τις επιθέσεις. Και σύντομα θα ήθελα να αναφερθώ στη σημασία που έχει εδώ η παιδεία. Το εκπαιδευτικό σύστημα είναι το ιδεώδες πλαίσιο για να καταπολεμήσουμε αυτή την κοινωνική μάστιγα που είναι η βία κατά των γυναικών. Είναι το πιο σημαντικό εργαλείο και το πιο δυνατό για να ενημερώνονται οι νέοι και να μην αναπαράγονται στερεότυπα βίας. Δεν θα πρέπει να το παραγνωρίζουμε. Η κοινωνία πρέπει να δράσει, Αλλιώ θα έχουμε αιωνίω θύματα διαφόρων μορφών βία καθ' όλη τη διάρκεια τη ζωή του. Θυμάμαι μία πρόταση που λέει ότι ο σεβασμός είναι κάτι το σημαντικό και θα πρέπει να στο διδάσκουν όταν είσαι μικρός. Ε, ακριβώς. Ε, ε, τα ε, θύματα ε, και οι θύτες μάλλον έχουν υπάρξει θύματα σε μικρή ηλικία και το αναπαράγουν στη συνέχεια. Η βία κατά των γυναικών θα πρέπει να καταπολεμείται από τις αίθουσες των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και από τα εκπαιδευτικά κέντρα γιατί όταν κάτι δεν ε, αποτελεί αντικείμενο συζήτησης δεν υπάρχει. Μια κοινωνία που δεν εκπαιδεύει σε όρους σεβασμού, ανοχής και ισότητας δεν πιστεύει ούτε στη δημοκρατία ούτε στην ελευθερία. Η καλύτερη παιδεία και εκπαίδευση είναι αυτή που γίνεται με όρους ισότητας. Και τελειώνω λέγοντας ότι κάθε γυναίκα ε, που σώζεται είναι ε, μια κοινή επιτυχία όλης της κοινωνίας των πολιτών και τελικά και της ίδιας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ πολύ και εγώ σας ευχαριστώ και τώρα το λόγο έχει η κυρία ε, Παΐς από την Πορτογαλία. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, να ξεκινήσω λέγοντα ότι τα δικαιώματα των γυναικών είναι ανθρώπινα δικαιώματα. Γι' αυτό πρέπει να έχουμε ενεργό ρόλο σε αυτόν τον αγώνα. Δεν είναι αγώνα των γυναικών, δεν είναι αγώνα μόνο δικός τους, αλλά είναι και των ανδρών. Είναι ένας αγώνας για τους ανθρώπους, και γι' αυτό έχει και πολιτικέ διαστάσει. Τα δεδομένα του οργανισμού για τα θεμελιώδη δικαιώματα δείχνουν ότι μία στι τρει γυναίκε είναι θύμα μια μορφή βία. Μιλάμε για μια πράξη βαρβαρότητα στην Ευρώπη των δικαιωμάτων. Και δεν μιλάμε για θανάτου, διότι όταν μιλήσουμε για θανάτου, πραγματικά τρομάζουμε στην Πορτογαλία, τη χώρα μου, κατά μέσο όρο χάνουν τη ζωή του 40 γυναίκε ετησίω. θύματα τη ενδοικογενειακής βία, πέραν των άλλων μορφών τη βία. Η βία λοιπόν και η παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των γυναικών ζημιώνει τους πάντες, όχι μόνο τις γυναίκες. Βλάπτει την ανάπτυξη, βλάπτει την ανταγωνιστικότητα, βλάπτει την ανταγωνιστικότητα των γυναικών. Άρα είναι επιζήμια για την ανάπτυξη ολόκληρη της κοινωνίας. Γι' αυτό δεν πρέπει να ε, ξεχνάμε ότι το θέμα αυτό είναι καθοριστική σημασία ακόμη και στην περίοδο της κρίσης. Μάλλον καλύτερα κατεξοχήν επειδή υπάρχει κρίση πρέπει να λάβει τις διαστάσεις προτεραιότητας που τις αρμόζουν η ε, ε πολιτική αυτή. Θα πρέπει λοιπόν να προωθήσουμε, να επιδιώξουμε μια κοινωνία δίκαιη, όπου θα ε, καλλιεργείται η ισότητα, όπου θα καταπολεμούνται όλες οι μορφές διάκρισης διακριτικής μεταχείρισης διάκριση κατά της μισής ανθρωπότητας βάσει του φύλου. Γι' αυτό μιλάμε. Από κοινωνική σκοπιά λοιπόν δεν μπορούμε να το ξεχνάμε. Υπάρχουν τόσες μορφές διακριτικής μεταχείρισης κατά των γυναικών. Πάντοτε ε, πέφτουν θύματα διακριτικής μεταχείρισης. Εάν μιλάμε για την έμφυλη αυτό είναι ένα κομμάτι. Αλλά υπάρχουν και τόσες άλλες μορφές διακρίσεων. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να περάσουμε από τους νόμους στις πράξεις. Η ισότητα και η μη διάκριση είτε αντιμετωπίζεται ως ένα πραγματικό φαινόμενο με συγκεκριμένες εκφάνσεις είτε δεν αντιμετωπίζεται καθόλου. Η σύμβαση της Κωνσταντινούπολης μας θέτει ορισμένους στόχους. Δεν μπορούμε λοιπόν απλώς να συζητούμε θεωρητικά, πρέπει να δράσουμε. Πρέπει να προβλεφθεί μια οδηγία ώστε να υποχρεωθούν όλα τα γιατί μέλη να, πάρουν ρόλο να λάβουν ρόλο σε αυτόν τον αγώνα. Και θα πρέπει να γίνουμε μαχητικοί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτή η στρατηγική δεν μπορεί να είναι βραχυπρόθεσμη. Είναι μια στρατηγική και βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη. Και το λέω και το ξαναλέω. Την αγώνα αυτό μπορούμε να τον κερδίσουμε. Είναι μία πρώτη μάχη και είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να προβλεφθεί και στο εκπαιδευτικό σύστημα. Με ε, συγκεκριμένη πρόβλεψη για την ιδιότητα του πολίτη και για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Εάν δεν ξεκινήσει τώρα αυτή η μάχη, δεν θα κερδίσουμε ποτέ. Κανείς δεν μπορεί να κερδίσει εάν δεν γίνει προτεραιότητα για όλους και για την οικονομία και ω οικονομική προτεραιότητα είναι σημαντικό και θα ήταν ενδιαφέρον να οργανώσουμε μια προσοχή διάσκεψη ακριβώ με αυτή την προβληματική στο κέντρο τη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο λόγο στην Τέπορα. Ευχαριστώ ο στην Σάμπρη από τη Μάλτα. Και μετά στην κυρία Μέρφυ πριν δώσω το λόγο στους ομιλητές του πάνελ. Από όταν ήμασταν παιδιά, μας έλεγαν ότι συνήθως τιμωρούμαστε όταν κάνουμε κάτι κακό, μια ταξία. Επίσης, μας μάθαιναν ότι οι γυναίκες θα πρέπει να κρατούν ενωμένη την οικογένειά τους. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα από τα πιο σημαντικά προβλήματα, τα σχετιζόμενα με την ενδοοικογενειακή βία. Πρέπει να μάθουμε στις γυναίκες να πάψουν να νιώθουν ένοχες πρέπει να σταματήσουμε να τις κάνουμε να πιστεύουν ότι άξιζαν ή αξίζουν αυτή τη βία. Εγώ είμαι οικογενειακή δικηγόρο και ένα από τα βασικά προβλήματα που βλέπουμε τι πελάτησέ μου είναι αυτό ακριβώ. Οι γυναίκε πιστεύουν ότι αξίζουν αυτό που παίρνουν. Αξίζουν την κακομεταχείριση. Δεν είναι καλό αυτό. Δεν είναι καλό ω νοοτροπία. Δεν είναι καλό να πιστεύει η γυναίκα ότι δεν μπορεί να βγει από αυτό το αδιέξοδο διότι θα διαρρήξει την οικογένειά της με αυτόν τον τρόπο. Όχι, πρέπει να ε, διδάξουμε τις γυναίκες ότι είναι καλό να κρατάνε δεμένη την οικογένεια αν αυτή η οικογένεια είναι ειρηνική, αν είναι η οικογένεια που διέπεται από αγάπη. Αλλά οι οικογένειες οι οποίες είναι δυσλειτουργικές είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Μερικές φορές εξαιτία και χάρη στα παιδιά μας, για χάρη των παιδιών μας θα πρέπει να φεύγουμε από την οικογένεια. Και αν διδάξουμε αυτό το πράγμα στις γυναίκες μας, και δεν μπορούμε να μιλάμε για συμβάσεις με ανθρώπους που δύσκολα γράφουν ή διαβάζουν. Πρέπει να τους μιλάμε με τη γλώσσα που καταλαβαίνουν. Πρέπει να μάθουμε στις γυναίκες, να διδάξουμε στις γυναίκες ότι ε, ποτέ δεν αξίζουν την κακομεταχείριση πρέπει να διατηρούν ενωμένε τις, γυναί- τις οικογένειές τους όταν είναι καλές, αλλά όταν είναι δυσλειτουργικές πρέπει να τις εγκαταλείπουν και θα πρέπει να αναζητούν βοήθεια και στήριξη. Και οι συμβάσεις θα πρέπει να είναι ευανάγνωστες. Τα νομοθετικά κείμενα θα πρέπει να συντάσσονται με γλώσσα την οποία να καταλαβαίνουν οι γυναίκες. Χρειάζονται περισσότερες εκστρατείες ε, προώθησης αυτών των συμβάσεων και περισσότερη προβολή των προτεραιοτήτων μας, των, ε, συγγνώμη, των πρωτοβουλειών μας. Είναι πολύ σημαντικό αυτό να γίνει και σε εθνικό επίπεδο, στα εθνικά κοινοβούλια και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Χρειάζεται να είμαστε όμως ευαίσθητοι έναντι των αναγκών των γυναικών ε, που, που έχουμε, βλέπουμε καθημερινά. Ευχαριστώ. Τελευταία ομιλήτρια από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Ισότητας των Φύλων, η κυρία Μέρφη. Έχετε το λόγο. Ε, δεν, έχω πάντοτε, δεν έχω πολύ συχνά τον τελευταίο λόγο, θα το χαρώ σήμερα. Ε, θέλω να σχολιάσω αυτά που είπε η Ισπανίδα ε, ομιλήτρια στο προηγούμενο πάνελ. Μίλησε για την σημασία της εμπειρίας της Ισπανίας σε ό,τι αφορά τις εκστρατείες ευαισθητοποίησης και επιμόρφωσης ε, των επαγγελματιών. Αυτό επιβεβαιώνεται και στη δική μας μελέτη. Είναι πολύ σημαντική πτυχή της καταπολέμησης και της πρόληψης, ιδιαίτερα της ενδοοικογενειακής βίας. Να σας ε, δώσω και κάποια καλά νέα ενδεχομένως. Ε, θα ήθελα να διατρέξω το έργο του Ινστιτούτου μας. Είναι μια μακροσκελής λίστα, ένα μακροσκελής κατάλογος. Ένα από τα πράγματα τα οποία κάνουμε είναι εξετάζουμε τα στοιχεία προέρχονται από διοικητικέ πηγές από τα 28 κράτη-μέλη. Τα πρώτα μας πορίσματα θα τα υποβάλουμε στις 20 Μαρτίου. Δημιουργούμε και μια βάση δεδομένων σεξουαλικής βίας που θα είναι διαθέσιμη στο μισθό τοπό μας. Κάνουμε μια μελέτη για το κόστος της βίας. Ε, έχουμε ήδη καταγράψει καλές πρακτικές βέλτιστες πρακτικές για την πρόληψη και αυτές είναι στο, νηστό τοπό μας. Έχουμε μία μελέτη το 2012 ε, για τον ακροτηριασμό γεννητικών οργάνων, θα συνεχίσουμε και φέτος. Ε, ε, εξετάζουμε το, σε ποια κατάσταση βρίσκεται η εφαρμογή της πλατφόρμας του δράση του Πεκίνου. Κάναμε το 2012 μια μελέτη για την υποστήριξη των θυμάτων με πολύ εντυπωσιακά αποτελέσματα. Ελπίζω να την έχετε διαβάσει. Είναι πολύ καλή πηγή για βέλτιστες πρακτικές. Επίση, αναμένουμε να εργαστούμε με τα στοιχεία της μελέτης ε, που προέκυψε και παρουσιάστηκε σήμερα και να τα συγκρίνουμε τα δικά μας στοιχεία. Η συλλογή δεδομένων είναι πάρα πολύ σημαντική. Και η Κομισιόν θα πρέπει να υποστηρίξει τα κράτη μέλη σε ό,τι αφορά ε, τη συλλογή δεδομένων ε, τη, σχετικών με τα θύματα βίας. Είναι πολύ σημαντικό να ενοποιηθούν μεθοδολογίες στη συλλογή των δεδομένων. Αυτά είναι τα, αυτές είναι οι περιοχές στις οποίες εργαζόμαστε και ήθελα να σας το αναφέρω γιατί όλα αυτά είναι κομμάτια του ίδιου παζλ ενός στρατηγικού πλαισίου σε ευρωπαϊκό επίπεδο ενός ε, σχεδίου για τα βήματα που θα πρέπει να κάνουμε τα επόμενα 45 χρόνια σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ε, συγγνώμη, τα επόμενα 4-5 χρόνια ε, ε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να καταπολεμήσουμε το φαινόμενο της ε, βίας κατά των γυναικών. Thank Σας ευχαριστώ πολύ. Κυρία Μέρφη, από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Ισότητας των Φίλων. Τώρα θα έχουν την ευκαιρία οι κυρίες του πάνελ σύντομα να απαντήσουν. Δυστυχώς δύο πρέπει να αποχωρήσουν. Το ξέραμε από την αρχή αυτό. Με ποια σειρά θέλετε, κύριε Γόλμπη. Δεν είστε υποχρεωμένοι, αν θέλετε να πείτε κάτι. Πολύ γρήγορα, νομίζω. Είναι υπέροχο που η κάθε ομιλήτρια θέλει και θέλησε να μιλήσει με καμάρι για την καλή δουλειά που γίνεται στη χώρα της. Δεν είναι υπέροχο αυτό. Όλοι θέλησαν να πούν κάτι για την πρόοδο που έχει επιτελέσει η χώρα τους. Ε, τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης μίλησαν για τη δική τους τη δουλειά. Όλα αυτά όμως, τα κομμάτια δουλειάς, πρέπει κάποια στιγμή να συνδυαστούν και να υπάρξει στρατηγικό συντονισμός, ώστε να μπορέσουμε στην πράξη να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα που απασχολεί όλες μας. Δεν άκουσα να υπάρχει τέτοια συνένεση και συμφωνία και ομοψυχία σε ομάδα πολιτικών. Είναι νομίζω υπέροχο αυτό. Ευχαριστώ. Να προσθέσω ίσως απλώς ότι βεβαίως οι γυναίκες δεν είναι απλώς μόνο θύματα αλλά είναι και μια θαυμάσια δύναμη, πηγή ενέργειας και νομίζω ότι πρέπει και αυτό να το έχουμε κατά νου. Σε αυτό το επίπεδο επίσης πρέπει να εργαστούμε, διότι η βία δεν μπορεί να είναι ένα πρόβλημα μόνον των γυναικών. Πρέπει να γίνει πρόβλημα της κοινωνίας. Γι' αυτό μας ενδιαφέρει κάποια εργαλεία να τα ενεργοποιήσουμε πραγματικά, να τα χρησιμοποιούμε οι γυναίκες πρέπει να έχουν στα χέρια τους τα μέσα, τα εργαλεία για να μπορούν να ασκήσουν και την ε, δική τους την εξουσία, τη δύναμη όταν χρειάζεται. Αλλά να μην ξεχνάμε την ενέργεια που έχουν όλες οι γυναίκες, τα δίκτυα των γυναικών και πώς συνεργάζονται. Πάντως, αυτό που θέλω να πω εδώ μπροστά σας και νομίζω όλοι συμφωνείτε, είναι ότι χρειαζόμαστε περισσότερη εκπαίδευση, παιδεία, νομοθεσία και σεβασμό. Από εκεί ξεκινούν όλα από τις ε, πρώιμες ηλικίε. Περισσότερα δεδομένα επίσης, έχουμε πολλά εργαλεία και είμαστε ευγνώμονες γι' αυτό, αλλά νομίζω μόνον όλα αυτά συνδυασμένα μπορεί να οδηγήσουν σε αλλαγή. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ, δεν θα μπορούσα να τα είχα πει καλύτερα. Και τώρα ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τα μέλη του πάνελ που ε, ήρθατε και μιλήσατε. Για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Τώρα θα υπάρξουν κάποιες ανακατατάξεις, δυστυχώς θα αποχωρήσετε ορισμένες. Παρακαλώ την κυρία Κόλια και την κυρία Παρβάνοβα να έρθουν στο Προεδρείο για να ε, αρχίσουμε σε λίγο, σε πολύ λίγο την τελευταία ενότητα. Uh, Μπορούμε να συνεχίσουμε. Έχουμε ακόμη δύο παρεμβάσεις. Πρωτού ολοκληρωθεί η διάσκεψή μας αυτή. Μετά τη λήξη της, να σας πω ότι έχουμε εδώ μια μικρή δεξίωση, έξω από την αίθουσα ακριβώς. Αλλά πριν από αυτό, μείνετε, να μείνετε μέσα παρακαλώ. Πρώτα θα ακούσουμε την παρέμβαση της κυρίας Κόλια, Γενικού, Γενικής Γραμματέως, για την ισότητα των φίλων του Υπουργείου Ευτερικών και εκ μέρους της Ελληνικής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχετε το λόγο. Για 10 λεπτά κι εσείς. Thank you, Mr. President. Κυρίε και κύριοι, το... σήμερα το πρωί ήδη θα το έχετε ακούσει και θα έχουν αναφερθεί οι προηγούμενοι ομιλητέ αρκετέ φορέ αυτό. Παρουσιάστηκαν σε ειδική εκδήλωση υπό την αιγίδα τη Ελληνική Προεδρία τα αποτελέσματα μια πανευρωπαϊκή έρευνα που έκανε ο ΦΡΑ, που διεξήγαγε ο ΦΡΑ. Είναι μία από τι μεγαλύτερε έρευνε που έχει διεξαχθεί παγκοσμίω για τη βία κατά των γυναικών. Σήμερα με την έρευνα αυτή έχουμε μια ακτινογραφία στα χέρια μας του φαινομένου, μια ακτινογραφία του φαινομένου, που για πρώτη φορά μας δείχνει μια ανατριχιαστική καθαρότητα, θα νομούσα να πω, τι συμβαίνει μεταξύ γυναικών και ανδρών. Τα στοιχεία μας ξαφνιάζουν. Το πρωί όσοι τα ακούσαμε πάθαμε σοκ. Αποκαλύπτεται μια απροσδόκητη ποσοτικά και ποιοτικά έκταση βίας κατά των γυναικών στο σπίτι, στη δουλειά, σε δημόσιους χώρους, στο διαδίκτυο μιας βίας που δεν γνωρίζει γεωγραφικούς, κοινωνικούς, οικονομικούς, πολιτισμικούς ή ηλικιακού περιορισμούς, που δεν σταματά στον ιδιωτικό χώρο, αλλά βρίσκει τα θύματά της μπροστά σε χιλιάδες ή και εκατομμύρια μάτια στον πραγματικό αλλά και στον ψηφιακό κόσμο και χώρο. Τα πρόσωπα, κυρίες και κύριοι, τη έμφυλης βία είναι πολλά και ποικίλα. Από βία μεταξύ συντρόφων, σεξουαλική βία. Νομίζω ότι τα ακούτε πρώτη φορά, αλλά καλό είναι να τα επαναλαμβάνουμε, να τα θυμόμαστε. Διακίνηση ανθρώπων, σύγχρονες μορφές δουλείας, αναγκαστικούς γάμους, ακροτηριασμό ε, γυναικείων αναπαραγωγικών οργάνων, εγκλήματα τιμής όπως τα αποκαλούνται, αλλά και νέες μορφές βίας, όπως η βία μέσω του διαδικτύου, η ηλεκτρονική παρενόχληση, η επίμονη παρακολούθηση και ο εκφοβισμός. Κυρίε και κύριοι, όπω ίσω να έχετε ακούσει, συγχωρέστε με αν επαναλαμβάνομαι γιατί καθυστέρησα να έρθω, η μία στι τρει γυναίκε τη Ευρώπη έχει πέσει θύμα σωματική ή και σεξουαλική βία από την ηλικία των 15 ετών και άνω. Πρόκειται ουσιαστικά για 60, 62 εκατομμύρια γυναίκες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ταυτόχρονα όμως διαπιστώνουμε από την έρευνα που διεξήγαγε ο ΦΡΑ ότι η Ευρωπαία φαίνεται να αρνείται να καταγγείλει το περιστατικό βίας στην αστυνομία ή σε άλλη οργάνωση και, να, και προστατεύει έτσι ή θελημένα πολλές φορές θέλει να προστατεύσει τον θήτη. Επιδεικνύει μειωμένη εμπιστοσύνη απέναντι στους μηχανισμούς άσκησης δίωξης εναντίον του θήτη. Ίσως πάλι να φταίει ο φόβος, ίσως η πίεση του περίγυρου, ίσως οι επιταγές ενός ακραίου πολυπολιτιστικού πλαισίου. Διερωτώ με ποια θα ήταν τα ποσοστά εάν οι γυναίκες μιλούσαν ελεύθερα για τις εμπειρίες τους στο θέμα της έμφυλης βίας. Για σκεφτείτε το λίγο. Το φαινόμενο από ό,τι αποκάλυψε η έρευνα είναι πολύ πιο πολύπλοκο από όσο πιστεύαμε μέχρι σύμφωνα. Και δυστυχώς βρίσκεται απλωμένο σε όλη την Ευρώπη, σε όλο τον ευρωπαϊκό χάρτη. Ένα γενικό έβριμα Επίση ανησυχητικό από την έκθεση, από την έρευνα του ΦΡΑΜ, είναι ότι ο πολίτη δεν, δεν φαίνεται να έχει αντίληψη της έκτασης του φαινομένου στην δική του χώρα. Οι αποκλίσεις μεταξύ της πρόσληψης του μεγέθους του προβλήματος και της πραγματικότητας είναι σημαντικές. Άραγε ο Ευρωπαίος πολίτης αρνείται να δεχτεί αυτή την εικόνα της πραγματικότητας. Μήπως γιατί η βία κατά των γυναικών είναι συχνά θέμα ταμπού. Μήπως άραγε ο πολίτης δεν γνωρίζει επαρκώς τελικά τι σημαίνει εμφυλβία. Είμαι βέβαιη κυρίε και κύριοι ότι κάποιες μορφές της έμφυλης βίας είναι βαθιά ριζωμένες στην καθημερινότητα, στην καθημερινότητα της Ευρώπης, στην καθημερινότητα του Ευρωπαίου πολίτη, φθάνοντας να θεωρούνται και φυσικές. Με την ολοκλήρωση τη έρευνα του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων τη Ευρωπαϊκή Ένωση του ΦΡΑ, ανοίγουν μεγάλα ζητήματα τα οποία χρήζουν εκτεταμένη διαβούλευση και προβληματισμού. Γιατί άραγε η βία κατά των γυναικών επιμένει σε τέτοιο βαθμό και έκταση σε μια ενωμένη Ευρώπη που για πολλέ περιοχέ τη Ιφιλίου θεωρείται η γη της επαγγελίας, κάτι που τόνισα και το πρωί. Πώς θα περάσουμε από το επίπεδο των θεσμών τελικά στο επίπεδο της δράσης, στο επίπεδο του πολίτη. Όλοι όσοι έχουμε την πολιτική ευθύνη, κυρίε και κύριοι, για τις προσπάθειες αντιμετώπισης αυτού του επιδεινούμενου κοινωνικού προβλήματος, πρέπει να επανεξετάσουμε την επάρκεια των σημερινών πολιτικών πρέπει να μας προβληματίσει το γεγονός ότι παρά τη κατά το χείρο των δικαιωμάτων των γυναικών, οι κοινωνίες μας αρνούνται έναν de facto σεβασμό και ιδιαίτερα στο θέμα της βίας κατά των γυναικών, ακόμη και των κοριτσιών. Δεν μπορούμε πλέον να κρύβουμε από τους εαυτούς μας το γεγονός ότι οι κοινωνίες μας, αναμφισβήτητα στην καρδιά του επιτυχμένου κόσμου, επιτρέπουν, αν όχι αρκετές φορές υποθάλπουν την έμφυλη βία. Τα συστατικά της έμφυλης βίας Κυρίε και κύριοι, φαίνεται να βρίσκονται ευρέω διαθέσιμα γύρω μα. Η άνηση κοινωνική ιεραρχία των φύλων εμποτίζει τον καθημερινό μα πολιτισμό. Οι σύγχρονε κοινωνικέ παθογένειε, ο απάνθρωπο ανταγωνισμό και οι αντικοινωνικέ συμπεριφορέ προκαλούν την ανάφλεξη τη έμφυλη βία. Σε κάθε περίπτωση, όπω καταλαβαίνετε, το θέμα της βίας κατά των γυναικών, η εξάλληψη της βίας κατά των γυναικών δεν θα μπορούσε παρά να αποτελεί προτεραιότητα της ελληνική προεδρίας επιλέξαμε να εξετάσουμε το θέμα αυτό και από τη σκοπιά της οικονομικής κρίσης. Όχι γιατί πιστεύουμε, όχι γιατί θεωρούμε ότι η κρίση οδηγεί ευθύγραμμα στη βία κατά των γυναικών. Είμαστε όμως πεπισμένοι ότι περισσότερες γυναίκες θα αναζητήσουν διέξοδο από μια κακοποιητική σχέση αν έχουν την ψυχολογική στήριξη των ειδικών αλλά και την οικονομική ανεξαρτησία. Όπως και στην υπόλοιπη Ευρώπη, έτσι και στη χώρα μου, έτσι και στην Ελλάδα, το πρόβλημα της βίας κατά των γυναικών δεν είχε μέχρι πρόσφατα αναδειχθεί επαρκώς. Η κοινωνία μας, η ελληνική κοινωνία εννοώ, στη προσπάθεια να ελέγξει αυτό το κλιμακούμενο φαινόμενο έκανε βήματα προς την σωστή κατεύθυνση. Η κάθε μορφή βίας, ψυχολογική και σωματική, κατά των γυναικών, όπως σας ανέφερε πριν λίγο η κυρία Ρεπούση, μέλος του Ελληνικού Κοινοβουλίου, απαγορεύτηκε και τυπικά πριν λίγα χρόνια με τον νόμο 3500. Αυτό έγινε το 2006. Ο νόμος αυτός ρυθμίζει τις σχέσεις όλων των μελών της οικογένειας, αλλά και τις σχέσεις μεταξύ μόνιμων συντρόφων, εκτός γάμου, περιλαμβάνοντας και τα παιδιά τους. Αυστηροποιείται το πλαίσιο των κυρώσεων που αφορούν σε πράξεις εντός του οικογενειακού πλαισίου, όπως η σωματική κακοποίηση και η άσκηση ή η απειλή άσκησης βίας. Η ενδοοικογενειακή βία πλέον, σύμφωνα με τον νόμο, θεωρείται τεκμήριο ισχυρού κλονισμού του γάμου προϋπόθεση για την έκδοση διαζυγίου. Γίνεται ειδική μνήα για άσκηση βία σε βάρος εγγύου, προβλέποντας ακόμα πιο αυστηρές ποινές. Για πρώτη φορά αναγνωρίζεται ως αδίκημα η σεξουαλική κακοποίηση και ο βιασμός της γυναίκας εντός του οικογενειακού θεσμού. Ε, επειδή έχω μόνο 10 λεπτά, για τον νόμο θα ήθελα να συμπληρώσω ότι προβλέπεται στο, στο νόμο αυτό προβλέπεται και η διαδικασία παροχής αρρωγής στα θύματα ενδοοικογενειακής βίας και αυτό φαίνεται η βούληση από το νόμο αυτό του νομοθέτη, η βούληση της πολιτείας να προστατέψει τα θύματα, είτε αυτά είναι οι γυναίκες είτε τα παιδιά τους. Μάλιστα, για να εφαρμοστεί στην πράξη αυτή η διαδικασία, επειδή αντιμετωπίσαμε αρκετά κενά στην εφαρμογή, όχι τόσο στο νόμο, ε, ήταν αναγκαίο καταρχά να εφοδιαστεί η ελληνική αστυνομία με την κατάλληλη, με την κατάλληλη πληροφορία ω προ το είδο τη βοήθεια που χρειάζεται το θύμα τη ενδοοικογενειακή βία, που συνήθω είναι γυναίκα. Έτσι. Έτσι ξεκινήσαμε τον Αύγουστο που μας πέρασε, ενώ η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φίλων και η Ελληνική Αστυνομία, μια στενή συνεργασία, στη βάση συγκεκριμένου κειμένου οδηγίας για το χειρισμό υποθέσεων ενδοοικογενειακής βία ένα κείμενο που έφυγε με το σύστημα Police Online σε όλες τις αστυνομικές αρχές της επικράτειας. Θα σταματήσω εδώ για τον νόμο και θα ήθελα να αναφέρω το εξής. Στην Ελλάδα, προκειμένου να αντιμετωπιστεί σφαιρικά το πολύπλοκο αυτό πρόβλημα και φαινόμενο, οι προσπάθειες ξεκίνησαν ήδη από το 1980, από τη δεκαετία του 1980. Το πρώτο, το πρώτο συμβουλευτικό κέντρο για γυναίκες θύματα έμφυλης βίας δημιουργήθηκε το 1988. Λίγο αργότερα, το 1993, σε συνεργασία με τον πρώτο Δήμο της χώρας, με την πρωτεύουσα της χώρας, με το Δήμο Αθηναίων, λειτουργήσε ο πρώτος ξενώνας για τις γυναίκες θύματα βίας. Σήμερα. Σήμερα στη Γενική Γραμματεία στη Γενική Γραμματεία των Φίλων, υλοποιούμε ένα συγκροτημένο εθνικό πρόγραμμα για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών. Το πρόγραμμα αυτό χρηματοδοτείται, συγχρηματοδοτείται από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους. Περιλαμβάνει καταρχάς την ανάπτυξη υποδομών, οι οποίες έχουν σχεδόν στο σύνολό τους ολοκληρωθεί. Έτσι μιλάμε για 14 συμβουλευτικά κέντρα στις έδρες των περιφερειών της χώρας, προκειμένου να παρέχουν ψυχοκοινωνική και νομική στήριξη στις γυναίκες θύματα βίας, 25 συμβουλευτικά κέντρα, τα οποία είναι υπό την ευθύνη της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ε, στην ολοκλήρωση του προγράμματος θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα έχουμε, 21 ξενώνες, θα έχουμε δημιουργήσει 21 ξενώνες φιλοξενίας. Αυτή τη στιγμή ήδη έχουν ε, παραδοθεί οι 13, αναμένεται μέσα στους επόμενους μήνες να παραδοθούν οι άλλοι 9 και ήδη ε, λειτουργούν δύο ξενώνες οι οποίοι έχουν αναβαθμιστεί του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Υπουργείου Υγείας. Στο τέλος του προγράμματος ελπίζουμε οι ξενώνες να είναι 21, οι οποίοι είναι 21 ξενώνες διάσπαρτοι σε όλη τη χώρα. Όπως καταλαβαίνετε, οι υπηρεσίες των δομών αυτών παρέχονται δωρεάν και καλύπτονται από το απόλυτο απόρριτο της συμβουλευτικής. Οι εργαζόμενοι τόσο στα συμβουλευτικά κέντρα όσο και στους ε, ξενώνες φιλοξενίες λαμβάνουν ειδική επιμόρφωση. Στα συμβουλευτικά κέντρα υπάρχει και ειδικό πρωτόκολλο συνεργασία με του κατατόπου δικηγορικού συλλόγου, προκειμένου να παρέχεται και νομική στήριξη στι γυναίκε θύματα βία. Ε, δεν θα αναφερθώ ποιε γυναίκε απευθύνονται στα συμβουλευτικά κέντρα, γιατί φαντάζομαι όλε αντιλαμβάνεστε ποιε. Και απλά θα συμπληρώσω στο σημείο αυτό ότι τα δύο πρώτα χρόνια που άρχισαν να λειτουργούν σταδιακά όμως, και θέλω να το τονίσω αυτό, τα συμβουλευτικά κέντρα, υποδέχτηκαν περισσότερο από 2.650 γυναίκες. Αριθμός καθόλου μικρός, αν σκεφτούμε ότι μιλάμε για μια χώρα των 10 εκατομμυρίων κατοίκων και ότι μιλάμε για τις γυναίκες εκείνες που τόλμησαν να καταγγείλουν την εις βία για τις γυναίκες εκείνες που τόλμησαν να ζητήσουν βοήθεια. Εδώ πέρα βέβαια θα πρέπει να μας προβληματίσει όπως και για την έρευνα ο σκοτεινός αριθμός των γυναικών αυτών, οι οποίες δεν τολμούν να μοιραστούν το πρόβλημά τους. Έχει πραγματοποιηθεί συνεργασία ε, και δια, ε, δικτύωση με φορείς και υπηρεσίες όπως η αστυνομία, η εισαγγελία, τα νοσοκομεία, οι κοινωνικές υπηρεσίες. Ε, οι δομές αυτές συμπληρώνονται από την τηλεφωνική γραμμή 24 ώρες λειτουργίας ε, όπου δίνεται άμεση κοινωνική και ψυχολογική αλλά και νομική βοήθεια. Ε, τρέχω γρήγορα γιατί ο πρόεδρος μου κάνει σήμα να τελειώνω. Ε, θεωρώ κλείνοντας ότι πρωτοβουλίες σε επίπεδο κρατών μελών θα πρέπει να προχωρούν με βάση ένα κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο. Καλές οι ενέργειες και πρωτοβουλίες που παίρνουμε ως χώρα μέλος, ως ξεχωριστή χώρα μέλος αλλά νομίζουμε ότι και σε αυτό, νομίζω ότι και σε αυτό το θέμα θα πρέπει να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και να το δούμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο γιατί είναι ντροπή για την Ευρωπαϊκή Ένωση του 21ου αιώνα να, έχει ακόμα, να μην έχει λύσει αυτό το πρόβλημα. Τέλος, και τελειώνω πράγματι με αυτό, στη διάρκεια της ελληνικής προεδρίας επιδιώκουμε, και νομίζω ότι σε μεγάλο ε, ε, βαθμό το έχουμε καταφέρει, την ένταξη του θέματος αυτού στο αρμόδιο Συμβούλιο Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων και την αϊοθέτηση αντίστοιχων συμπερασμάτων στη φάση της προετοιμασίας του σχεδίου συμπερασμάτων, πολύτιμο εργαλείο, όπως καταλαβαίνετε, αποτέλεσαν και αποτελούν ε, τα στοιχεία που είχαμε σήμερα από την έρευνα του ΦΡΑ. Θα κλείσω με κάτι το οποίο αναφέρω κάθε φορά που επισκέπτομαι κάποιο συμβουλευτικό κέντρο ξενών φιλοξενίας και στην πατρίδα μου. Μίλησα πριν για ευρείες κοινωνικέ συμμαχίε, για συμμαχίες προκειμένου να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα αυτό. Νομίζω η σημαντικότερη όμως συμμαχία είναι μία. Η συμμαχία με τους άντρες. Γιατί κυρίε και κύριοι, αυτό το δρόμο δεν μπορούμε να τον διανύσουμε μόνες μας. Όπως και κανένα άλλο δρόμο δεν μπορούμε να διανύσουμε μόνες μας. Διότι δεν θα υπάρξει ισότητα χωρίς τον άντρα και μόνο με τη γυναίκα. Η ισότητα για να επιτευχθεί χρειάζονται και τα δύο φύλλα, και ο άντρα και η γυναίκα. Και θεωρώ ότι στην πορεία μας αυτή πρέπει να είμαστε κοντά με το συνοδοιπόρο, συνοδοιπόρο της ζωής μας τον άντρα. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. 14 λεπτά μίλησα, λέει κυρία Κούλη. Σας ευχαριστώ πολύ για την ε, παρέμβασή σας. Εκτιμούμε πάρα πολύ το γεγονός ότι βρήκατε το χρόνο να έρθετε και να μας παρουσιάσετε και τις θέσεις Ελληνικής Προεδρίας και ως Προεδρία πραγματικά μπορείτε να επηρεάσετε τις πολιτικές σε επίπεδο Συμβουλίου που είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν για μας να ακούσουμε τις θέσεις σας. Σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Λοιπόν, στρέφομαι στην τελευταία ομιλήτριά μας ε, που είναι η κυρία Αντωνία Παρβάνοβο. Συνεργαζόμαστε πολύ στην Επιτροπή Γυναικών, είναι και συντονίστρια ε, των φιλελευθέρων. Ε, συναντιόμαστε συχνά και συζητούμε και εκτιμώ πάρα πολύ ε, ε, το έργο της. Είναι πάρα πολύ ε, ένθερμη υπερασπίστρια των θεμάτων. Ήταν και η συγκήτρια της έκθεσης που εγκρίναμε πριν από μία εβδομάδα. Και χαίρομαι πάρα πολύ που εγκρίθηκε η έκθεση αυτή και ε, τώρα έχουμε και πιο ισχυρά εργαλεία για να αγωνιστούμε, γιατί πραγματικά θέλουμε να έχουμε νομοθετική πρόταση από πλευρά Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Παρακαλώ, ε, η Αντώνια θα μας εξηγήσει περισσότερο. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Συζητήσαμε ολόκληρη την ημέρα για τη βία κατά των γυναικών. Πολλέ από εμά το συζητούμε αυτό από χρόνια. Και είμαστε πολύ αποφασισμένες να βρούμε λύσεις ή τουλάχιστον να κάνουμε ένα βήμα πρόοδου. Και δεν είναι μόνο η έκθεση αυτή το ζήτημα. Δεν είναι η δέσμευση του Ευρωκοινοβουλίου της Επιτροπής ΦΑΜ για να αντιμετωπιστεί το θέμα της εξάλληψης της βίας κατά των γυναικών. Έχουμε και άλλα βήματα και άλλες κινήσεις με την προσπάθεια όλων των ε, ε, ευρωβουλευτών, όλων των εκπροσώπων των εθνικών κυβερνήσεων. Θέλουμε αλλαγή στο καθένα κράτος μέλος. Εδώ και τόσο καιρό συνεργαζόμαστε με το λόμπι, το Ευρωπαϊκό Λόμπι των Γυναικών, με ακτιβίστριες και ακτιβιστές μπορούμε επιτέλους να έχουμε κάποια επίδραση και πολιτική βαρύτητα. Απλώς πρέπει να είμαστε πιο αποφασιστικές. Όταν ξεκίνησα ήμουν απλώς παρατηρήτρια, όταν πρότεινα να προβλεφθεί η, ο συντονιστής για το θέμα της εμπορίας. Δεν με πίστευαν καν οι συναδελφοί μου. Κι όμως οι επικεφαλείς της ομάδας μου μου είπαν Ξεκίνατο. μίλα στους υπόλοιπους βουλευτές. Και έτσι προτάθηκε και υποβλήθηκαν τροπολογίες. Μετά για κανένα εξάμεινο ήμουν μέλος του Ευρωκοινοβουλίου Ιανουάριο του 2007 έως Ιούνιο του 2007 και δεν είχαμε καν εκλογές ακόμα στην ε, Βουλγαρία. Αλλά υπέβαλα την πρόταση για τη θέσπιση της θέσης αυτής του συντονιστή για την καταπολέμηση της ε, εμπορίας ανθρώπων. Ε, είναι τουλάχιστον ένα αξίωμα και θα υπάρχει μια πολιτική και μια χρηματοδότηση για να μπορέσουν τα κράτη-μέλη να συντονίσουν τη δράση του τομέα αυτό και να ανταλλάξουν πρακτικές. Και μόνο έτσι θα μπορέσουν να συλλέξουν δεδομένα. Και δεν μου ήρθε στα ξαφνικά, σαν κεραυνό σε ουρανό ενεθρία. Όχι, το συζητήσαμε με μη κυβερνητικέ οργανώσει και με την Επιτροπή μας Και Επιτέλους τώρα η Επιτροπή μας πίεσε τις Επιτροπές Δικαιωμάτων των Πολιτών και νομικών υποθέσεων στη δική τους δουλειά, στην οδηγία για τα θύματα και τα δικαιώματά τους και την ε, εντολή προστασίας να ε, λάβουν μέρημνα των όσων μας απασχολούν. Και με τη στήριξη της Επιτροπής των, ε, Δικαιωμάτων των Γυναικών και του Ευρωπαϊκού Λόμπι για τις Γυναίκες καταφέραμε να έχουμε έναν ορισμό για τη βία κατά των γυναικών σε αυτήν την νομοθετική πράξη. Είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο. Έχουμε μια ποινική, ε, στον ποινικό κώδικα των κρατών μελών έναν ορισμό για τη βία κατά των γυναικών. Εγώ αρχικά είχα μιλήσει για την έμφυλη βία, για τη σεξουαλική βία και τη βία τις ε, στενές σχέσεις. Είναι τρεις διαφορετικές μορφές, τρεις διαφορετικές συνδυασμοί, κατά των γυναικών και τρεις, αλλά υπό διαφορετικές περιστάσεις. Εγώ λοιπόν, λόγω της πρότασης της Επιτροπής ΦΕΜ και με τη δική σας την έμπνευση, τη δική σας τη στήριξη, κατάφερα να ε, ε, πετύχουμε ξεχωριστές αποτιμήσεις των αναγκών των θυμάτων, ώστε να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις γυναίκες θύματα εγκληματικών ενεργειών. Το ίδιο και για, τα, για την εντολή προστασίας. Είναι κάτι που γίνεται. Δεν αρκεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας λέει ότι δεν, αρκεί, δεν υπάρχει νομική βάση για το ένα ή για το άλλο για, νομοθετική, για έκθεση πρωτοβουλία. Πρέπει να ε, υπάρξει ε, ανταπόκριση στις οκτώ εκκλήσεις μας. Βάσει του άρθρου 84 της συνθήκης ζητούμε εκπαίδευση και κατάρτιση των ε, ε υπαλλήλων που συμμετέχουν, των αστυνομικών που ασχολούνται με αυτά. Μην κάνετε καμία προσπάθεια να το ε, παρακάμψετε αυτό, παρακαλώ. Υπάρχει νομική βάση για την ανταλλαγή πρακτικών. Επίσης, το, βάση του άρθρου 83.1 μπορεί να προσθεθεί η έμφυλη βία στα ε, εγκλήματα που ονομάζονται Eurocrimes με διασυνοριακές προεκτάσεις. Και μαζί με το οργανωμένο έγκλημα, την τρομοκρατία, το κυβερνοέγκλημα είναι ένα σοβαρότατο πρόβλημα στην Ευρώπη να μην αμφιβάλλετε, διότι η επικουρικότητα δεν σημαίνει ανεξαρτησία για κάθε κατός μέλος, δεν σημαίνει να κάνουν ό,τι τους κατέβει ο καθένας και να το λύσουν όπως τους αρέσει. Όχι, επικουρικότητα σημαίνει ότι αν ένα θέμα δεν μπορεί να επιληθεί σε περιφερειακό επίπεδο, πάει στο εθνικό. Και αν δεν μπορεί να επιληθεί στο εθνικό, τότε πάει στο ευρωπαϊκό, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπωσδήποτε η έμφυλη βία είναι ένα θέμα που δεν έχει επιληθεί στο εθνικό επίπεδο. Ιδάλω δεν θα είχαμε την έκθεση ΦΡΑ όπως την λάβαμε με αυτά τα τόσο ανησυχητικά, αυτά τα τόσο απέσια δεδομένα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν θα πρέπει να προβλέψει μια πρόταση για να στηρίξει και να παρατρύνει τη δράση των κατομελών ώστε να κάνουν κάτι για την βία κατά των γυναικών. Μπορεί να υπάρξει μια πράξη για την πρόληψη. Επίσης, ε, έκλεισε για τα στατιστικά δεδομένα. Μπλοκαρίστηκε στο κοινοβούλιο η έκθεση για τα στατιστικά δεδομένα. Δεν σημαίνει όμως ότι δεν μπορεί να πάει πίσω, να αναπευθεί και να ξανασυνταχθεί, να ξαναεποβληθεί, συμπεριλαμβάνοντας την ε, έμφυλη βία. Παρακαλώ λοιπόν, υπάρχουν κάτι μέλη που θεωρούν ότι δεν θα έπρεπε να συλλέγονται στοιχεία για την αφιληβία ή για τα έμφυλα δεδομένα γενικότερα α, λένε ότι είναι αντισυγματικό. Όμω, όταν τρώνε ξύλο γυναίκε, θα έπρεπε να συγκεντρώνονται στοιχεία, ό,τι και αν λέει ένα σύνταγμα. Διότι πρόκειται για αδίκημα, πρόκειται για έγκλημα. Δεν, δεν νομίζω ότι μπορούμε να ονομάζουμε έγκλημα τον ξυλοδαρμό ανδρών από άντρε, ενώ όταν οι γυναίκε ε, μπορεί να είναι θύματα ξυλοδαρμού, να είναι ένα ζήτημα που θα μείνει στα... στο σπίτι. Then we call on... Επίσης, θέλουμε ένα πρόγραμμα δράσης τον ακροτηριασμό των γυναικείων ε, γενετικών οργάνων. Και εκεί χρειάζεται ε, περισσότερα, στοιχεία. Πάνω από 7.000, πάνω από, πάνω από 500.000 γυναίκες έχουν πέσει θύματα αυτού του φαινομένου και στην επικράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης πώς γίνεται τόσες γυναίκες να έχουν πέσει θύματα, πώς μπορούμε να κάνουμε κήρυγμα σε άλλους, σε τρίτες χώρες και να λέμε ότι εμείς είμαστε σύγχρονοι, ότι έχουμε τις καλύτερες πρακτικές, ότι είμαστε παράγων, πρωταγωνιστής στα ανθρώπινα δικαιώματα. Πώ μπορούμε κάθε χρόνο να δημοσιεύουμε μια έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα, εάν επιτρέπουμε στην ίδια την επικράτη τη Ευρωπαϊκή Ένωση ο ακροτηριασμό αυτό να συνεχίζεται. Είναι απίστευτο. Δεν θα μα πιστέψουν ποτέ, δεν μπορούμε να του πείσουμε Έχουμε το βραβείο Ζαχάροφ. Πώ μπορούμε κάθε χρόνο να έχουμε την απονομή ενό τέτοιου βραβείου, ενώ δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε μια τόσο σοβαρή, μια τόσο εγκληματική ενέργεια στην επικράτεια τη Ένωση. Για τη σύμβαση επίση τη Κωνσταντινούπολη. Πρέπει να κυρωθεί. Θα πρέπει επιτέλου η Ένωση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να έχουν μια σαφή δήλωση. Πότε θα γίνει ένα νομικό εργαλείο. Θα γίνει ή όχι. Τα στηρίζουμε ή όχι. Δεν αρκεί να πηγαίνουμε στον ΟΗΕ και να πηγαίνει το κάθε κάτω μέλο ξεχωριστά ή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή όλοι μας και να λέμε ότι μας ανησυχεί πάρα πολύ η βία κατά των γυναικών αλλά ταυτόχρονα με την κυρώνουμε την ε, σύμβαση. Δεν είναι δίκαιο. Δεν είναι λογικό. Δεν μπορούμε να δίνουμε εμεί ε, το παράδειγμα στους άλλους και να πετάμε στην Τουρκία τις βέλτιστες πρακτικές μας ε, δίνοντας κηρύγματα για το πώς να γίνουν πιο Ευρωπαίοι και χώρα της ε, ένταξης, εάν δεν μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημα στη δική μας την επικράτεια και δεν μπορούμε να κυρώσουμε τη σύμβαση της Κωνσταντινούπολης. Επίσης, θέλουμε ένα ευρωπαϊκό παρατηρητήριο. Παρατηρητήριο για τη βία κατά των γυναικών. Είναι πολύ σημαντικό. Έχουμε το συντονιστή για την αντιμετώπιση της διακίνησης, αλλά πρέπει να υπάρξει και ε, παρατηρητήριο για τη βία κατά των γυναικών. Και επίσης ευρωπαϊκό έτος ειδικά αφιερωμένο στην καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών. Αυτές είναι οι πρωτοβουλίες του, λόμπι, του Ευρωπαϊκού Λόμπι για τις γυναίκες. Δεν είναι πρόβλημα, είναι ένα θέμα που πρέπει να το κάνουμε. Ναι, είναι ένα πρόβλημα που σοκάρει ή είναι κάτι που ξαφνιάζει. Πρέπει να γίνει. Η Επιτροπή των Δικαιωμάτων των Γυναικών και της Ισότητας των Φύλων έκανε έκκληση ώστε να προβλεφθεί ένα ευρωπαϊκό βραβείο για όσους βουλευτές πραγματικά ασχολούνται με τα δικαιώματα των γυναικών. Πέρσι έγινε. Το προτείναμε και έγινε. Και είμαι ιδιαίτερα υπερήφανη που η Επιτροπή ΦΑΜ ε, επέμεινε. Και το βραβείο αυτό απονεμήθη στον συνάδελφο συντονιστή του ΕΛΚ, ε, του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην Επιτροπή των Γυναικών. Έτσι πρέπει να προχωράμε βήμα-βήμα και θα υπάρξει σοβαρός αντίκτυπος, όχι μόνο στην νομοθεσία, αλλά θα υπάρξουν αποτελέσματα και στις εξελίξεις της κοινωνίας μας. Δεν πρέπει απλώς να ασχολούμαστε με τα οικονομικά ζητήματα. Και αν μιλούμε από οικονομική σκοπιά όσο κοινικό και αν ακούγεται, προκαλεί βία κατά των γυναικών. 220 δις ευρώ απώλεια ετησίως για την οικονομία της Ένωσης. Υπάρχει λοιπόν και οικονομικό υπόβαθρο αν θέλουμε να είμαστε κοινικοί. Όμως νομίζω είναι πιο σημαντικό να μιλάμε για ανθρώπινα δικαιώματα παρά για τους αριθμούς δις ευρώ που μπορεί να χαθούν. Σα ευχαριστώ λοιπόν πολύ. Πραγματικά στηριζόμαστε στι δικέ σα προσπάθειε σε εθνικό επίπεδο και επίπεδο ένωση. Σα ευχαριστώ. Καλή τύχη σε όλε. Σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε και όπω είπα η εκθέσή σας είναι εξαιρετική και την υποστήριξα απολύτω. Πριν κλείσουμε θα ήθελα να πω ότι όλοι εδώ κατανοούμε και αναγνωρίζουμε ότι είναι έγκλημα η βία κατά των γυναικών και κατά των θεμελιδών δικαιωμάτων των γυναικών. Η μελέτη του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων ε, της Ένωσης μας δίνει πολύ συγκεκριμένα επιχειρήματα και πάρα πολύ καλά όπλα για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε, γιατί έχουμε και τώρα τα αριθμητικά στοιχεία να τα τεκμηριώνουμε αυτά που λέμε. Η Επιτροπή ε, Γυναικών και Ισότητας θα εργαστεί πάρα πολύ σκληρά σε αυτά τα θέματα, όπως κάναμε την περασμένη πενταετία, είτε δια της νομοθετικής οδού, ζητώντας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δράσει, είτε μέσω της Σύμβασης της ε, Κωνσταντινούπολης, είτε και ε, με τα δύο. Και σας υπόσχομαι ότι η Επιτροπή μας Ανεξαρτήτως του αποτελέσματος των ευρωεκλογών θα εξακολουθήσει να αγωνίζεται για αυτά τα θέματα και να παλεύει και γενικότερα για την ισότητα των φύλων. Να πω κάτι τελευταίο, ότι ακόμα και είναι πάρα πολύ σημαντικό να αγωνίζεσαι και να καταπολεμάς τη βία κατά των γυναικών, θα πρέπει να θυμόμαστε ότι ο λόγος που υπάρχει η βία είναι η ανισότητα του φίλου στην κοινωνία. Γιατί διαρθρώνεται η κοινωνία με βάση το φύλλο, έχουν οι άνδρες πλέον και οι γυναίκες υφίστανται διακρίσεις σε σχέση με τους άνδρες. Και η βία κατά των γυναικών είναι ακριβώς η χειρότερη επίπτωση αυτού του πατριαρχικού συστήματος της κοινωνίας που ζούμε αυτό χρειάζεται καταπολέμηση αλλά και άλλα πολλά ζητήματα που συνδέονται με αυτό και να είστε βέβαιοι ότι η Επιτροπή Γυναικών θα εξακολουθήσει να παλεύει πολύ σκληρά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε και ε, για τη συμμετοχή σας ε, και όλους τους ομιλητές και ομιλήτριες. Μας δώσατε πολύτιμα στοιχεία και πληροφορίες για πάρα πολλά θέματα και ποικίλα. Ευχαριστώ τα μέλη του τελευταίου πάνελ και ιδιαίτερα την κυρία ε, Κόλια. Ευχαριστώ και τους διερμηνείς. Όπως πάντα, εξαιρετική δουλειά σας. Προσπαθείτε να μας φέρετε σε επαφή και να ε, μας κάνετε να καταλάβουμε ένα τον άλλον και θα σας θαυμάζω γι' αυτό. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω και τη γραμματεία και το προσωπικό που εργάστηκε για την εκδήλωση αυτή. Μπορείτε να φανταστείτε ότι είναι πολλή δουλειά ε, όλη αυτή η διοργάνωση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ένα τελευταίο, όπως είπα στην αρχή, εδώ ε, αμέσως έξω από την αίθουσα θα ακολουθήσει η δεξίωση. Παρακαλώ παραμείνετε για να μπορέσουμε να ανταλλάξουμε περισσότερες απόψεις και κατηδίαν. Ευχαριστώ πολύ.